Dear colleagues, uh, it's a pleasure to welcome you. Αγαπητοί συνάδελφοι, σας καλωσορίζω στη σημερινή ακρόαση για το πακέτο για τις θεωρήσεις που θα αρχίσει μετά την συνεδρίαση της ΛΥΒΕ. Ε, καλωσορίζω τους εμπειρογνώμενους που ήρθαν για να συμβάλλουν στη συζήτησή μας. Ε, το πρώτο τμήμα, νέος κώδικας θεωρήσεων. Θα δώσω το λόγο πρώτα απ' όλα στην κυρία Φαγιόν, που είναι η συγκήτριά μας. Και μετά έκαστος 10 λεπτά για τους εμπειρογνώμους κατόπιν συζήτηση. Έχουμε πολύ μεγάλο αριθμό μιλητών. Παρακαλώ, λοιπόν, να μην υπερβαίνετε το χρόνο αγόρευσης. Θα αναγκαστώ να σας διακόψω, εάν τον υπερβείτε. Η κυρία Φαγιόν. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Χαίρομαι που σήμερα έχω την ευκαιρία να συζητήσω μαζί σας ένα από τους σημαντικότερους φακέλους που εξετάζει αυτή τη στιγμή το Κοινοβούλιο και θα ήθελα τώρα να κάνω τις αγωγικέ μου παρατηρήσεις και στη συνέχεια θα είμαι στη διάθεσή σας για κάποιε καταληκτικέ ε, παρατηρήσει. Η πρόταση τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την αναθεώρηση του κώδικα θεωρήσεων γίνεται σε μια χρονική περίοδο που πρέπει να αντεπεξέλθουμε σε μια σειρά από προκλήσεις. Καταρχάς, ένας από τους στόχους θα πρέπει να είναι να τονώσουμε ε, την οικονομία μας, κυρίως στον τομέα του τουρισμού και να δημιουργήσουμε νέες θέσεις εργασίας, ε, διότι μετά την κρίση αυτό χρειαζόμαστε απομονισμένα στην Ευρώπη. Κατόπιν, ε, πρέπει να ξεχνάμε ότι αυξάνεται διαρκώ η μεταναστευτική πίεση, η ανθρώπινη τραγωδία στη Μεσόγειο και κυρίως για λόγους ασφαλείας, εξτρεμισμός, λαϊκισμός ρατσισμός και η ξενοφοβία είναι δυνάμει που μας αναγκάζουν ε, να ε, συσπηρωθούμε γύρω από τις βασικές μας αξίες όπως η ελευθερία τη κυκλοφορία των ατόμων διότι τίθεται να αμφιβόλω η ίδια λειτουργία της ζώνης Σέγγεν. Θα πρέπει λοιπόν να συζητήσουμε με τις προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, να ακούσουμε τους εμπειρογνώμονες και του εμπλεκόμενου φορείς για να διαμορφώσουμε τη θέση μας. Θα ήθελα να σας καλωσορίσω. Σας ευχαριστώ που ήρθατε. Παρότι πριν από λίγες εβδομάδες με διόρισαν εισηγήτρια, ε, θα ήθελα να ευχαριστήσω παρόλα αυτά τους σκιώδες τη γραμματεία, διότι σε αυτές τις λίγες εβδομάδες ήδη έχω δει έμπρακτη υποστήριξη. Θα ήθελα να καλωσορίσω την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ο στόχος της είναι να δυναμώσει την ευρωπαϊκή διάσταση, να διευκολύνει τις μετακινήσεις ε, για όσους μόνιμα μετακινούνται, να διευκολυνθεί η διαδικασία για την έκδοση θεωρήσεων και να ε, βελτιωθεί η λειτουργία του συστήματος ε, Schengen, διότι αυτό είναι απαραίτητο για τους πολίτες μας. Ε, θα πρέπει να εξυπηρετήσουμε τον ίδιο στόχο, να γίνει ευρωπαϊκή, ε, σύγχρονη και ευφυής ε, η πολιτική. Οι νέες τεχνολογικές αλλαγές θα μας επιτρέψουν να είναι λίγο επαφής η διαδικασία και να διευκολυνθεί θα ήθελα λοιπόν να ασχοληθούμε με το θέμα των προξενικών διαδικασιών για τους ετούντες. Ε, θα πρέπει να ενισχύσουμε την ε, διευκόλυνση της διαδικασίας κυρίως για όσους έχουν ταξινομηθεί ως ε, συνήθις ταξιδιώτες που μετακινούνται συχνά δηλαδή στη ζώνη Σέγγεν για κάποιες κατηγορίες, παραδείγματος χάρη για τους ναυτικούς, θα πρέπει να έχουμε απλουστευμένες διαδικασίες. Καλωσορίζουμε αυτή τη ριζοσπαθία συμβαστική πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, για, ε, που απαριθμεί όλα τα στοιχεία που θα πρέπει να εξετάσουμε. Παρόλα αυτά κάνουμε και εμείς επιπρόσθετες προτάσεις ε, για την περαιτέρω απλούστευση της διαδικασίας. Ε, ε, ζούμε σε ένα παγκοσμιοποιημένο και ψηφιοποιημένο κόσμο, άρα η ε, επιγραμμική αίτηση πρέπει να είναι κάτι που θα ενθαρρύνουμε και θα πρέπει επίση να καταστεί δυνατό εννέα μήνε πριν από την προβλεπόμενη επίσκεψη να μπορεί να δρομολογηθεί αυτή η διαδικασία. Ή ακόμη και νωρίτερα, αν μπορεί να αιτιολογηθεί αυτό, κυρίω αυτοί που μετακινούνται τακτικά μπορούν έτσι να εξοικονομήσουν μεγάλο κόστος από τα αεροπορικά εισιτήρια παραδείγματο χάρη. Τα, οι διαδικασίες στα αρμόδια προξενία είναι ιδιαίτερα ε, μακροσκελής και υπάρχει ένα υπερβολικό διοικητικό άκθος που βαραίνει τον ετούντα. Θα πρέπει λοιπόν να έχει τη δυνατότητα στο προξενείο να καταθέτει την αίτηση του ε, όποιος επιθυμεί να ε, μετακινηθεί και κυρίως στο μέρος που είναι εγκύτρο στον τόπο διαμονής ακόμη και αν δεν είναι η χώρα στην οποία θα ταξιδέψει, που εκπροσωπείται σε αυτό το προξενείο. Στη συνέχεια ε, θα πρέπει να είναι δυνατή η προσφυγή ενώπιον ε, τη δικαστική αρχή ε, για τι εφέσει, διότι ορισμένα κράτη-μέλη πρόκειται μόνο για διοικητικέ διαδικασίε. Το συμφέρον του ταξιδιώτη θα πρέπει να το έχουμε κατά νου όταν πρόκειται για θεωρήσει που έχουν ανακληθεί χωρί τη δέουσα διολόγηση λόγω των ζημιών και των απολειών για τον ταξιδιώτη. Παραδείγματο χάρη, ακύρωση του αεροπορικού εισιτηρίου ή τη ε, διαμονή στο ξενοδοχείο. Δεύτερον, για, ε, για τα προξενία και τις θεωρήσεις, συνεργασία ανάμεσα στα κράτη-μέλη και τα κοινά κέντρα υποβολής αιτήσεων ε, πρέπει να διέπονται από τον κανονισμό. Είναι ιδιαίτερα υποφελή αυτή τη λύση για τον ταξιδιώτη. Ε, το διοικητικό άρθρο όμω εξακολουθεί να βαρύνει τα κράτη-μέλη. Με τι μελλοντικέ εξελίξει θα μπορούσαμε να έχουμε ελκυστικέ εναλλακτικέ λύσει ε, και για τα κράτη-μέλη. Επίση αυτό είναι ένα άλλο βήμα προ ε, τον απότερο στόχο, δηλαδή να καταστεί πραγματικά ευρωπαϊκή πολιτική για τι θεωρήσει. Ακόμη και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην αξιολόγηση αντικτύπου αναφέρεται στα κέντρα θεωρήσεων, του, γιατί, οπότε ε, έχουμε όλοι κατά νου ε, ε, την μελλοντική δυνατότητα να έχουμε τέτοια ευρωπαϊκά κέντρα. Χρειάζονται οι πληροφορίες όπως η συνολική διάρκεια σε κάθε κράτος μέλος, ε, δηλαδή όχι πάνω από 90 ημέρες, οποιαδήποτε περίοδο 180 ημερών, αλλά θα πρέπει να είναι ενήμεροι και οι ταξιδιώτες για αυτόν τον κανόνα. Για τους εξωτερικούς παρόχους υπηρεσιών θα επιμείνω να χρησιμοποιηθεί αυτό ως ίστατη λύση και μόνο. Ε, Παρ' θα παραμείνει η διάταξη στον κανονισμό, παρότι καταλαβαίνω καταλαβαίνω το συλλογισμό και την επιχειρηματολογία γιατί σε ορισμένε περιπτώσει ε, ε, χρειάζεται φιναλλακτική όταν είναι προβληματική η κατάσταση προ την ασφάλεια σε τρίτε χώρε. Παρόλα αυτά έχουν εκφραστεί ε, ανησυχίε στο Κοινοβούλιο και θα πρέπει με κάποιο τρόπο να δώσουμε μια απάντηση. Τα κράτη-μέλη θα πρέπει επίση να διατηρήσουν τη δυνατότητα όλοι οι αιτούντε να μπορούν να υποβάλουν στι δημοκρατικέ αποστολέ ή στα προξενία απευθεία τη αιτή Όμω όμως ε, ε, θα πρέπει ταυτόχρονα να βελτιωθεί η διαδικασία η συνεργασία με εξωτερικούς παρόχου υπηρεσιών, διότι ε, χρειάζεται να εξασφαλιστεί και η ανταλλαγή πληροφοριών βάσει του συστήματο ΒΙΣΕ με του εξωτερικού παρόχου υπηρεσιών. Τέλος, αλεξίου σημαντικό, υπάρχει το θέμα των ανθρωπιστικών θεωρήσεων. Πέρα από κάποια επιχειρημάτα, αν δηλαδή ε, είναι πρόσφορη αυτή η νομική πράξη για τις ανθρωπιστικές θεωρήσεις. Μην ξεχνούμε ότι υπάρχει αυτή η διάταξη και στον κανονισμό για τον κώδικα Σέγγινα και στον ισχύοντα κανονισμό για τις θεωρήσεις. Ε, η φτάμενη διάταξη όμως θα πρέπει να ευθυγραμμιστεί με τον συνεργειακό κώδικα του Σέγγεν και σε ολόκληρο τον κανονισμό θα πρέπει να προσθέσουμε και τις διεθνείς υποχρεώσει που έχουμε καθώς και μια νέα αιτιολογική σκέψη για να υπάρχει αντιστοίχηση με το διατακτικό. Δεν νομίζω να μπορούμε να ε, δείξουμε μεγαλύτερη φιλοδοξία για αυτό το ανθρωπιστικό ζήτημα πάντως ε, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τι υφιστάμενες διατάξει του γεκτημένου του Σέγγεν ε, και μην ξεχνάμε ότι μόνο λίγε χώρε προσφεύγουν σε αυτή την εναλλακτική που ήδη υπάρχει δηλαδή για την έκδοση ανθρωπιστικών θεωρήσεων. Αυτά λοιπόν από μένα και ε, ε, θα είμαι στη διάθεσή σα. προσβλέπω στη μελλοντική μα συνεργασία και ελπίζω να παραμείνουμε φιλόδοξοι ω προς τον προγραμματισμό των μελλοντικών μας εργασιών εδώ στην Επιτροπή. Ευχαριστώ πολύ, πολύ ενδιαφέρουσα η παρουσίαση. Θέλουμε να ακούσουμε τι απόψει των διαφόρων ομιλητών. Ο κ. Τζάγκαρ. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ που καλέσατε έναν πρώην Γενικό Σύμβουλο. Γενικό πρόξενο. Λοιπόν, θέλω να παρουσιαστώ. Ήμουν ε, πρόξενο στο Αμπιτζάν, στο Τόκιο, στο Βανκούβερ και στο Αργέρι και τώρα έχω συνταξιδοτηθεί. Μπορώ να εκφραστώ με πλήρη ελευθερία λόγου και δράτω με τις ευκαιρίες. Καταρχάς, σε ένα προξενείο ε, είναι μόνιμη αντιπαράθεση με την πραγματικότητα η έκδοση των θεωρήσεων. Η πρώτη πραγματικότητα είναι η ετούντες ε, θεώρηση. Μεγάλος αριθμός αυτών που αυξάνεται. Κάθε τρίτος ε, αλλοδαπός που πρέπει να έχει θεώρηση είναι ενδεχόμενος ε, τον Βίζα. Έχουμε πολλά εκατομμύρια ανθρώπου σε κάθε προξενείο σαν υποψήφιου πελάτε. Δεν υπάρχουν πολλέ διοικητικέ δραστηριότητε όπου το ενδεχόμενο προσωπικό, το, η πελατεία είναι τόσο μεγάλη και όπου πρέπει να πάρουμε τόσε πολλέ ε, καθημερινέ αποφάσει. Στο Αλγέρι ήταν και είναι ακόμα 1.200 ετούντε ε, την ημέρα στο προξενείο της Γαλλίας. 1.200 αποφάσεις προσλήψη καθημερινά και αν οι δυνατότητες ήταν ακόμα μεγαλύτερες είμαι πεπισμένος ότι αυτό το στοιχείο θα ήταν ακόμα μεγαλύτερο αυτός ο αριθμός. Ε, υπάρχουν ποικιλόμορφες καταστάσεις. Έχουμε την απλή επόσταση κάποιος υποψήφιος που θέλει να κάνει οργανωμένο τουριστικό γύρο ή ένα επιχειρηματικό ταξίδι που το αναλαμβάνει με επιχείρηση. Αλλά πολύ συχνά πιο περίπλοκα τα πράγματα από αυτά, διαδοχικά ταξίδια για λόγους διαφορετικούς, αβεβαιότητες, όσον αφορά την ακριβή ημερομηνία του ταξιδίου και όσον αφορά τις συνθήκες στέγασης. Αυτά τα στοιχεία συνεπάγονται φυσικές, φυσικούς περιορισμούς. Πρώτα απ' όλα θα πρέπει να υποδεχτούμε τους ετούντες σε εξωπρεπείς συνθήκες και διαπιστώνουμε ότι υπάρχει αυξανόμενη απέτηση για ποιότητα όσον αφορά το χώρο υποδοχή. Πρέπει να εξεταστεί σημαντικό αριθμό φακέλων και εντό όλο και πιο σύντομων χρονικών διαστημάτων. Διότι ζούμε σε μια εποχή όπου η ταχύτητα έχει γίνει και αυτό μια απέτηση Πρέπει να εφαρμόσουμε κανονισμούς περίπλοκους, περιοριστικούς. Πρέπει προφανώς ε, να διαπράττουμε τα ελάχιστα δυνατά σφάλματα ούτε προς την ε, κατά μία έννοια δεν πρέπει να δίνουμε θεώρηση σε κάποιον που δεν πληρεί τις προϋποθέσεις ή που αντιπροσωπεύει ένα κίνδυνο, θα μας κατηγορούσαν γι' αυτό, ούτε από την άλλη κατεύθυνση θα κάνουμε λάθος. Δεν πρέπει να αρνούμε θα μία θεώρηση σε ένα άτομο που πληρεί τις συνθήκες και τους όρους και δεν παρουσιάζει κανένα ε, κίνδυνο. Θα μας κατηγορούσαν. Λοιπόν, οι αποφάσεις δεν είναι πάντα εύκολες να ληφθούν διότι τίποτα δεν μοιάζει περισσότερο με έναν ετούντα ε, ε, καλή την πίστη με έναν ετούντα κακή την πίστη. Τίποτα δεν μοιάζει με έναν πραγματικό τουρίστα με έναν ψεύδο τουρίστα. Τίποτα δεν μοιάζει περισσότερο με έναν πραγματικό καλλιτέχνη με έναν ψεύτικο. Πρέπει κάθε φορά να αξιολογείται ο κίνδυνος όμως ένας κίνδυνος δεν αποτελεί βεβαιότητα. Όταν αξιολογούμε έναν κίνδυνο ποτέ δεν είναι όλα λευκά και ε, μαύρα. Υπάρχει πάντα η γκρίζα ζώνη. Πρέπει πάντα να βρούμε μια θέση ανάμεσα στο ναι και στο όχι. Ε, το πρόβλημα είναι ότι η απόφαση είναι ε, διαδική. Είτε χορηγώ τη θεώρηση είτε αρνούμε. Χρειάζεται ριζοσπαστική απόφαση. Λοιπόν, πρέπει να κάνουμε μια σωστή αξιολόγηση. Και σας διαβεβαιώνω ότι σαν γενικός πρόξενος πρέπει να πω ότι η όλη προσπάθεια έχει κόστος. Λοιπόν, τα δικαιολογητικά που μας παρουσιάζεται από την άλλη πλευρά δεν αντιστοιχούν πάντα στις προδιαγραφές των ευρωπαϊκών κοινωνιών που αστυνομεύονται σωστά και βαστίζονται στα γραπτά και αξιόπιστα στοιχεία που επιτρέπουν την εμπιστεύεται κανείς το έγγραφο. Η καθημερινή ζωή στο προξενείο που βρίσκεται σε κάποιες χώρες είναι οι ψευδείς δηλώσεις όσον αφορά τα ψευδή, τραπεζικά έγγραφα ε, ή πραγματικά έγγραφα που χορηγούνται ενώ δεν δικαιούται ο, ο κάτοχος τα ψευδοαληθεί όπως λέμε και υπάρχουν και κάποιες συγκεκριμένες τιμές να αγοράζει κάποια ε, στοιχεία ταυτότητα σε κάποιες χώρες που δεν κατονομάζω και πρέπει να ομολογήσω ότι το προσωπικό των υπηρεσιών της θεώρησης δεν απαρτίζεται αποκλειστικά από επιφανείς νομικούς. Οι περισσότεροι είναι εκτελιστικοί αξιωματούχοι που κάνουν με τίμιο τρόπο τη δουλειά τους αλλά διαθέτουν πολύ σπάνια μια νομική εκπαίδευση υψηλού επίπεδου. Επιπλέον η άρνηση και η απόρριψη πολύ συχνά είναι κάτι που αμφισβητείται. Προσφυγές όλο και αυξάνονται. Πρέπει να εξετάζετε κάθε προσφυγή και να δίδετε μια απάντηση. Είσαστε σε καλή θέση να το γνωρίζετε ότι οι κυβερνήσεις αντιμετωπίζουν δημοσιονομικούς περιορισμούς και αυτό σημαίνει πιο συχνά ότι τα μέσα παραμένουν στάσιμα ή καμιά φορά μειώνονται ότι το προσωπικό έχει την τάση να μειώνεται από πλευράς αριθμού ε, προσωπικού και το κόστος της λειτουργίας θα πρέπει να μειωθεί. Το πρόβλημα ενός προξενείου είναι το εξής για να το συνοψίσω. Πώς να δεχούμε με αξιοπρέπεια έναν αριθμό ήδη αυξημένο και πάντα αυξανόμενο ετούντων και ταχαίως να λαμβάνονται αποφάσεις επί την ε, βάση των δικαιολογητικών, να είναι δίκαια η απόφαση, βάσει δικαιολογητικών που δεν είμαστε σίγουροι ότι είναι αυθεντικά, που υποβάλλονται από άτομα που είναι δύσκολο να εκτιμήσουμε αν είναι καλή την πίστη που κινούνται, εκτιμώντα έναν κίνδυνο που από τη φύση του είναι κάτι αβέβαιο με περιορισμένα μέσα που έχουν την τάση να μειώνονται. Λοιπόν, χρειαζόμαστε βοήθεια των ε, νομοθετών για να επιληθεί αυτή η δύσκολη εξίσωση. Αυτό που σας ζητούμε είναι να λάβουμε υπόψη τις επιτόπιες πραγματικότητες, δηλαδή να προσμετήσουμε τον αντίκτυπο των αποφάσεών σας επί των εργασιών ενός προξενείου. Δεν έχω το χρόνο να αναφερθώ σε όλες τις αλλαγές που προτάθηκαν από την Ευρωπαϊκή ε, Επιτροπή. Θα περιοριστώ σε κάποια σημεία γνωρίζοντας ότι είμαι πάντα στη διάθεσή σας για να σας εκθέσω αν χρειαστεί κάποια άλλα σημεία. Η εξωτερήκευση πρώτα απ' όλα είναι μια πραγματικότητα είναι αυτή που επέτρεψε στα προξενία να δέχονται υπό συνθήκες αξιοπρεπής έναν αυξανόμενο αριθμό ετούντων, είναι η εξωτερήκευση που επέτρεψε στα προξενία να επικεντρωθούν επί της εξετάσεως των, διαφόρων υποθέσεων και αυτή η εξωτερήκευση επιτρέπει να εξετάζονται περισσότερα θέματα και να δεχόμαστε περισσότερους ετούντες. Σας ομολογώ ότι δεν ήμουν ο ίδιος υπέρ της εξωτερικεύσεως στην αρχή λίγο λόγω ιδεολογίας και επίσης διότι φοβόμουν κάποιες παρεκκλήσεις. Σήμερα θα πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι η εξωτερήκευση απέδειξε ότι είναι αποτελεσματική. Εγκρίνω λοιπόν απόλυτα τις προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, που ε, έχουν αποτελέσματα και μιλάμε τώρα για την επίσης πραγματικότητα. Η εξωτερήκευση ε, δεν είναι παρά τελευταία δεν είναι πλέον η τελευταία προσφυγή, είναι η πλέον λογική προσφυγή. Η άμεση πρόσβαση των ετούντων στα προξενία προφανώς δεν είναι κάτι διαχειρίσιμο στην πράξη, εκτός ε, από ορισμένε περιπτώσεις ατόμων, των οποίων το αίτημα θεώρηση πρέπει να είναι στα πλαίσια εμπιστευτικού χαρακτήρα και τον και πρέπει να το χειριστούν σωστά τα προξενία. Και οι πάροχοι θα πρέπει όλο και περισσότερο να ελέγχονται για να απεφευχθούν οι παρεκκλήσεις. Αυτοί που δίνουν τη θεώρηση. Λοιπόν, έχουμε και διάφορε διάρκειε όσον αφορά τη θεώρηση. Ε, είδα ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είχε υποβάλει κάποιον, κάποια σειρά προτάσεων. Ε, λοιπόν, το γαλλικό προξενείο το θεωρεί αυτό θεώρηση κυκλοφορία ισχύ τη είναι ίση ή μεγαλύτερη από ένα έτος. Ε, δύσκολο να μεταφραστεί ο όρο αυτό γαλλικά, να μιλήσουμε για traffic visa. Στα γαλλικά θα έλεγα ότι είναι frequent traveler visa για τα συχνά ταξίδια, οπότε ο δικαιούχο ο κάτοχο θεώρηση έχει ελευθερία κυκλοφορία προσωρινά. Αυτή η θεώρηση θεωρώ ότι προσαρμόζεται πολύ καλή ε, σε ανθρώπους αυτούς που θεωρούμε ότι δεν αντιπροσωπεύουν μεγάλο κίνδυνο. Τώρα οι προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ακολουθούν την σωστή κατεύθυνση, αλλά ο αυτόματος χαρακτήρας της χορηγήσεως, της θεωρήσεως κυκλοφορίας το ότι είναι κάτι παρακινδυνευμένο. Από τη στιγμή όπου δημιουργείται ένα, μια, ένας αυτοματισμός υπάρχουν καταχρήσεις και πρέπει κανείς να είναι προσεκτικός και κάθε αυτόματη χορήγηση να εξαιρείται. Θα πρέπει το προξενείο να έχει το δικαίωμα να περιορίζει την διάρκεια ε, μιας θεωρήσεως ή να αρνηθεί την χορήγηση για να μπορεί να αντιταχθεί στι καταχρήσει. Κάποια προξενία ποτέ δεν δίνουν ε, αυτές τις θεωρήσεις κυκλοφορίας. Θα πρέπει να βρούμε έναν τρόπο για να του κάνουμε να το κάνουν. Για να το καταφέρουμε εγώ θα πρότεινα να δώσουμε ένα όνομα ιδιαίτερο σε αυτή των πολλαπλών εισόδων θεώρηση για ένα χρόνο ή λιγότερο ή περισσότερο. Να πούμε visa τη. circulation στα γαλλικά ή frequent traveler visa στα αγγλικά ούτω ώστε να μπορέσουν να ανταποκρίνονται στι ανάγκε πραγματικέ των προξενείων. Τη στιγμή λοιπόν όπου είναι καλά καθορισμένη αυτή η έννοια, μπορούμε να καθορίσουμε πολύ πιο εύκολα συγκεκριμένου κανόνε που θα διευκολύνει τη χορήγησή του και την ανανέωση, συγγνώμη, των θεωρήσεων. Αυτό που σα ζητούμε και σα εκλυπαρούμε είναι να πλουστεύσετε τι διαδικασίε. Βλέπω τους νέους κανόνες για τις κατεπίγουσες ανάγκες. Θα πρέπει αμέσως Βέβαια δεν είναι δυνατόν αυτό. Αν δίνουμε αμέσως ένα ραντεβού σε κάποιον ή αν έχουμε ένα πλήρες χρονοδιάγραμμα, σημαίνει ότι για να το βρούμε αυτού θέση πρέπει να πάρουμε τη θέση κάποιου άλλου. Και σε, με τι σχετίζεται το κατεπήγον. Ο καθένα έχει τη δική του αντίληψη περί του κατεπήγοντο. Ο δωρεάν χαρακτήρα, προσοχή σε αυτό, αυτό μπορεί να έχει αντίστροφα αποτελέσματα. Ιδού λοιπόν, Έκλεισα διότι είχα 10 λεπτά ακριβώς τη θέση μου, αλλά σας ευχαριστώ για την προσοχή σας. Ακριβώς. Την ώρα σας, την ώρα σας ακριβώς. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τις σκέψεις αυτές που μας παρουσιάσατε και ιδιαίτερα επειδή βασίζονταν οι παρατηρήσεις που κάνετε στις ε, εμπειρίες σας, τις ίδιες. Ο κ. Μπενισό τώρα από την από Έχετε το λόγο. σου. Θα ήθελα να ευχαριστήσω το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο που ζήτησε από την VFS Global να έρθει σε αυτή την δημόσια ακρόαση για να παρουσιάσει την τοποθέτηση των εξωτερικών παρόχων υπηρεσιών. Η εταιρεία VFS Global ιδρύθηκε το 2001. Είναι πολύ γνωστή στις κυβερνήσεις. Πρόκειται για μια θηγατρική του ελβετικού ομίλου Κόνη. Εξυπηρετεί 45 κυβερνήσεις σε 121 χώρες ε, μέσω 1.600 κέντρων. Και εξάλλου ε, μόλις κάναμε και το εκατοστό, εκατομμυριοστό ε, φάκελο για αίτηση θεώρησης σε ένα από τα κέντρα μας. Θα ήθελα να σα εξηγήσω την έννοια της εξωτερικής ανάθεση ή εξωτερήκευσης ε, που είναι σχετικά νέα. Θα ήθελα επίσης να σας παρουσιάσω τις βελτιώσεις ε, που έγιναν χάρη στην εξωτερήκευση τόσο για τις κυβερνήσει, όσο και για τους ετούντε άσυλο. Και στο τέλος θα ήθελα, αν μου επιτρέπετε, να κάνω και κάποιες προτάσεις για να βελτιωθεί περαιτέρω το νομικό πλαίσιο. αρχίσουμε πρώτα με την έννοια της εξωτερικής ανάθεσης για τις θεωρίες λύσεις, ούτως ώστε να, να μην δημιουργούνται παρανοήσει. Λοιπόν, ε, τι σημαίνει εξωτερική ανάθεση. Δεν σημαίνει ότι εκχωρείται αρμοδιότητα για τη λήψη απόφαση σε έναν εξωτερικό πάροχο υπηρεσία, όπως ορισμένοι ε, ισχυρίζονται. Η αρμοδιότητα για την έκδοση θεώρησης ε, ανήκει αποκλειστικά και μόνο στις κυβερνήσεις ε, που εκχωρούν αυτό το δικαίωμα στα προξενία. Οπότε δεν έχουν καμία αρμοδιότητα και δεν μπορούν να επηρεάσουν την ε, λήψη απόφαση για την έκδοση θεώρησης η εξωτερική πάροχη. Πρόκειται λοιπόν για, για μια λύση ούτω ώστε να αντιπεξέλθουν οι κυβερνήσεις στις νέες προκλήσεις βελτιώνοντα ταυτόχρονα τις υπηρεσίες που παρέχουμε στου ετούντε. Είναι πολλαπλέ οι προκλήσει διότι ο μεγαλύτερο αριθμό των κρατών Σέγγεν αντιμετωπίζει μία αύξηση του αριθμού αιτήσεων για θεωρήση, κυρίω από πλευρά των οπτιζομένων χωρών, οπότε χρειάζονται επιπρόσθετα μέσα. Στη συνέχεια, η προσφυγή στα βιομετρικά δεδομένα καθιστά υποχρεωτική την παράσταση, παράσταση των ετούντων, ενώ ε, σε ορισμένε χώρε χρησιμοποιούνταν ω δημοσιολαβητέ τα ταξιδιωτικά γραφεία. Οπότε χρειαζόμαστε επιπρόσθετε θηρίδε και χρειάζεται περισσότερο προσωπικό καθώ και υλικοτεχνική υποστήριξη για τη συλλογή των βιομετρικών ε, δεδομένων. Ε, προσωπική παράσταση λοιπόν, ε, έτσι έχουμε μια αύξηση τη ζήτηση των υπηρεσιών εγκύτητα όπω ονομάζονται. Επίση, εκτίθεται λένε και μεγαλύτερου κινδύνου σε τα προξενία προ την ασφάλειά του, και ο αυξημένο αριθμό αιτήσεων θεωρήσεων συνεπάγεται και αυξημένο αριθμό επισκέψεων αυξάνοντα έτσι του κινδύνου για την ασφάλεια. Λοιπόν, αναπόφευκτα αυτό συνεπάγεται πρόσθετο κόστο για το προσωπικό, για, τους, το, για τον τόπο παροχή υπηρεσιών και τι συνθήκε ασφαλεία που επικρατούν εκεί. Ταυτόχρονα όμω περικόπτει ο προπολογισμό των προξενείων που δεν μπορούν να αντεπεξέλθουν διότι ε, ε, ε, καλούνται να προσφέρουν αυξημένε υπηρεσίε με λιγότερα μέσα. Είναι μια λύση λοιπόν εξωτερική ανάθεση για να μειώσουμε το κόστο. Λοιπόν, δεν αντιβαποκρινόμαστε μόνο στα προβλήματα των ε, κυβερνήσεων, αλλά βελτιώνουμε και την ποιότητα των υπηρεσιών ε, των πελατών, δηλαδή αυτών που αιτούνται ε, την έκδοση θεώρησης. Σχηματικά μπορούμε να πούμε ότι ή τι θα κάνουμε για να αντιπεξέλθουμε στην αυξημένη ανάγκη ή θα προσαρμόσουμε τον αριθμό των ετούντων ε, στην ικανότητα υποδοχή ή το αντίστροφο. Λοιπόν, χάρη στην εξωτερική ανάπτυξη μπορούμε να προσαρμόσουμε την ικανότητα υποδοχή, ε, δηλαδή ανάλογα με τον αριθμό των ετούντων ε, που καταβάλουν το τέλο για την υπηρεσία. Οπότε, όσο ο πάροχο υπηρεσία έχει περισσότερου ετούντε, τόσο λαμβάνει αυξημένα τέλη και άρα μπορεί να επενδύσει τους ώστε να υποδεχθεί ακόμη περισσότερο σε Με την εξωτερική ανάθεση έχουμε λοιπόν μια σχέση που αναπτύσσεται ανάμεσα στον πάροχο και στον πελάτη. Ο πάροχος λοιπόν μπορεί να προσαρμόσει τα γραφεία του ε, ούτω ώστε να προσαρμόσει και το προσωπικό του στη συνέχεια ε, στα αναμενόμενο, στον αναμενόμενο αριθμό των αιτήσεων ε, θεωρήσεων. Επίσης μπορεί να προσαρμοστεί στις διακοιμάνσεις, διότι ξέρετε υπάρχουν τόσο μεγάλες ουρές ορισμένες φορές που ξεκινάει με, στη νύχτα να έρχεται ο κόσμος περιμένοντας ε, και πέφτοντα θύμα εκβιασμών ε, και άλλων παρανόμων ενεργειών και αυτό φυσικά οδηγεί σε αυξημένο κόστος. Όμως ε, για την πρόσβαση στις ειδικέ υπηρεσίες, ειδικέ θηρίδες των προξενείων, ενώ θεωρητικά δεν υπάρχει κανένα κόστος, ορισμένες φορές κόστιζε πάρα πολύ ακριβά αυτό στους ετούντες. Χάρη στην εξωτερική ανάθεση μπορούμε να οργανώσουμε καλύτερα την υποδοχή. Τα προξενεία που έχουν αναλάβει την υποδοχή του κοινού μπορούν πλέον χάρη στην εξωτερική ανάθεση να χρησιμοποιήσουν την ενέργειά του για να διεκπαιρεώσουν μεγαλύτερο αριθμό φακέλων. Οι ετούντε δεν έχουν δεχτεί και είναι πολύ ικανοποιημένοι με την εξωτερική ανάθεση. επίση. χάρη στην εξωτερική ανάθεση μπορούμε ε, να έχουμε σε κοινά κέντρα υποδοχή του κοινού για ε, πάνω από ένα κράτη ε, Σέγγεν. Χάρη στην εξωτερική ανάθεση, τα κράτη Σέγγεν επιλέγουν τον ίδιο παρόχο ορισμένε φορέ και άρα χρησιμοποιούν χώρους υποδοχής. Από πλευράς υλικοτεχνική υποστήριξης, λοιπόν, ε, τα κράτη Σέγγεν έχουν κέρδο διότι επιλέγουν κοινό πάροχο. Ε, χάρη σε αυτό, ε, ο χώρο Σέγγεν αντιστοιχεί πλέον στην ευρωπαϊκή πραγματικότητα, δηλαδή στον αυξημένο αριθμό αιτήσεων. Για τους ε, παρόχους, για να μπορέσουν να βελτιώσουν τις υπηρεσίες, ε, χρειαζόμαστε ένα ε, ευέλικτο ρυθμιστικό πλαίσιο. Ο κώδικας των θεωρήσεων εγκρίθηκε το 2009, ενώ η εξωτερική ανάθεση για τα κράτη Σέγγεν ακόμη τότε ε, το. ήταν στις αρχές. Και έκτοτε έχει μετεξελιχθεί η έννοια της εξωτερικής ανάθεσης και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει λάβει υπόψη αυτή την πραγματικότητα στις προτάσεις που κάνει και που καλωσορίζουμε. Παρ' όλα αυτά θα μπορούσε, έχετε περαιτέρω βελτιώσει στο κείμενο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής τόσο ώστε οι παρόχοι να μπορέσουν να παράσχουν ένα, μια ακόμη καλύτερη υπηρεσία στους ετούντε μια καλύτερη εφαρμογή της, του κανόνα των 59 μηνών για τη συλλογή βιομετρικών δεδομένων. Οι ετούντες που έχουν στο παρελθόν ζητήσει θεώρηση Σέγγεν και τα δεκτυλικά του υποτυπώματα έχουν καταχωρηθεί στο VIS για περίοδο μικρότερο των 59 μηνών απαλλάσσονται από την υποχρέωση συλλογή δακτυλικών δεδομένων βάσει του κώδικα θεωρήσεων. Θέλουμε να τροποποιηθεί το κείμενο ώστε η απαλλαγή να συνδέεται με την παρουσίαση από πλευρά του ετώντα Μία απόδειξη για την καταχώρηση των δακτυλικών του αποτιμάτων στο VIS για περίοδο κάτω των 59 μηνών, τόσο ώστε να μπορέσουμε εμεί ω παρόχοι να εφαρμόσουμε αυτή τη διάταξη. Θα μπορούσε αυτό να υλοποιηθεί μέσα από την παρουσίαση, παραδείγματο χάρη από πλευρά του ετούντα τη θεώρηση, όπου θα αναφέρεται ε, ότι ανήκει στο σύστημα VIS ή παραδείγματο χάρη από ένα, μια απόδειξη όταν έγινε η πρώτη συλλογή δακτυλικών ε, αποτιμάτων. τώρα στι πόλει όπου δεν υπάρχει προξενείο μπορούν να χρησιμοποιηθούν οι δορυφορικοί σταθμοί, οι οποίοι προσφέρουν μια υπηρεσία εγκύτητα, χάρη στην οποία αποφεύγεται το κόστο τη μετακίνηση, γιατί ορισμένε φορέ απέχει πάρα πολύ από το τοποκατοικία στο προξενείο έτσι, οι πάροχοι μπορούν να χρησιμοποιήσουν επιπρόσθετους πόρους ε, για ε, ένα περιορισμένο αριθμό ετών. Παραδείγματο χάρη πρόκειται για τα γραφεία, το προσωπικό, ε, το υλικό που χρειάζεται, καθώς και η μετακίνηση για την παροχή των απαιτούμενων εγγράφων και του διαβατήριου. Όμως, στον τωρινό κώδικα θεωρήσεων υπάρχουν μόνο προαιρετικά ειδικά τέλη για τις επιπρόσθετες υπηρεσίες. Ε, χρειαζόμαστε λοιπόν μια ρητή διάδεξη για το άνοιγμα τέτοιων δορυφορικών κέντρων και η πρόβλεψη αυτών των επιπρόσθετων ε, τελών ε, παροχής υπηρεσιών με ανώτατο όριο τα 30 ευρώ, ούτως ώστε να μπορέσουμε να αυξήσουμε τον αριθμό των υπηρεσιών εγκύτητας μέσα από τα δορυφορικά κέντρα. Σε σχέση τώρα με τα 30 ευρώ και τον περιορισμό αυτών των τελών υπηρεσίας. Καταρχάς, ε, δεν υπάρχει ε, διευκρίνηση αν είναι πριν ή μετά της φορολόγησης ε, αυτό το ποσό των 30 ευρώ. Εμείς θα θέλαμε να αναφέρετε ότι πρόκειται για 30 ευρώ προφορολόγησης, ούτως ώστε να έχουμε μια ισχυρή οικονομική βάση και να μπορέσουμε επ' αυτής να οικοδομήσουμε τις νέες υπηρεσίες που θα προσφέρουμε. Αυτό το ποσό διορίστηκε, ορίστηκε συγγνώμη, το 2008. Όμως, έκτοτε σε πολλά κράτη έχει απογειώσει μειωθεί ο Το κόστος των νοικίων για τα γραφεία μας, παραδείγματος χώρε που βρίσκονται, ε, τα γραφεία είναι πλέον απαγορευτικό και επίσης ε, η, με βάση της ε, μεστολογικής νομοθεσίας δεν μπορούμε να έχουμε το κατάλληλο εκπαιδευμένο προσωπικό με τις παλαιότερες διατάξεις. Επίση, χρειαζόμαστε νέο υλικό για συλλογή βιομετρικών δεδομένων, ψηφιοποίηση των φακέλων, ε, ηλεκτρονική αρχαιοθέτηση ε, και ούτω καθεξή. Ε, χρειάζονται αυξημένοι έλεγχοι επίση λόγω των τεχνολογικών καινοτομιών και νομίζουμε ότι θα πρέπει να επιδιωχθεί μια αύξηση των του ωρίου ορίου των 30 ευρώ, ώστε διαρκώ να συνεχίσουν να αυξηθούν βελτιώνονται οι υπηρεσίε που προσφέρουμε σε αυτού του ετούντε. Για να μην υπερβώ τα 10 λεπτά, κλείνοντα, θα ήθελα να σα πω ότι ε, ό,τι περνάει από το χέρι μα το κάνουμε, χρησιμοποιούμε όλα τα πετούμενα μέσα και ό,τι μέσα έχουμε στη διάθεσή μα για να εξυπηρετήσουμε τι ανάγκε των κυβερνήσεων αλλά και των ετούντων. Θα ήθελα να σα ευχαριστήσω για την προσοχή που δείξατε. Thank you. Thank you very much. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και τώρα θα συνεχίσουμε με την κυρία Μροζέκα από την συνασπισμό για την Ευρώπη χωρίς ε, θεωρήσεις και θα με παρουσιάσετε τις ε, εμπειρίες των υποβάλλοντων ε, αιτήματα των ετούντων θεωρήσεων. Σα ευχαριστώ κύριε και κύριε για την ευκαιρία που μου δίνετε να συμμετάσχω σε αυτέ τι διαβουλεύσει, σε αυτή την ακρόαση και όπω ξέρετε η πρόταση με το θέμα των θεωρήσεων. Ονομάζομαι Κρίστοφ Μρόζεκ και εκπροσωπώ τη Visa Free Europe Coalition για μια Ευρώπη χωρί ε, θεωρήσει από την Πολωνία. Θα πρέπει να σα πω ότι οι προτινόμενε αλλαγέ στην υφιστάμενη νομοθεσία συμπεριλαμβανομένων και των παρατηρήσεων που έγιναν από την κυρία Φαγιόν νομίζω ότι κινούνται προ τη σωστή κατεύθυνση. Εν μέρη διαφωνώ με αυτά που είπαν οι συνάδελφοι, οι προηγούμενοι συνάδελφοι για το outsourcing. Θεωρώ ότι θα πρέπει να είναι μια πρόσφατη λύση, όχι η βασική μας προσέγγιση στο θέμα της, ε, των θεωρήσεων. Θα πρέπει να αναζητήσουμε λύσεις που δεν δημιουργούν επιπρόσθετο κόστος για τους ετούντες θεώρηση. Επί τέσσερα χρόνια ε, έχουμε ένα πρόγραμμα με πληροφοριοδότες, ε, άτομα τα οποία δεν είναι ικανοποιημένα με τον τρόπο που αντιμετωπίστηκε η αιτήσή τους για τις θεωρήσεις. Μας γράφουν λοιπόν ανώνυμα τα παραπονά τους. Χιλιάδες τέτοια παράπονα ενστάσεις λάβαμε κάθε ένα εκ των οποίων ήταν πραγματικά δραματική υπόθεση. Θα ήθελα λοιπόν σήμερα να σα πω ότι πίσω από τον κανονισμό αυτόν, πίσω από τις νομοθεσίε που συζητιούνται, είναι πραγματικοί άνθρωποι, κρύβονται πραγματικοί άνθρωποι που ζητούν θεωρήσει και η ιστορία του η ζωή του. και βάσει των ιστοριών αυτών λοιπόν θα ήθελα να εντοπίσω τρία βασικά προβλήματα στην υφιστάμενη νομοθεσία και να προτείνω κάποιε αλλαγές. Πρώτον, πρώτη πρόκληση που αντιμετωπίζουν οι ετούντες θεώρηση είναι το θέμα των, πολλαπλών θεωρήσεων, των πολλών θεωρήσεων πολλαπλής εισόδου για με μικρό διάστημα. Μας είπε λοιπόν ένας ε, πληροφοριοδότης ότι έκανε αίτηση για θεώρηση, ήταν μια θεώρηση πολλαπλής εισόδου, για, ουσιαστικά όμως για μία είσοδο και ενώ είχε πρόσκληση για 34, 34 μέρες, έλαβε βίζα για 34 μέρες. Ένας εκτίμησης από την Ουκρανία, μια άλλη ιστορία. Μια εκτιμήθεια, λοιπόν ζήτησε για μια, μια τριετή θεώρηση παραπλής εισόδου, την οποία και δικαιούταν με την ιστορία που είχε. αλλά τη θεωρούσαν ε, θεώρηση ενός ατούς. Δεν ακολουθήθηκαν δηλαδή οι συστάσεις ε, της πολιτικής ε, για τις θεωρήσεις. Η δική μας σύσταση λοιπόν είναι να εισαχθεί μια κατηγορία VAS τακτικών ταξιδετών με θεωρήσει δηλαδή πολλαπλής εισόδου και να εξετάσουμε το ενδεχόμενο κατηγορίας ε, θεωρήσεων 10 ετών. Ε, σύστημα το οποίο έχει εφαρμοστεί στην Αμερική χωρίς ε, πρόβλημα. Δεν υπάρχει λόγος να υπάρχει περιορισμός πενταετής για τις θεωρήσεις. Και αυτό θα έχει θετικό αντίκτυπο και στο φόρτο εργασία στα προξενία. Και στις ουρές που φυσικά υπόκειται ο κόσμος. Δεύτερη πρόκληση η πολύ προβληματική διαδικασία εφαρμογή. Δεν πολύ πρόβλημα η συνέντευξη με τον πρόξενο, είναι η κατάθεση της αίτηση στο προξενείο ή στο κέντρο θεωρήσεων. Συχνά δεν υπάρχουν για δύο-τρεις μήνες χρονοθυρίδες στο προξενείο ή στο κέντρο θεωρήσεων. Άλλη μία κατάθεση. Είναι αδύνατον να καταθέσει κανεί αίτηση χωρί επιπρόσθετα έξοδα Ε, δεν κατάφερα να καταχωριστώ ε, και να γραφτώ στο προξενείο. Και πάλι κάθε φορά μου δίνουν διαφορετικέ εξηγήσει. Μια τρίτη κατάσταση, ε, το πολωνικό προξενείο στο ΔΙΒ καθιστά αδύνατη την κατάσταση αιτήσεων χωρί να χρησιμοποιηθούν ύποπτη πάροχή υπηρεσιών. Και θα μπορούσε να εισαχθεί επίση ένα σύστημα online. Υποστηρίξαμε τέτοια συστήματα άλλωστε. Θα θέλαμε να δούμε, θα θέλαμε να υπάρχουν νομικά μέσα, νομικά εργαλεία για να εξασφαλιστεί η δυνατότητα υποβολή αίτηση για θεωρήσει κατευθείαν στο προξενείο, όπω ορίζεται από τον κωδικά για τι θεωρήσει. Γιατί στην Ουκρανία αυτό παραμένει ω θεωρητική. Παραμένει θεωρητική δυνατότητα. Στην πράξη δεν είναι δυνατόν στην πράξη επιβαρύνονται με επιπλέον χρέωσεις οι ετούντες. Τελευταία πρόκληση την οποία θα ήθελα να επισημάνω είναι η υπόθεση το θέμα των ε, ε, εγγράφων τεκμηρίωσης. Ε, ζητούνται πάρα πολλά, υπερβολικά πολλά έγγραφα από τις αρχές του προξενείων και υπερβολικά πολλές εξηγήσει ε, για το σκοπό της ε, θεώρησης που ζητείτε. Άλλη μια κατάσταση ενό ε, Αρμενίου που ήθελε να δουλέψει ως οθελοντής στη Γερμανία. Του ζητήθηκε λοιπόν να καταθέσει στα γερμανικά ένα, μια επιστολή για τους λόγους που τον οδηγούν στην εθελοντική αυτή εργασία, ενώ η βίζα ήταν στα αγγλικά. Η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής προτείνει έναν εξαιρετικό κατάλογο υποστηρικτικών εγγράφων. Αυτό θα πρέπει να το υποστηρίξουμε. Αλλά παράλληλα να εξασφαλίσουμε ότι ο εξαιρετικό αυτός κατάλογος δεν θα καλύπτει όλα τα δυνατά έγγραφα τα οποία ενδεχομένω να ζητηθούν από τις προξενικές αρχές. Αυτό το είδαμε στην Ουκρανία πέρυσι όταν δημοσιεύτηκε ο κατάλογος. Ουσιαστικά περιλαμβάνονται όλα τα δυνατά έγγραφα. Και οι Ουκρανοί ετούντες παραπονιούνται γιατί τα πολωνικά προξενία ζητούσαν λίγα έγγραφα, τώρα πλέον ζητάνε πιο πολλά βάσει του καταλόγου υποστηρικτικών εγγράφων. Τέλος για να συνοψίσω. Να ακούσουμε άλλον έναν πληροφοριοδότη, μια δραματική ιστορία την οποία μοιράστηκε το άτομο αυτό μαζί μας. Είπε λοιπόν το άτομο αυτό ότι ακόμα δεν κατανοώ γιατί οι Ουκρανοί ε, αποτελούν αντικείμενο έχθρας και μίσος. Εγκληματίες είμαστε, παράνομοι μετανάστες. Γιατί τέτοια στερεότυπα. Αυτό ακούγεται σχεδόν, αυτό ακούγεται ναζιστικό και όταν τα γράφω αυτά, ένα πράγμα έχω στο μυαλό μου. Ελπίζω οι σύνοντες, αυτοί που ε, λαμβάνουν αποφάσει και που θα διαβάσουν ε, την κατάσταση αυτή, θα προσπαθήσουν να διαμορφώσουν με διαφορετικό τρόπο ε, τι εργασίε αυτές και να είναι ο κόσμος λίγο πιο φιλικός με τον συνάνθρωπό του. πραγματικά προβληματίστηκα για το κατά πόσο θα συμπεριλάμβανα αυτή την αναφορά στους Ναζί. Είναι πραγματικά υπερβολικό ίσως. Αλλά αυτό δείχνει πόσο απολυπισμένος είναι ο κόσμος. Και πόσο πέφτει η Ευρωπαϊκή Ένωση στα μάτια τους. Επειδή είναι τόσο αναποτελεσματική η πολιτική για τις θεωρήσεις. Να σας ευχαριστήσω για την προσοχή σας και σας παρακαλώ όταν εγκρίνουμε την νέα νομοθεσία, α έχουμε υπόψη μα ότι είναι πραγματικοί άνθρωποι που κρύβονται πίσω από τι παραγράφου αυτέ που εγκρίνετε εσεί. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ, λέει πρόεδρο Και τώρα το, ρόλο, το λόγο έχει η κυρία Γεωργάλη από το European Youth Forum. Έχετε το λόγο. Και θα μα παρουσιάσετε τι απόψει των ε, ενό νέων. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρο. σα ευχαριστώ για την πρόσκληση στο Ευρωπαϊκό Youth Forum. Φόρουμ της Νεολαίας, όπως και ο προηγούμενος συνάδελφος ε, σας παρουσίασε την πλευρά των ετούντων. Εγώ θα είμαι πιο συγκεκριμένη. Θα σας ε, παρουσιάσω την άποψη των νέων ετούντων. Το European Youth Forum αποτελεί μια πλατφόρμα που εκπροσωπεί οργανώσεις για τους νέους στην Ευρώπη. Έχουμε περίπου 100 μέλη και μεγάλο ποσοστό αυτών είναι οργανώσεις που οργανώνουν ανταλλαγές, εργασία, των νέων που συχνά σε πολλέ περιπτώσει περιλαμβάνουν κινητικότητα, δηλαδή μετακίνηση των νέων ατόμων στην Ευρωπαϊκή Ένωση και σε παγκόσμιο επίπεδο. Αυτό ασφαλώ επηρεάζει τον τρόπο εργασία πολλών οργανώσεων. Και για να σα εξηγήσω τι θα σας παρουσιάσω, δεν θα επισέλθω τόσο πολύ σε οικονομικέ ε, συνέπειε τη αλλαγή διαδικασία θεωρήσεων ξέρουμε και έχουμε διαβάσει διάφορες μελέτες για το θέμα αυτό. Αυτό που θα ήθελα εγώ να σας παρουσιάσω είναι ο βραχυπρόθεσμος αντίκτυπος, ο μακροπρόθεσμος αντίκτυπος. Ο αντίκτυπος των ανταλλαγών αυτών των νέων, τη συνεργασία των νέων με νέους από διαφορετικό ιστορικό υπόβαθρο, από διαφορετικές χώρες, από διαφορετικούς πολιτισμούς, τον ε, διαπολιτισμικό διάλογο που προκύπτει και τις διαπολιτισμικές συνταλλαγές που προκύπτουν, ιδιαίτερα εν ώψη του κινδύνου ριζοσπαθικοποίησης των νέων. Είναι λοιπόν μια σημαντική λύση αυτή για ένα ευρωπαϊκό και παγκόσμιο ζήτημα. Να σας πω λοιπόν ποιο είναι το πλαίσιο σήμερα. Όλοι ακούμε πολλά για την κατάσταση με την απασχόληση των νέων ε, στην Ευρώπη. Αυτό αποτελεί μακροπρόθεσμο πρόβλημα και χρήζει ασφαλώς μακροπρόθεσμων λύσεων. Η διευκόλυνση όμως των μετακινήσεων των νέων στην Ευρώπη και σε παγκόσμιο επίπεδο όντως μπορεί να βοηθήσει και το θέμα της ανεργίας. Ε, πραγματοποιήθηκε πρόσφατα μια έρευνα που καταδεικνύει ότι οι ικανότητες που κερδίζουν οι νέοι από τέτοιες ανταλλαγές, από εργασία στο εξωτερικό, από προγράμματα κινητικότητας, είναι κάτι το οποίο ε, τους κάνει ε, επιθυμητούς από τους εργοδότες. Να σας δείξω λοιπόν το ευρύτερο πλαίσιο της συζήτησης σήμερα, πρώτο περάσω στα θέματα του κώδικα για τις θεωρήσεις και για την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Κάποιες προτάσεις ε, είναι υποτροποποίηση και καταρχάς θα ήθελα να ευκρινίσω ότι καλωσορίζουμε την ε, πρόταση. Εμείς ως εκπρόσωποι των ε, ενώσεων των νέων αποτελεί ένα πάρα πολύ καλό βήμα για να διασφαλίσουμε και να προωθήσουμε την κινητικότητα των νέων στην Ευρώπη. Αλλά θα θέλαμε και πιο πολλά και θα αναφέρω κάποια από τα ζητήματα που ήδη έχουν συζητηθεί και θα είναι σημαντικό να επανέλθουμε σε αυτά και από την οπτική γωνία των νέων και το πόσο μπορούν να ωφελήσουν τον νέο, τους νέους. Το πρώτο στοιχείο λοιπόν για τα τέλη θεωρήσεων και υπηρεσιών. Εμείς ζητούμε να μην υπάρχουν τέλα για τους, τέλτα, για τους εκπροσώπους των μη κυβερνητικών οργανώσεων και των μη των ε, οργανώσεων με μη κερδοσκοπικό σκοπό και για τα άτομα κάτω των 35. Γιατί διαλέγουμε λοιπόν την ηλικία των 35, γιατί έτσι έχει πραγματικότητα στην Ευρώπη και σε παγκόσμιο επίπεδο σήμερα. Αυτή η περίοδος της νέότητα μπορεί να φτάσει μέχρι εκείνη την ηλικία. Οι νέοι καθυστερούν σε ό,τι αφορά την μετάβασή τους στην αυτονομία, στην εξαρτησία. και θεωρούμε ότι αυτό πρέπει να αποτυπώνεται και αν προκειμένου στην νομοθεσία. Έχουμε πολλές ε, μελέτες από τις οργανώσεις μας που οργανώνουν ανταλλαγές και φιλοξενούν νέους και οι τρέχουσες εξαιρέσεις για τις θεωρήσεις δεν εφαρμόζονται και αυτό θα πρέπει ε, να επιληθεί ως ζήτημα καλύτερη παρακολούθηση της εφαρμογής προκειμένου να μην υπάρχουν τέτοιες παρατυπίες στις ε, αιτήσει. Να περάσουμε τώρα σε ένα άλλο ζήτημα. Το θέμα των ε, σε ό,τι αφορά το θέμα των δικαιολογητικών, των παστατικών. Είναι καλό να υπάρχει γραπτός κατάλογος και έχουμε δει διάφορες περιστάσεις όπου η απόρριψη των θεωρήσεων δικαιολογείται με έλλειψη τέτοιων δικαιολογητικών. Πολλοί ετούντε ε, είναι από την Αφρική σε γενικέ γραμμέ για την Ευρώπη και σε πολλές περιπτώσεις του ζητείτε να αποδείξουν ότι είναι παντρεμένοι. Αυτό θεωρούμε ότι αποτελεί διακριτική μεταχείριση βασιλικία. Γιατί οι νέοι που συμμετέχουν σε τέτοιες ανταλλαγές δεν είναι απαραίτητα παντρεμένοι. Και αυτό συχνά επικαλείται ως λόγος απόρριψης της θεώρησης. Αυτό λοιπόν θα πρέπει να επιληθεί και μάλιστα με ένα γενικό και συνεκτικό τρόπο. Και αυτό με οδηγεί σε ένα πιο ευρύ ζήτημα για τη διακριτική μεταχείριση βασιλικίας. Σε πολλές περιπτώσεις βλέπουμε αδικαιολόγητες απορρίψεις αιτήσεων βάση ηλικία και μόνο ή καταστάσεων που συνδέονται με την νεότητα. Αυτό πραγματικά είναι παράδεκτο. Και τέτοιες πρακτικές ε, από τα κράτη-μέλη αποτελούν παραβίαση του άρθρου 21 του Χάρτη των Ανθρωπινών Δικαιωμάτων, των θεμελιωδών δικαιωμάτων. Θα πρέπει να αποτυπώνεται αυτό λοιπόν στην τρέχουσα νομοθεσία. Για το ζήτημα τώρα των κοινών κέντρων αιτήσεων. Και αυτό αναφέρθηκε. Και πάλι έχουμε πάρα πολλέ γελιότητε να σα αναφέρουμε. ναι, οι οποίοι αναγκάζονται να ταξιδεύουν χιλιάδε χιλιόμετρα για να κάτσουν ε, τρει-τέσσερι νύχτε και αναγκάζονται να χρεωθούν και το ταξίδι και τα έξοδα ξενοδοχείου πέρα από τα τέλη θεωρήσεων και τελικά είναι πολύ απλά αδύνατον για άτομα που δεν έχουν χρήματα να συμμετέχουν σε τέτοια προγράμματα κινητικότητα. Θέλουμε κοινά κέντρα λοιπόν αιτήσεων για να είναι κεντρική και απλή η μέθοδος υποβολής αίτησης θεωρήσεων. Τέλος, έχουμε φυσικά μακρύ κατάλογο προτάσεων, αλλά θα τη συζητήσουμε αργότερα. Θα ήθελα να κλείσω αναφέροντας κάτι που πραγματικά επηρεάζει τις οργανώσεις μας. Αυτή η πρόταση για μια διαδικασία ταχείας ε, αντιεκπαιρέωσης, fast track, για, τους, ε, για τα μέλη κοιό και ε, μη κερδοσκοπικών οργανισμών. Θα θέλαμε συγκεκριμένα να αναφέρονται αυτές οι οργανώσεις μη κερδοσκοπικού σκοπού ως τμήμα των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων Γιατί συχνά αυτές οι θαυμάσιε ευκαιρίες για εκπαίδευση, μετεκπαίδευση και εργασία των νέων διακυβεύονται λόγω των τεράστιων καθυστερήσεων και της τεράστιας διαρκείας των ειδικασιών. Θα κλείσω στο σημείο αυτό και νομίζω ότι ο προηγούμενος συνάδελφος παρουσίασε την πλευρά του Ετούντα τα ρίσκα που παίρνουμε, τον κίνδυνο που διατρέχουμε αν δεν εξετάσουμε στην τρέχουσα αναθεώρηση του κώδικα θεωρήσεων την ευκαιρία που δίδεται στους νέους να έρθουν στην Ευρώπη, να αναπτυχθούν, να αναπτύξουν τις κοινωνίες μας και να συμβάλλουν στο ευρωπαϊκό έργο. Ευχαριστώ. Thank you. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και τώρα για το θέμα του τουρισμού τώρα. Ο κύριος Προύστη έχει το λόγο. έχει το λόγο. Κυρία Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, αξιότιμα μέλη του Κοινοβουλίου, καλησπέρα. Ευχαριστώ που μου δίνετε το λόγο, που δίνετε το λόγο για να είμαι στο, στον τομέα που είναι ο τρίτος συνεισφορέας στο ΑΕΠ Ευρωπαϊκό. Σήμερα το απόγευμα, κυρία Πρόεδρε, συζητήσουμε απλώς διαδικαστικά ζητήματα και μέτρα που θα εφαρμοστούν για να διευκολύνουν την έκδοση θεωρήσεων, το διακύβευμα, είναι το μέλλον της ανάπτυξης του ευρωπαϊκού τουριστικού τομέα. Πριν μπω σε αυτό το τμήμα της παρουσιάσεως μου, θα ήθελα Εν συντομία να παρουσιάσω τον οργανισμό μας, αυτόν που εκπροσωπώ, το NET, είναι το δίκτυο του Ευρωπαϊκού Ιδιωτικού Τομέα στον Τουρισμό. Ομαδοποιούμε και συναθρίζουμε 7 σημαντικούς φορείς των αλυσίδων των τουριστικών στην Ευρώπη από εταιρείε κρουαζιερών, λεωφορείων, πούλμαν, ταξί, τις ε, συνδέσεις ε, των ε, πάρκων Λούνα Πάρκ και λοιπά και των πάρκων αναψυχής, ξενοδοχείων, εστιατορίων, καφενείων και την Ένωση Τουρισμού της Ευρώπης και επίσης το Σύλλογο Κατασκηνώσεων και Διαφόρων Πάρκων και επίσης και τα ταξιδιωτικά γραφεία και τις ενώσεις των διαφόρων τουριστικών εταιριών που εκπροσωπώ. Εκπροσωπώ όλους αυτούς. Λοιπόν, Σήμερα το απόγευμα έχουμε την εξή πρόκληση, που είναι και ριζοσπαστική πρόκληση. Ο τουρισμός στην Ευρώπη συμβάλλει στο 10% του ευρωπαϊκού ΑΕΠ. Παρέχουμε πάνω από 10 εκατομμύρια θέσεις απασχόλησης στην Ευρώπη. Ο τουρισμός είναι ο τρίτος, η τρίτη σε μέγεθος οικονομική δραστηριότητα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και κάτι πιο σημαντικό. Τα τελευταία έξι χρόνια Τώρα που η Ήπειρός μας αντιμετώπιζε άνευ προηγουμένου οικονομική και χρηματοπιστωτική κρίση, ο τουρισμός ήταν ένας από τους ελάχιστους τομείς που άντεχε στην κρίση. Και εμπιστευτείτε με, αυτό ήταν ιδιαίτερα σημαντικό για τα κράτη-μέλη εκείνα που επλήγησαν πιο πολύ από την χρηματοπιστωτική και οικονομική κρίση. Βλέποντας λοιπόν το που βρισκόμαστε σήμερα. Είμαστε υπαριθμόν ένας προορισμός στον κόσμο. Σταδιακά όμως χάνουμε μερίδιο της αγοράς. Και αν δείτε το γράφημα πίσω μου, ε, βλέπετε ότι η Ευρώπη εξακολουθεί να είναι νούμερο ένα, αλλά άλλες περιοχές του κόσμου κερδίζουν, κερδίζουν μερίδιο της αγοράς. Άρα πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι δεν κλείνουμε τις πόρτες μας σε βασικές αγορές που είναι οι πρώτοι συντελεστές για τον τουρισμό στην Ευρώπη, όπως είναι η Κίνα, όπως είναι η Ινδία και διάφορες άλλες χώρες της Νότιο-Ανατολικής Ασίας, όπως η Ρωσία. Δεν θα, σα σας εκπίσει το γεγονός το ότι σας λέω ότι όταν υπάρχει στον κόσμο τουρισμό, τουριστικός προορισμός που θα περιπλέξει πολύ τις θεωρήσεις, οι τουριστικές εταιρείες θα φύγουν. Θα βρουν καλύτερες εναλλακτικέ λύσεις για να προσφέρουν στους καταναλωτές τους. Βλέποντας διάφορα δημοσιεύματα, όπως πρόσφατη μελέτη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, τι βλέπουμε. Βλέπουμε ότι αν οι διαδικασίες για την θεώρηση γίνουν πιο εύκολες, αυτό θα μπορούσε να παράγει πάνω από 25 δισεκατομμύρια ευρώ παραπάνω εισόδημα για τον τομέα στην Ευρώπη και θα, θα δούμε αύξηση 13, κατά 13 με 14 εκατομμύρια επισκέπτες από άλλες χώρες. Αυτό είναι το πλαίσιο λοιπόν και γι' αυτό καλωσορίσαμε την πρόταση Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τους λόγους που προανέφερα. Καλωσορίσαμε τη δέσμη μέτρων για τις θεωρήσεις. Είναι σημαντικό να σημειώσουμε ότι δεν είναι μόνο ο τουριστικός τομέας που καλωσορίζει τη δέσμη μέτρων, αλλά και τα συνδικάτα. Διότι τα συνδικάτα καταλαβαίνουν ότι πράγματι η δέσμη μέτρων για τις θεωρήσεις θα τονώσει την απασχόληση στον τουριστικό τομέα. Και όλα τα κράτη-μέλη, όλες οι κυβερνήσεις θέλουν αύξηση της ε, απασχόλησης. Τι περιμένουμε λοιπόν από αυτή τη δέσμη μέτρων για τις θεωρήσεις. Βασική προτεραιότητα, αγαπητά μέλη του Κοινοβουλίου, είναι η αίτηση για θεώρηση να πρέπει να είναι σαφής, απλή, προσβάσιμη, φθηνή και αποτελεσματική για τον τομέα και για εκείνους που εργάζονται στον τομέα και όλος ιδιαίτερος για τους ναυτικούς. Αυτό που μας αρέσει στη διευθυντική πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι η πρόταση που αφορά την αύξηση της προξενικής κάλυψης, τη διευκόλυνση για τους τακτικούς ταξιδιώτες μέσω θεωρήσεων πολλαπλών εισόδων, η μείωση του χρόνου επεξεργασίας, η κατάργηση της ιατρικής ασφάλισης κλπ. Όλες αυτές οι προτάσεις έχουν σημασία απόλυτη ούτω ώστε η διαδικασία χορηγής θεωρήσεων να απλουστευτεί. Άκουγα με τα μεγάλο ενδιαφέροντο. Τα εισαγωγικά σχόλια τη ηγετρίας τη κυρία Φαγιών. Να σας πω ότι σα στηρίζουμε, είμαστε πίσω σας. Και θα χαρούμε να συνεργαστούμε μαζί σας. Διότι κάνατε σημαντικότατε προτάσει. Εντάχει, να διατρέξω κάποιες προτάσεις που θα θέλαμε να κάνουμε. Πρώτα απ' όλα, όσον αφορά τον ορισμό του τακτικού ταξιδιώτη. Θα θέλαμε αυτός ο ορισμός του regular traveler να συμπεριλαμβάνει κριτήρια. Δηλαδή, αν, αν είναι καταχωρημένο στο σύστημα VIS, να μπορούν να έχουν θεωρήσει για πολλαπλές ε, εισόδους και να μειωθούν οι διατυπώσεις τα σημερινά μέτρα θα αποκλείουν όμως τους τακτικούς ταξιδιώτες που ήδη έχουν λάβει θεώρηση μακράς διαρκείας ή θεώρηση για παραμονή μακράς διαρκείας τύπου D και άδεια διαμονής. Όλα αυτά πρέπει να συμπεριλαμβάνονται στα κριτήρια. Εξίσου, όσον αφορά την προξενική κάλυψη, υποχρεωτική παρουσία είναι πρόσδεκτη θα πρέπει να επεκταθεί ούτω ώστε ο ετών όχι μόνο να μπορεί να προσφεύγει σε αρμόδιες χώρες αλλά δεν εκπροσωπείται το κράτος μέλος και αν η απόσταση από το προξενείο είναι πάνω από 500 χιλιόμετρα θα πρέπει να επιτρέπεται η ευελιξία να μπορεί δηλαδή ο ετών να χρησιμοποιεί άλλο προξενείο κράτους μέλους. Μια άλλη σημαντική πτυχή ε, που μπορεί να θεωρηθεί σαν θέμα μικρής ζώνης, λεπτομέρεια, αλλά δεν είναι, αφορά ένα κομμάτι του τουριστικού τομέα που αυξάνεται με τους ρυθμούς. Μιλώ τώρα για τις κουραζιέρες. Στα κουραζιερόπλια έχουμε πολλούς ναυτικούς από τίτες χώρες. Αυτοί χρειάζονται θεωρήσεις Σέγγεν για να μπορέσουν να μπαρκάρουν στο κουραζιερόπλιο στο οποίο θα εργαστούν. Πρέπει αυτό να καλυφθεί συγκεκριμένα το θέμα των ναυτικών. Παραδείγματο χάρη, να μπορούν να υποβάλουν αίτηση θεωρήσεω μέχρι 12 μήνε πριν να ξεκινήσει η, η επίσκεψη, να συμπεριλαμβάνονται στο... αρχείο τακτικών ταξιδιωτών του VIS, αν έχουν πάρει μια θεώρηση για 12 μήνο, δοθέντως ότι έχουν εποχιακή απασχόληση, άρα θα χρειαστούν πάνω από μια θεώρηση κατά τη διάρκεια της εποχής. Δεν θα αναφερθώ στις άλλες απαιτήσει γιατί είναι τεχνικές λεπτομέρειες. Έχετε υπόψη παρακαλώ ότι οι ναυτικοί ελέγχονται τη στιγμή που προσλαμβάνονται. Ελέγχονται για λόγους ασφαλείας όταν μπαρκάρουν και ελέγχονται όταν αποβιβάζονται από τα σκάφη μετά την εκτέλεση των καθηκόντων. Αυτό λοιπόν θα πρέπει να λαμβάνετε υπόψη. Κυρία Συγγήτρια, με τα χαράς να κάνω και σχετικές προτάσεις για τα διάφορα δικαιολογητικά που απαιτούνται και κυρίως όταν αφορά την απόδειξη επαρκών οικονομικών μέσων για τη στέγαση και θα προτείνω σχετική τροπολογία. Να προσέξουμε ιδιαίτερα πρέπει την κοινή στο σελίδα του Σέγγεν, τις γλώσσες, δεν μιλούν όλοι τα αγγλικά, διασυνδέσεις ε, και διευθύνσεις για τα προξενία των κρατών μελών, αυτό θα διευκολύνει τους ετούντες. Σας ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε για την προσοχή σας. Κλείνοντας, να πω κάτι. Προσπάθησα να το υπογραμμίσω και επαναλαμβάνομαι τώρα. Είναι οικονομικό ζήτημα που διακυβεύεται. Δεν είναι μόνο ένα διοικητικό μέτρο, ένας κανονισμός. Ευχαριστώ, λέει Πρόεδρος. Έχουμε άλλους τρεις ομιλητές. Κύριο Μπέρ, Κάρκοφ και Γκούρθεμπεργκ. Αν δεν σας πειράζει, μείνετε εκεί που είσαστε, στη θέση σας, κύριε Γκιμπέρ, Ευρωπαϊκή Ένωση για την υπεράσπιση ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Θα συγκεντρωθούμε στο θέμα των ανθρωπιστικών θεωρήσεων. Ευχαριστώ. Είμαι ο Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την υπεράσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Ε, πάνω από 29.000 άνθρωποι τα τελευταία 20 χρόνια πέθαναν ε, στα σύνορα ε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης από το 2015 σχεδόν 2.000 στη Μεσόγειο. Πρόκειται για μια επαναλαμβανόμενη τραγωδία που στις 25 26 Ιουνίου θα συζητηθεί από τους κρατών και κυβερνήσεων. Στις 10 Ιουνίου είχαμε τα τελευταία στατιστικά στοιχεία και ε, και βλέπουμε ότι πρόκειται 105.000 άνθρωποι σε σχέση με τους 215.000 ε, για το 2014 προσπαθούν να μπουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Παρ' όλα αυτά, ε, παρά τη μείωση, μας λένε ότι υπάρχει εκθετική αύξηση και ότι υπάρχει φοβερή πίεση, ενώ τα στατιστικά τυχαία άλλο δείχνουν. Βλέπουμε λοιπόν ότι με πλημελή στατιστικά στοιχεία δεν μπορούμε να μιλάμε συγκεκριμένα για αυτά που συμβαίνουν στη Μεσόγειο και πιο συγκεκριμένα στα εξωτερικά σύνορα τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Πρόκειται για ζητήματα ε, ζωή ή θανάτου και οι θεσμικά όργανα τη Ευρωπαϊκή Ένωση φαίνεται ότι δεν συμφωνούν ω προ την ιεράρχηση των προτεραιοτήτων, ε, όπου πρώτη προτεραιότητα θα πρέπει να είναι η διάσωση των ε, ανθρώπινων ζωών. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα κράτη-μέλη παρόλα αυτά δεν είχαν δυσκολία να συμφωνήσουν για την ενίσχυση των συστημάτων ασφαλεία που ευθύνουν σε μεγάλο βαθμό για την απώλεια ζώων και ο Frontex μπορεί πλέον ένοπλα να παρεμβαίνει και ξέρετε ότι αυτό αμφισβητείται από χώρες ε, γύρω από τη Μεσόγειο όπως από τη Λιβύα παραδείγματος χάρη και αυτό με φέρνει στο θέμα μου. Στι ανθρωπιστικές θεωρήσεις, η πρώτη Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, για τις ε, θεωρήσεις εστιάζεται στα τεχνικά ζητήματα. Παραδείγματος χάρη πώς πρέπει να γίνουν πιο αξιόπιστες θεωρήσει, να είναι πιο αποτελεσματική έλεγχη και όταν φτάνουν οι υπήκοοι τρίτων χωρών στα σύνορα τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Ε, ξέρουμε ότι είναι πολύ μεγάλη πρόκληση για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, διότι ε, υπάρχει και το πακέτο των ευφυών σύνορων που αναμένεται. Όμω, τέλο πάντων, δεν θα ασχοληθώ με αυτό, γιατί δεν είναι το αντικείμενο τη παρέμβασή μου. Αυτό που θέλω να σχολιάσω είναι η τραγωδία των χιλιάδων ανθρώπων που προσπαθούν να μπουν στη γη τη επαγγελία ε, και για να το κάνουν αυτό περνάνε από επικίνδυνε ατραπού, διότι ακριβώ δεν έχουν την απατούμενη θεώρηση. 31 με 2015 ε, στο Κουβέιτ. Εκεί ανέλαβαν ε, τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης να δώσουν 1,1 δισεκατομμύρια για το τραγωδία των προσφύγων στη Συρία. Είναι το τριπλάσιο ποσό σε σχέση με το 2014 και το μεγαλύτερο στην ιστορία. Πολύ ωραία. Αλλά δεν μπορούμε έτσι να προστατεύσουμε μόνο τους Σύρους πρόσφυγες, ε, δεν μπορούμε να τους βοηθήσουμε να επανέλθουν σε μια φυσιολογική ζωή ακόμη και μακριά από την πατρίδα τους. Λοιπόν, οι ανθρωπιστικές θεωρήσεις εκδίδονται από την πρεσβεία ή από ένα προξενείο βάσει κριτηρίων εθνικών που δεν απαριθμούνται στον κώδικα των σύνορων τη Ευρωπαϊκής Ένωσης, ούτως ώστε να μπορέσει κάποιο να φύγει από τη χώρα του και να επιζητήσει την διεθνή προστασία σε κάποιο κράτος μέρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι απλή διαδικασία, όμως δεν ακολουθείται από τα κράτη-μέλη. Η Επίτροπος Μάλμστρομ στο Συμβούλιο Τζάι ε, το Σεπτέμβριο του 2013 όπως συζητήθηκε το θέμα της ε, Task Force ε, της Ευρώπης, ε, βλέπουμε ότι υπάρχει ένα σοβαρό αντίτυπο και τα κράτη-μέλη προσπάθησαν, όχι να διεκο... ε, συγγνώμη, προτίμησαν να ενισχύσουν το μηχανισμό ασφαλείας. Εχθέ το βράδυ στο Λουξεμβούργο, το νέο Τζάι, υπάρχει κατανομή, αν είναι δυνατόν να μιλάμε έτσι για ανθρώπους, την κατανομή των προσφύγων και συνέχεια έχουμε και το εφεδρικό σχέδιο που δείχνει με σαφήνεια πλέον ότι υπάρχουν σοβαρές αντιφάσεις στην πολιτική τη Ευρωπαϊκή Ένωση και ω προ το κόστο. Ε, διότι αντί για σύγκληση και αλληλεγγύη, ουσιαστικά τι κάνουμε, μειοδοτούμε και ενισχύουμε τον ανταγωνισμό ανάμεσα στα κράτη-μέλη για να υποδεχθεί το κάθε κράτο μέλο το μικρότερο δυνατό αριθμό των προσφύγων με το μικρότερο δυνατό κόστο. Αυτό δείχνει ότι δεν είναι καθόλου αξιόπιστα αυτά που λένε ε, από την πλευρά τη νέα κοινοβουλευτική ομάδα Ευρωπαϊκού, ε, τη νέα πολιτική ομάδα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που έχει ο σλόγγαν κυρίως μην έρθετε στην Ευρώπη. Ε, βλέπουμε ε, ότι ε, παρά τις δηλώσεις ανθρωπιστικού χαρακτήρα που κάνουν διάφοροι αρχηγοί κρατών κυβερνήσεων και παρά αυτά που λέει η ΥΠΑΤΗ εκπρόσωπος, αντίθετες αποφάσεις λαμβάνονται σε διάφορες χώρες, στην Ουγγαρία, στη Γαλλία, στο Λουξεμβούργο, στο Ηνωμένο Βασίλειο. Έχουμε διαφορετικούς λόγους και αιτιολόγηση για την χορήγηση ανθρωπιστικής ώρες παραδείγματο χάρη για τους ε, χριστιανούς ε, του Ιράκ. Ε, υπάρχουν ευνοϊκές διατάξεις στη Γαλλία, όμως μην ξεχνάμε ότι υπάρχουν και ανθρωπιστικές θεωρήσεις έγκαινη για σύντομη διαμονή, παραδείγματο χάρη στη Μάλτα, στην Ιταλία, στην Πορτογαλία. Υπάρχουν, υπάρχει ένα συνδυασμό των δύο για την Αστρία, για την Γαλλία, για την Πολωνία, τις κάτω χώρες και άλλες χώρες. Βλέπουμε δεν υπάρχει ομοιομορφία, δεν υπάρχει εναρμόνιση, πολύ διαφορετικά κριτήρια και 16 κρατημέλη χρησιμοποιούν την αρμοδιότητα που έχουν για την έκδοση ανθρωπιστικών θεωρήσεων. Μόνο 16. Για την πίεση, σε σχέση με την πίεση που υπάρχει για τι προξενικέ αποφάσει ε, και την υποδοχή των προσφύγων ε, στο χώρο Σέγγεν, δεν φτάνει αυτό. Δηλαδή θα πρέπει ε, να ξέρουμε ότι σε κάθε προξενείο δεν έχει ο, τον, τις ίδιες δυνατότητες να εκδοθεί μια τέτοια ανθρωπιστική θεώρηση και οι εθνικές ανθρωπιστικές θεωρήσεις δίνει πρόσβαση μόνο σε 10 κράτη-μέλη και όσοι έχουν αυτή την θεώρηση περιορίζονται σε αυτά τα 10 κράτη-μέλη. Δηλαδή αυτό καθιστά αδύνατο, αδύνατη την οικογενειακή επανένωση αν η οικογένεια βρίσκεται σε διαφορετικό κράτος μέλος ε, και ε, είναι σημαντικό πρόσκομα για έναν ετούντα. Θα χρειαστεί ένα σύστημα αυτόματης αναγνώρισης ε, των ανθρωπιστικών θεωρήσεων που εκδίδουν τα κράτη-μέλη. Φυσικά υπάρχουν ενδιασμοί και υπάρχουν διαφορετικές απαιτήσει, παραδείγματο χάρη διαφορετικοί πόροι που διοχετεύονται Τη ανθρωπιστική θεωρήση, ε, και ό,τι καθεξής. Ε, ε, εκεί εντοπίζουμε το ρόλο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ώστε να υπάρχουν κοινοί ρυθμιστικοί κανόνες, κατευθυντήριες γραμμές, τόσο για την έκδοση των ανθρωπιστικών θεωρήσεων, όσο και για τον τρόπο έκδοσής τους, για την προθεσμία, για την απλουστευμένη διαδικασία και αιτιολόγηση, για την απόρριψη της αίτησης ανθρωπιστικής θεωρήσης. Σας ευχαριστώ. Thank you very much. Ευχαριστώ πολύ. Σα ευχαριστούμε κύριε Λιμπέρ. Ο κύριο Γκάρκοφ, εκτελεστικό ευθυντή του Τζουζουλίδα, θα μα μιλήσει για το σύστημα πληροφόρηση θεωρήσεων. Έχετε το λόγο. Thank you, Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, Πρόεδρε, και σας ευχαριστώ και για την ευκαιρία που μου δίνετε να κάνω την παρουσίαση αυτή και να συμμετάσχουμε στη συζήτηση. Έχουμε καλούς ε, λόγους. Το σύστημα αυτό είναι ένα πρακτικό σύστημα για την εφαρμογή της κοινής, πρακτικής, πολιτικής για τις ε, θεωρήσεις και διευκολύνει τις προσπάθειες των κρατών μελών δίνοντας ε, καταρχάς ασφαλείς και αξιόπιστες και γρήγορε ε, μεθόδους ε, ελέγχου της αξιοπιστίας των υπηκών τρίτων χωρών που ζητούν θεωρήσεις και βελτιώνοντας τις εργασίες των προξενικών αρχών μέσω την ανταλλαγή τέτοιων δεδομένων. Και αυτό αποτυπώνεται σε περιορισμένες ευκαιρίες για επιλογή σημείου θεώρησης έτσι θεωρήσεις και επίσης για ε, καλύτερο έλεγχο των, των συνορών. Και όλα αυτά ε, με υψηλά πρότυπα προστασία των δεδομένων και πλήρη συμμόρφωση με τη σχετική νομική βάση. Ω εκ τούτου, αναγνωρίζουμε τη σημασία των συστημάτων αυτών τα τελευταία δύο χρόνια. Έχουμε διεξαγάγει και έχουμε αναλάβει πρωτοβουλίε για διάφορα έργα, προκειμένου το σύστημα να πληρεί τι σημερινέ και τι μελλοντικέ απαιτήσει. Ιδιαίτερα για τα συστήματα πληροφόρηση θεωρήσεων, θα πρέπει να αναφέρω ότι για την περίοδο αυτή οι ικανότητε έχουν τετραπλασιαστεί του συστήματο σε σχέση με το 2011, όταν τέθηκε σχέση το σύστημα. Ένα σημαντικό ε, παράγοντα είναι το βιομετρικό σύστημα που παρέχει σημαντικέ ε, πληροφορίε και σημαντικά εργαλεία για τι προξενικέ αρχέ όταν γίνεται επεξεργασία των αιτήσεων. Ε, εξαπλή αύξηση των ικανοτήτων εδώ. Με όλα αυτά λοιπόν που έχουν επιτευχθεί, πρέπει να πω ότι σήμερα το σύστημα πληροφόρηση θεωρήσεων μαζί με το βιομετρικό σύστημα είναι απόλυτα σε θέση να ανταπεξέλθουν στι ανάγκε των κρατών μελών που προκύπτουν από τον συνεχιζόμενο ρόλο των συστημάτων ε, πληροφόρηση για θέματα θεωρήσεων σε παγκόσμιο προσκήνιο. Εκ το σύστημα είναι σε θέση να ανταπεξέλθει, να ανάγκε στις ανάγκες του συστήματος πληροφόρησης θεωρήσεων μέχρι το τέλη της ε, διαδικασίας αυτές. Θα δούμε την επόμενη εβδομάδα μια πρώτη έκθεση όπου και προγραμματίζουμε μια έκθεση για την Ουκρανία. Να σας πω ότι αναμένονται πολύ ομαλές διαδικασίες από την υπηρεσία όπως έχει γίνει ως τώρα η μετάβαση και το ίδιο προβλέπουμε και για όλες τις υπόλοιπες περιφέρειες μέχρι τα τέλη του έτους που θα γίνει η μετάβαση για την τελευταία χώρα τα τέλη Νοεμβρίου συγκεκριμένα, ακούγοντα τι παρεμβάσει των προηγούμενων ομιλητών, καθίσταται εκ παραλίλου σαφέ ότι είναι μεγάλη, μεγάλες οι πολλέ εικόνες που ακούγονται για τη διευκόλυνση των θεωρήσεων και πολλέ είναι οι εμπειρίε υπηκών τρίτων χωρών που ζητούν θεωρήσει ε, με άσχημε εμπειρίε. Αυτή η διευκόλυνση λοιπόν μπορεί να γίνει με ευφυή χρήση τη τεχνολογία που δίδεται στην VAS και σε άλλε τεχνολογικές μορφές. Και υπό την έννοια αυτή είμαστε έτοιμοι να υποστηρίξουμε τις προσπάθειες αυτές και να δώσουμε τα απαραίτητα εργαλεία για την πρακτική εφαρμογή των νέων στοιχείων που προβάλλονται στον κώδικα για τις θεωρήσεις. Σύντομα, ελπίζουμε. Ευχαριστούμε πολύ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, λέει η Πρόεδρος. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και για την σύντομη αυτή παρουσίασή σα. Τέλο. Στέφαν Κούρτεμπεκ. Πώς θα μας παρουσιάσετε την πλευρά των αρχών στα κάτι που ευθύνονται για την ασφάλεια. Έχετε το λόγο. Καλησπέρα, είμαι ο Στέφαν Χερτμπέκα, υπεύθυνο για τη μονάδα ελέγχου των συνόρων στο αεροδρόμιο των Βρυξελών, National. Αυτό που θα σας πω είναι η άποψή μου. Είμαι κάποιος που πρέπει να εφαρμόζει το σύστημα αυτό. Το σύστημα VIS, το VIS. Σύμφωνα με τους κανόνες σας και το νομικό σας σύστημα. Θα δώσω μια απάντηση στις βασικές ερωτήσεις που αναφερόταν στην πρόσκληση που έλαβα. Η πρώτη ερώτηση είναι τι προβλήματα βλέπετε με τον κώδικα για τις θεωρήσεις που εφαρμόζεται. Καταρχάς, το σύστημα VIS, το ριζοσφιστικό αυτό σύστημα που εφαρμόστηκε είναι πάρα πολύ καλό. Βλέπουμε στα σύνορα λοιπόν ότι οι απάτες όσον αφορά τις θεωρήσεις έχουν σχεδόν μηδενιστεί στο αεροδρόμιο των Βρυξελών. Σημαίνει λοιπόν ότι ένα από τα βασικά θέματα της ασφαλείας, δηλαδή διαπιστώνει κανείς αν ένα έγγραφο μία θεώρηση είναι αυθεντικά και εντάξει, έχει διευκολυνθεί πάρα πολύ σαν έργο. Ριζοσπαστική αλλαγή. Αυτό που είναι το όφελο του συστήματο είναι ότι για να πάρουμε τα δαχτυλικά αποτυπώματα πρέπει να χρειαστούμε χρόνο. Έχουμε ουρέ λοιπόν στο αεροδρόμιο. Και αν το σύστημα επεκταθεί πρέπει να έχει κανεί υπόψη του ότι από τώρα μέχρι το 2035, μετά από μία εικοσαετία, μπορεί να έχουμε το διπλάσιο αριθμό επιβατών που διέρχονται από τα αεροδρόμια. Οπότε αν συνεχιστεί το σύστημα θα πρέπει να έχετε υπόψη, θα χρειαστεί ριζοσπαστικές αλλαγές όσον αφορά το προσωπικό. Και κάτι άλλο που είδαμε στο αεροδρόμιο. Έχουμε έναν χώρο Σέγγεν, αλλά δεν είναι όλοι οι κανόνες ίδιοι για τις διάφορες χώρες. Είναι δυνατόν κάποιος που έρχεται από τρίτη χώρα να χρειάζεται θεώρηση για μία χώρα και όχι για άλλη. Αυτό μπορεί να οδηγήσει στην περίπτωση όπου, παραδείγματος χάρη, ένα αεροσκάφος κατευθύνεται προς το αεροδρόμιο Α και κάποιος πληρεί όλες τις προϋποθέσεις, δεν χρειάζεται θεώρηση Σέγγεν σε αυτή τη χώρα και τελικά το αεροδρό... προσγειωθεί σε άλλο αεροδρόμιο, το αεροπλάνο αναγκαστεί να πάει, ίσως να του αρνηθούν την είσοδο, διότι σε αυτό το αεροδρόμιο το άλλο που πήγε το αεροπλάνο χρειάζεται θεώρηση. Προτείνουμε λοιπόν να υπάρχει πλήρης ριζοσπαστική ανανέωση του κώδικα θεωρήσεων σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του ευρωπαϊκού αυτού χώρου, του ενίου χώρου. Λοιπόν, αν έχουμε ένα καλό έγγραφο, παρόλα αυτά υπάρχουν προϋποθέσεις για την είσοδο που πρέπει να ελεγχθούν και ένας από τους όρους είναι ή η ε, ανανέωση της διαμονής στο χώρο Σέγγεν. Πρέπει να εξετάσουμε το διαβατήριο, να δούμε εισόδους, εξόδους. Είναι χρονοβόρα διαδικασία. Και επανέρχομαι στο αρχικό μου σχόλιο ότι αν είναι πιο μακροχρόνια η διάρκεια της ισχύω της θεωρήσεως, αν τώρα μένει κανείς 90 μέρες σε μια περίοδο 180 ημερών και έχει 20 σφραγίδες στο ε, διαβατήριο να βρει κανεί όλε όλες τις σφραγίδες και να υπολογίσει άλλο ένα εντάξει αυτό χρειάζεται χρόνο ε, και άρα σημαίνει ουρέ στο αεροδρόμιο άρα δημιουργούνται και οικονομικά προβλήματα και κάτι άλλο είναι ο έλεγχος των λόγων του ταξιδίου για το αεροδρόμιο των Βρυξελών έχουμε πολύ ψηλό ποσοστό αρνήσεων, απορρίψεων λόγω του λανθασμένου αιτίου, της λανθασμένης αιτιολόγησης του ταξιδίου. Δεν είναι σωστή πολιτική να κρίνεται μια θεώρηση που επιτρέπει το ταξίδι και κάποιος να πρέπει να σταματά στα σύνορα διότι βλέπουμε ότι οι λόγοι του ταξιδιού δεν είναι αυτοί που αναφέρονται, δεν είναι σωστοί. Δεν είναι καλό για τον ταξιδιώτη, έχασε πολύ χρόνο, χρήματα, δεν είναι καλό για τις επιχειρήσεις, οι αεροπορικές εταιρείες πρέπει να επιστρέψουν τον επιβάτη με το δικό τους κόστος, είναι κακό για τον τουρισμό, αυτά είναι αρνητικά στοιχεία. Τώρα, αυτό που βλέπουμε είναι ότι υπάρχουν διαφορές μεταξύ αρκετών χωρών. Στο δούμε των Βρυξελών όλους εκείνους που απορρίπτουμε την είσοδό του δεν επιτρέπουμε την είσοδό του στα σύνορα, η, μπορεί να φτάσει μέχρι 60% η απόρριψη, η άρνηση εισόδου, διότι παρουσιάζουν λάθος λόγο ταξιδίου. Γιατί γίνεται αυτό, από επαφέ που έχουμε συναδέλφου σε άλλε χώρε, τι παρατηρούμε, παρατηρούμε ότι αυτό που βλέπουμε στι Βρυξέλλε ισχύει. Χρησιμοποιούν καμιά φορά άλλη μέθοδο από εμά, οι άλλοι συνάδελφοι. Το Βέλγιο είναι μικρή χώρα. Οι περισσότεροι μεθοριοφύλακες είναι πολύγλωσσοι, μιλάνε τρεις, τέσσερις, πέντε γλώσσες. Άρα είναι πολύ ευκολότερο να ρωτήσουν πολλές ερωτήσεις πολλούς επιβάτες και αυτό δεν ισχύει πάντα σε άλλες χώρες. Ίσως και αυτός είναι ένας λόγος που έχουμε τόσες πολλές αρνήσεις εισόδου εμείς. Τώρα αν θέλουμε ένα ενιαίο σύστημα στην Ευρώπη θα πρέπει να βρούμε μία λύση σε αυτό το πρόβλημα. Ανταλλαγή πληροφοριών. Τι παρατηρούμε, ότι εντός του συστήματος VIS, αν υπάρχει κάποιος στον έλεγχο της, τον πρωτοβάθμιο, βλέπουμε ότι οι πληροφορίες που έχουμε στο σύστημα περιορίζονται σε αυτά που είναι τυπωμένο στο έγγραφο VIS, στη θεώρηση. Σε πολλές περιπτώσεις υπάρχουν και συμπροματικές πληροφορίες και έτσι έρχομαι στο λόγο πραγματοποίησης των ταξιδίων. Αυτές οι συμπροματικές πληροφορίες που έπρεπε να υπάρχουν στις περισσότερες περιπτώσεις απουσιάζουν. Και αυτό ίσως εάν καλυφθεί μπορεί να λύσει το πρόβλημα που σας ε, εξέθεσα. Τώρα η αλλαγή του συστήματος των θεωρήσεων. Και τι αντίκτυπο έχει αυτό στις υπηρεσίες ελέγχου και στην ασφάλεια. Όσο το σύστημα αυτό καθεαυτό είναι συνεκτικό, εναρμονισμένο και καλό, δεν επηρεάζει τους μεθοριακούς ελέγχους. Ποιες είναι οι απόψεις σας όσον αφορά τι προτάσει για τη διαχείριση τη ηγητρία, Όσον αφορά πρώτα απ' όλα τα δικαιολογητικά, θεωρούμε ότι δεν θα είναι αναγκαίο να παρουσιάσετε ένα έγγραφο που αφορά τη στέγαση, τη διαμονή. Κάποιο που παρουσιάζεται σε ένα αεροδρόμιο σήμερα, με κρατήσει σε ξενοδοχείο, ίσως να έκανε την κράτηση όταν κατέβηκε από το αεροπλάνο και μετά από 10 μέτρα αφού περάσει τον έλεγχο να ακυρώσει την κράτηση η ακύρωση αυτή δεν αλλάζει πολύ ε, το θέμα της ασφαλείας ε, σχετικά με το μεθοριακό έλεγχο. Μετά, η έφεση κατά της άρνησης χορηγήσεως θεωρήσεως. Δεν μπορώ να πω τίποτα. Γι' αυτό, για τα όσα γίνονται σε ένα προξενείο, για τη χορήγηση της θεώρησης. Αν ήταν δυνατόν όμως να υπάρχει έφεσης, να γίνει έφεση προσφυγή κατά αποφάσεως που λαμβάνεται στα σύνορα, εκεί πρέπει να σκεφτούν προσεκτικά πώς θα μπορεί να γίνει αυτό. Ίσως να έχει μεγάλο αντίκτυπο αυτό, ε, ριζοσπαστικό κίνδυνο όσον αφορά τη λειτουργία του μεθοριακού ελέγχου. όσον αφορά την ασφάλεια και τους μεταναστευτικούς κινδύνους. Η επαλήθευση των όρων για την διέξοδο των κατόχων τουριστικής βίζας ίσως να καθυστερεί ε, την είσοδο διότι χρειάζονται πολλές φραγίδες και έλεγχος φραγίδων. Η πρόκληση όμως είναι η διέλευση των εσωτερικών συνόρων όπως καταλαβαίνω. Μπορεί να ζητήσει κάποιο. Μια θεώρηση. Για το Βέλγιο Φερρυπίνη, για τη Γαλλία. Πρέπει να καταλάβουμε όμως ότι κάποιο που δεν χρειάζεται θεώρηση για την χώρα Α Από τη στιγμή που θα μπει στο χώρο Σέγγεν, δεν ξέρει που, θα που θα πάει αυτό. Δεν έχει εσωτερικά σύνορα πλέον να τον ελέγξουν. Άρα είναι καλή σκέψη, στην πραγματικότητα είναι πολύ δύσκολο να ελέγξουμε. Η αύξηση της διάρκειας ισχύω των θεωρήσεων ίσως να οδηγήσει σε περισσότερες καταχρήσεις. Όσο πιο μεγάλη διάρκεια της θεώρησης, τόσο πιο ενδιαφέρον για κάποιον είναι να ταξιδέψει στην Ευρώπη χρησιμοποιώντας τη θεώρηση αυτή. Και τελευταίο σημείο, για το πεδίο, αν θα πρέπει να περιοριστεί ή να επεκταθεί, όσον αφορά τα προαναφερθέντα, ένα σχόλιο έχω. Η ασφάλεια δεν περιερίζεται στο ΒΙΣ ή στο ΣΥΣ, αλλά πολλά άλλα στοιχεία θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη πριν να λαμβάνετε μια απόφαση στα σύνορα. Και σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Πολύ σας ευχαριστούμε κύριε Γκούρντεμπέκια. Ευχαριστώ όλους τους συναδέλφους. Πολύ ενδιαφέρουσες ε, οι απόψεις και παρατηρήσεις. Τώρα θα ήθελα να κάνουμε ένα γύρο ερωταπαντήσεων. Και μετά θα ακούσουμε και την εκπρόσωπο τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τη ε, Λετωνική προεδρία. Προεδρίας. Ο κύριος Μπάκερ, ε, γιατί είναι και σκιώδη εισηγητή από πλευρά ε, του ΕΛΚ. Σας ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε, ευχαριστώ όλου όσοι συμμετέχουν σε αυτή την πολύ σημαντική ακρόαση. Είναι ένα θέμα καθοριστικό για την ποιότητα αυτό που συζητάμε. Θα ήθελα Εν συντομία να πω ένα ευχαριστώ προς την κυρία εισηγήτρια. Η κυρία Φαγιών ανέλαβε πρόσφατα τον φάκελο αυτό και βλέπω πραγματικά ότι έχει κάνει ήδη ένα έργο αξιοσημείωτο. Θα ήθελα να συγχαρώ και την κυρία Περίσου για την απόδοση της οργάνωσης του. Είναι πάρα πολύ επαγγελματική η αντιμετώπιση με έναν πολύ ανθρώπινο τρόπο και με διευκρινήσεις που ε, είναι πραγματικά σημαντικές γιατί στην οργάνωση δεν λαμβάνονται αποφάσεις, μόνο στις προξενικές αρχές λαμβάνονται οι αποφάσεις σχετικά με τις διευκολύνσεις. Να κάνω μια ερώτηση προς τον κύριο Ντεγέγκερ. με κύριε Πρόξενε, θα ήθελα καταρχάς να σας ευχαριστήσω για το γεγονός ότι κυρίως εστιαστήκατε στον τομέα της ε, ασφάλειας. Να εκφράσω και τις τεράστιες αμφιβολίες που έχω όμως σε ό,τι αφορά το θέμα των ανθρωπιστικών θεωρήσεων. Δεν έχουν καμία θέση εδώ. Ασφαλώς υπάρχουν καταρχάς ε, οι θεωρήσεις ε, για εμπορικούς σκοπούς, για ε, επιχειρηματικά ταξίδια και νομίζω ότι θα πρέπει από την άλλη να είναι αυτονόητο ότι το ανθρωπιστικό ζήτημα είναι κάτι το οποίο με τόλμη θα πρέπει να προασπίσει. Όχι όμως εδώ, σε αυτό το φάκελο. Σας παρακαλώ να το διευκρινίσουμε αυτό. Δεν κατανοώ γιατί τα μπλέκουμε. Να ρωτήσω όμως ε, έναν άνθρωπο με τόσο μεγάλη εμπειρία. Ποια είναι η εμπειρία σα στι θεωρήσει πολλαπλή εισόδου με ανθρωπιστικές ε, θεωρήσεις και επίσης στον τομέα του βασίλου. Δεύτερη ερώτηση προς τον κύριο Κουτεμπέκα. Να τον ευχαριστήσω που τόσο γρήγορα, με τόσο σύντομη ειδοποίηση ήλθε εδώ στην ακρόαση. Μα βοηθάει πολύ το, ότι είσαστε εδώ. Γιατί σε τελική ανάλυση είσαστε οι υπάλληλοι οι οποίοι θα αντιμετωπίσετε αυτά τα οποία αποφασίζουμε. Μια συγκεκριμένη ερώτηση λοιπόν. Μια και είσαστε και ασχοληθείτε στην πράξη με τα θέματα αυτά, υπάρχει μια νέα μορφή για τις θεωρήσεις, το άρθρο 33, μία θεώρηση για το πρόθεσμο τουρισμό. Διαρκεί μόνο 15 ημέρες και μάλιστα ισχύει μόνο στο κράτος μέλος έκδοσης. Αλλά ούτε στο προξενείο, ούτε σε κάποια εξωτερική υπηρεσία ισχύει. Μόνο στα σύνορα. Πώς λοιπόν εσείς προσωπικά αξιολογείτε πρακτικά την πρόταση αυτή. Γιατί ο συνοριοφύλακας καλείται μέσα σε δευτερόλεπτα να αποφασίσει και να αποφανθεί για θέματα ασφαλείας και μάλιστα θέματα τα οποία ένα προξενείο χρειάζεται μέρες, μήπως εβδομάδε εβδομάδες σε κάποιες περιπτώσει για να, αποφασίσει. Πείτε μα λοιπόν, κάντε μια εκτίμηση. Εγώ νομίζω ότι δεν είναι δυνατόν να υπάρχει α, τέτοια συνοριακή εκπαιδεύση χωρίς προβλήματα με τέτοια πρόβλεψη. Θα ήθελα να ακούσω όπως και την δική σας άποψη. Πρόεδρος, ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Ντεπρέης. Έχει το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Συγχαρητήρια ε, και ευχαριστίες σε όλους τους εμπειρογνώμονες. Ε, ε, κυρίως ε, για τις ε, συγκεκριμένες και ριζοσπαστικές προτάσεις που κάνουν τις έχω σημειώσει και θα επανέλθω. Θέλω να κάνω μια ερώτηση στον κύριο Ντεγιάγκερ. Μας είπε ότι πρέπει να προσέξουμε για τις παράπλευρες επιπτώσεις το είπατε λίγο απλοϊκά. Μας είπατε ότι ο αυτόματος ε, μηχανισμός αυτός ε, για τις θεωρήσεις ελεύθερης μετακίνησης ε, δεν είναι καλός. Πολύ ριζοσπαστικό μου ακούγεται αυτό. Θα μπορούσατε να το εξηγήσετε. Για την ανθρωπιστική θεώρηση εγώ είμαι υπέρ. Και το έχουμε συζητήσει και παρουσία των εκπροσώπων τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή και μα είχαν πει ότι αυτό δεν αντάσσεται στον κώδικα των θεωρήσεων και δεν θα έπρεπε εκεί να προβλέψουμε την ανθρωπιστική θεώρηση. Όχι δηλαδή στα πλαίσια ε, της ε, τωρινής ε, συζήτησής μας. Και αυτό ριζοσπαστικό μου ακούγεται. Θα μπορούσατε επίσης να επιχειρηματολογήσετε, δηλαδή κύριε Γκυμπέρ, γιατί εσείς επιμένετε για το αντίθετο, διότι παρά το ριζοσπαστικό του πράγματος εγώ δεν έχω πιστεί. Ο κύριος Γκουρντεμπέκε μας είπε ότι έχει εκδοθεί εντελώς νόμιμα μια θεώρηση Φτάνει κάποιο ε, στο Ζάμεντεμ, αλλά δεν τον αφήνουν να μπει στην επικράτεια του Βελγίου. Άλλο πάλι αυτό ριζοσπαστικό. Βλέπουμε λοιπόν ότι ε, για απορρίπτεται το 60% των θεωρήσεων λόγω ε, ε, πλημελούς αιτίας μετακίνησης. Μπορείτε να μας πείτε περισσότερα πράγματα για να καταλάβουμε ε, την εμβέλεια αυτής της παρατήρησης που κάνετε και σας κατάλαβα καλά, είναι μέσα στο σύστημα VIES ε, αυτές οι αιτίες. Δηλαδή, πώς είναι δυνατόν να μειώσουμε το χάσμα που υπάρχει ανάμεσα στην έκδοση θεώρησης ε, και την ε, ε, έγκριση της εισόδου στη χώρα. Γιατί υπάρχει μια πάρα πολύ μεγάλη διαφορά. Σας ευχαριστούμε κύριος Πάνη. Σας ευχαριστώ για την δημόσια ακρόαση αυτή. Σας ευχαριστώ για όλες τις παρουσιάσεις που κάνατε. Θα ήθελα να αρχίσω με το εξής ερώτημα για τον κύριο Ντεχάγκερ. Προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, να λειτουργούν αυτόματα τα σύστηματα για τους τακτικούς και καταχωρημένους ταξιδιώτες, ε, τους registered travelers. Αν δεν υπάρχει πρόβλημα, εσείς θεωρείτε ε, σκόπιμο να ε, καλούνται ε, για συνέντευξη αυτή η καταχωρημένη ταξιότητα... αν υπάρχει διάταξη για προσωπική παράσταση. Δεύτερη ερώτηση προς τον κύριο Κάρκοφ. Μπορείτε να μας ενημερώσετε για το ρολάουτ του συστήματος με περισσότερες λεπτομέρειες. Όταν θα ολοκληρωθεί αυτή η ομολογουμένως ριζοσπαστική διαδικασία, ε, με απασχολεί ένα γενικότερο ερώτημα, διότι μιλάμε για την αναθεώρηση του κώδικα Σέγγεν στο Συμβούλιο και προτείνει η Προεδρία ένα νέο άρθρο για τα τέλη για τις θεωρήσεις. Ε, δεν υπήρχε όμως αυτό στην αρχική πρόταση, άλλο ένα ριζοσπαστικό στοιχείο. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή λοιπόν ε, προτείνει ε, να χρησιμοποιηθεί διαδικασία επιτροπολογίας για το VIS, καλύπτοντας και το διοικητικό κόστος. Τι πιστεύετε εσείς για μια τέτοια πρόταση. Θεωρείτε ότι είναι προ συμφέρον των ετούντων ε, θεώρηση ή μήπως ε, θα αποτελέσει ε, πρόσκομα για την Ευρωπαϊκή Ένωση και θα μειώσει την ελκυστικότητά τους ως τουριστικός ή επαγγελματικός προσανατολισμός. Σας ευχαριστούμε και τώρα η κυρία Στίβενς παρακαλώ έχετε το λόγο. Thank you. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ συνάδελφοι. Κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να πω δύο λόγια για τις ανθρωπιστικές θεωρήσεις από την νομική πλευρά. Βέβαια είμαι νομικός και προφανώς από αυτή την πλευρά θα μιλήσω. Δεν υπάρχει τέτοια δυνατότητα χορήγηση θεωρήσεων υπό τον παρόντα κώδικα ε, θεωρήσεων και είμαι πεπισμένη ότι πρόκειται για περιπτώσεις θεωρήσεων για 90 μέρες maximum που δεν ε, είναι το ίδιο με τους εθνικές άσυλο ε, που ζητούν να μείνουν παραπάνω. Αυτό λοιπόν μπορεί να αλλάξει, αλλά γιατί να χρησιμοποιήσουμε τη βίζα του Σέγγεν που ε, προορίζεται για επιχειρηματικούς σκόπους, για σκοπούς ανθρωπιστικούς. Θα συμφωνήσει μαζί μου και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή φαντάζομαι. Επίση, από πολυπλευρά πολιτική, πολιτική, αυτό θα σημαίνει ότι θα ανοίξουμε τα σύνορα χωρί προηγούμενο και στην παρούσα φάση αυτό αποτελεί εθνική αρμοδιότητα. Άρα θα μπορούσε να καταστεί ένα τυπικό δικαίωμα. Αυτό θα σημαίνει ότι τα ευρωπαϊκά δικαστήρια θα ξεκινούσαν να ερμηνεύουν την νομοθεσία και να υπαγορεύουν ουσιαστικά στα κράτη υπό οποίου όρου θα επιτρέπουν στον κόσμο να υπησέρχεται στην ε, επικρατεία του. Βλέπουμε μια παρόμοια τάση στο Δουβλίνο όπου μπορεί να αναγκαστούν να επιστρέψουν σε κάποιες χώρες ε, ε όταν συντρέχουν κάποιες συγκεκριμένη όροι. Σκεφτείτε το λοιπόν, αν εκδώσουμε μία θεώρηση και να την δώσουμε σε οποιοδήποτε ισχυρίζεται ότι έχει περιέλθει σε δινή κατάσταση, πραγματικά εύχομαι οι συνάδελφοί μου να διαβάζουν τον κώδικα για τις θεωρήσεις και τον κώδικα για το Σέγγεν και θα εξηγήσω και πιο πολλά στοιχεία αν το επιθυμείτε. Μόλις ε, γύρισα από επίσκεψη στα σύνορα της Συρίας, ε, επισκέφτηκα το ε, κατάλημα προσφύγων στην Ιορδανία, στο Τάρι, και δεν έχω καμία αμφιβολία ότι όλοι αύριο μεθαύριο θα στριμώχνονται και θα ζητάνε θεωρήσει. Νομίζω ότι και εμείς όλοι το ίδιο θα κάναμε στην θέση του. Έχω λοιπόν κάποια συγκεκριμένα ερωτήματα να θέσω για το ποιο θα είναι ο αντίκτυπο στην ασφάλεια για τα μεμονωμένα κράτη-μέλη. Οι όροι για την αίτηση θεωρήσεων ήταν πιο, λιγότερο αυστηροί σε κάποια από σε κάποιε περιπτώσει σήμερα. Επίσης, Πώς θα περιοριζόταν αυτό το δικαίωμα θεωρήσεων οι 90 μέρες ενώ ισχύει το 80 μέρες έως τώρα και πώς θα εφαρμοζόταν αυτό στην πράξη. Και ανησυχώ πραγματικά σε ό,τι αφορά την επέκταση του κώδικα θεωρήσεων και στις ανθρωπιστικές θεωρήσεις. Νομίζω ότι αυτό θα αύξανε, αύξανε σημαντικά το φόρτο εργασία των προξενείων και έτσι και την γραφειοκρατία και θα αύξανε και την διάρκεια χορηγήση θεωρήσεων και σε τι βαθμό θα υπονόμευε αυτή η επέκταση στους ήδη υφιστάμενους νόμους για το άσυλο και το CIS και σε ό,τι αφορά την ικανότητα των κρατών μελών να υποδεχτούν μετανάστες και να ταξιδέψουν σε άλλα κράτη-μέλη. Κάτι το οποίο βλέπουμε ότι απελείται ήδη το είδαμε αυτή την εβδομάδα. Ε, κύριε Πρόξενε, λοιπόν, αυτό θα σημαίνει περαιτέρω επιβάρυνση για τις προξενικές αρχές. Πώς πιστεύετε, λοιπόν, ότι οι ανθρωπιστικές αρχές θα μπορούσαν ενδεχομένω να διεπεραιώνονται. Σας παρακαλώ, σκεφτείτε το και ξανασκεφτείτε το θέμα αυτό. Ευχαριστώ πολύ, λέει η Πρόεδρος. Δεν έχουμε άλλες ερωτήσεις και τώρα να δώσουμε τις απαντήσεις. Euh, μου έθεσαν πολλές ερωτήσεις, προνόμιο μου να απαντήσω. Λοιπόν, καταρχάς όσον αφορά τις ανθρωπιστικές ε, θεωρήσεις, προσωπικά νομικός πώς έχω την εντύπωση ότι η ανθρωπιστική θεώρηση δεν υπησέρχεται καθόλου στο πλαίσιο του κώδικα των θεωρήσεων. Ο κώδικας αυτός αφορά τις θεωρήσεις βραχίας διαρκείας, 90 ημέρες κατά περίοδο 180 ημερών και μακροπρόθεσμα πριν την εκπνοή αυτής, μία αναχώρηση του ατόμου που απέκτησε τη θεώρηση. Είναι ξεκάθαρο, αυτά είναι τα προνόμια που διαθέτει. Αν θέλουμε να εισάγουμε ε, μία θεώρηση για μία διαμονή ε, μακρύτερη που θα χορηγείται σε ένα άτομο που θα έπρεπε να παραμείνει πολύ πιο πολύ στο χώρο Σέγγεν, τη αυτή η περίπτωση δεν βρισκόμαστε πλέον στη βραχία διάρκεια του κώδικα των θεωρήσεων, αλλά στη μακρά διάρκεια διαμονής. Και είναι το εθνικό δίκαιο που εφαρμόζει αφορά το προνόμιο αυτό. Νομίζω λοιπόν ότι δεν πρέπει να αναμειγνύουμε τα πράγματα. Δεν έχω τίποτα κατά τη ανθρωπιστική θεωρήσεω, αλλά δεν θα πρέπει εκεί να καλυφθεί. Αυτή είναι προσωπική άποψη. Τώρα, οι συνέπειε για τα προξενία, φαντάζομαι ότι ένα προξενείο στην Τουρκία. Υπάρχει ένα προξενείο Σέγγεν στην Τουρκία. Από τη στιγμή λοιπόν όπου υπάρχουν οι πληροφορίες σύμφωνα με τις οποίες το προξενείο Σέγγεν χωρίς δικαιολογητικά, χωρίς διαβατήριο προφανώς, χωρίς τίποτα, χορηγεί θεώρηση και δίνει το προνόμιο να εγκατασταθεί κανείς στο χώρο Σέγγεν, διότι αυτό είναι ο στόχος, αποκτώντας το άσυλο, φαντάζομαι τον αριθμό των ατόμων που θα κατέφθανε και θα προσπαθούσε να έρθει στο προξενείο προφανώς δεν θα είχαμε τη δυνατότητα υποδοχής. Και εκεί φαντάζομαι επίσης ε, τι κίνηση θα μπορούσε να δημιουργηθεί και τι προβλήματα. Ε, αν έχετε εκατοντάδες χιλιάδες αιτήσει, εν τη αυτή περιπτώση, ε, χρειάζονται χιλιάδες έλεγχοι. Διότι ανάμεσα στα άτομα που ζητούν αυτό το προνόμιο, αυτή τη θεώρηση, οπότε έμεσα ή άμεσα εξάλλου το άσυλο, έχετε ίσως εκείνους οι οποίοι έχουν υπησέλθει για άλλους λόγους λιγότερο ε, αξιόπιστους και σεβαστούς. Τι θα κάνουμε εκεί. Πώς μπορεί ένα προξενείο να εξετάσει τόσα αιτήματα και υποθέτω σε πολύ βραχή χρονικό διάστημα. Νομίζω ότι γρήγορα θα αντιμετωπίσουμε ένα φαινόμενο, αυτό που βλέπουμε σε κάποιους ε, ισπανικούς ε, στο Μαρόκο, Φερρυπίν. Φαντάζομαι λίγο πολύ αυτή την κατάσταση. Μπορεί να ασφάλω, κατά την άποψή μου όμως, αν θέλουμε να εισαγάγουμε αυτού του είδου τη θεώρηση, θα πρέπει να γίνει μελέτη αντικτύπου ε, που θα πρέπει να γίνει με κάθε σοβαρότητα. Αυτό για την ανθρωπιστική βίζα. Ε, αναφέρθηκα επίσης ε, στις αντίστροφες, ε, αντίθετες συνέπειες που θα είχε η δωρεάν χορήγηση αυτή η δωρεάν χορήγηση συνδέεται με κάποια αίτια χορηγήσεως του προνομίου αυτού της θεωρήσεω. Κάποιο που ζητά μια θεώρηση για να παραστεί σε ένα σεμινάριο που διοργανώνεται από μια ΜΚΟ θα, ε, θα διεκδικήσει τη δωρεάν χορήγηση. Αν αυτό το άτομο ή το προξενείο μπορούσε να του δώσει μια θεώρηση πολλαπλών εισόδων για μια διάρκεια μακράς χρήσεως ότι αυτή η περιπτώση μπορεί να του δώσει δωρεάν αυτή τη θεώρηση ή όχι. Ε, βλέπετε ότι δημιουργούνται προβλήματα. Πολύ συχνά στο Αλγέρι αντιμετώπισα αυτό το πρόβλημα. Έλεγα στον κόσμο ε, μπορείτε να έχετε τη δωρεάν χορήγηση. Αλλά αν σας δώσω δωρεάν ε, τη θεώρηση είναι για συγκεκριμένο σκοπό. Είναι μια είσοδος για τόσες μέρες, χι οι μισές θεωρήσεις στο Αλγέρι που χορηγούνται ήταν θεωρήσεις πολλαπλών εισόδων διαρκείας ισχύω τουλάχιστον ενός έτους, είναι σαφές ότι το άτομο προτιμούσε να πληρώσει για το προνόμιο αυτό. Πρέπει λοιπόν να προσέξουμε όταν εισάγουμε τον χαρακτήρα αυτή τη δωρεάν χορηγήσεω για κάποια αίτια, διότι επίση εισάγεται και άλλο περιορισμό, δηλαδή χορηγήσεω τη βίζα για συγκεκριμένο σκοπό. Ε, τρίτη ερώτηση όσον αφορά τον αυτόματο χαρακτήρα ε, των θεωρήσεων πολλαπλών εισόδων. Στο Αλγέρι εμείς ε, πολύ εύκολα χορηγούσαμε θεωρήσεις πολλαπλών εισόδων για πολλαπλούς λόγους. Φανταστείτε λοιπόν ότι κάποιος Αλγερινός που καταφθάνει στη Γαλλία έρχεται μία φορά για θέματα επαγγελματικά, μετά με την οικογένειά του για τουρισμό, εν συνεχεία για να πάει να επισκεφτεί ξάδερφο, ξαδέλφη ε, γαμπρό κλπ. Οπότε ε, υπάρχουν πολλοί λόγοι. Μπορεί να έρθει επίση για να πάει στο νοσοκομείο και να λησμονήσει να πληρώσει το λογαριασμό. Εγώ είχα ένα ντουλάπι ολόκαιρο στο προξενείο μου στο Αργέρι γεμάτο και κρατούσα τους απλήρωτου λογαριασμούς. 17 εκατομμύρια ευρώ ήταν οι απλήρωτοι λογαριασμοί ε, και ήταν απλώς η κορυφή του παγόβουνου. Εγώ θέλω να υπάρχει ένας αυτοματισμός, αλλά θα πρέπει να υπάρχει και ένας εκ των προτέρων έλεγχος. Ε, υπάρχουν χρέη, ο άνθρωπος αυτό σεβάστηκε κάποιους κανόνες. Εγώ θα υποστήριζα περισσότερο μια συνετή προσέγγιση. Αυτοματισμός στην πράξη, θεωρητικά μάλλον, αλλά στην πράξη ελέγχουμε και κάνουμε εξακριβούς. Αυτά. Ε, ε, ε, ε, ευχαριστώ. Ο κύριος Κούρτεμπέκε. Ακούω κάποια πράγματα και αναρωτιέμαι τι στο καλό κάνω εδώ. Συγγνώμη, αλλά για τις ανθρωπιστικές ε, θεωρίε ισχύουν άλλα πράγματα. Ε, εσείς μου μιλάτε για τις τουριστικές βίζες. Συγγνώμη, αλλά το αντικείμενο ήταν οι ανθρωπιστικές θεωρίες και προσπάθησα να σας πω γιατί πιστεύω εγώ όταν είναι τόσο καταστροφική η κατάσταση όπως αυτή που βλέπουμε στα σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης μπορείτε να μιλάτε υπάρχουν κίνδυνοι, επισύρουν κινδύνους ε, και μπορεί να είναι πλαστά τα έγγραφα. Εγώ σας λέω ότι από τις αρχές του 2015 έχουν πεθάνει 2.000 και έχουμε 100.000 από την Συρία από τη Λιβύη, από τη Σομαλία και έρχονται ε, ε, στο ισχυρότερο ε, οικονομικό κέντρο την Ευρωπαϊκή Ένωση με τα 500 εκατομμύρια και τι θα κάνετε με την περίπτωσή μου, τι προνόμια μπορείτε να μου δώσετε. Βλέπουμε λοιπόν ότι δεν ισχύουν οι ίδιες διατάξεις με αυτές του κώδικα ούτε και με του μελλοντικού κώδικα το θέμα είναι τι θα κάνετε με αυτούς που θέλουν να ε, ε, έχουν των ίδιων προνομίων. Ε, πιστεύω ότι ε, πέρα από τους λόγους ασφαλείας, πέρα από τα οικονομικά ζητήματα, τα νομικά ζητήματα και τα, ε, τα δικαιώματα, γιατί τα δικαιώματα συνδέονται με τους ανθρώπους, υπάρχουν και αναπόφευκτες καταστάσεις και υπάρχουν τρόπους να χειριστεί κανείς στις προβληματικές καταστάσεις. Μπορεί κάποιος να πει όχι, τίθενται αυτά τα ζητήματα, τα προβλήματα ασφαλείας, αφήστε που μπερδεύετε κυρίως τον κίνδυνο που μπορείτε να υπολογίσετε, αλλά όχι την ανασφάλεια που δεν μπορείτε να υπολογίσετε υπολογίσετε. Λοιπόν, όταν με ρωτάτε τι χρειάζεται για την ανθρωπιστική θεώρηση, μπορώ να σα πω τα προνόμια πρέπει να είναι τα ίδια και οι κανόνε πρέπει να είναι ίδιοι και να γίνονται σεβαστοί από τα κράτη-μέλη. Λοιπόν, για να υπάρχει ομοιομορφία, να μην υπάρχει ανθρωπιστική θεώρηση, να υπάρχει πολιτική υποδοχή για την παροχή αυτών των προνομίων ε, και για να αποφύγουμε πεθάνουν και άλλοι 50.000 φέτο. Ε, ε, Κύριε Γκάρκοφ, σας υπέβαλαν ένα ερώτημα. Θέλετε να απαντήσετε. Sorry for the... Ευχαριστώ και ζητώ συγγνώμη για τις τεχνικές δυσκολίες. Ε, πολύ σημαντικό το ερώτημα. Ε, στις 23 Ιανουαρίου την επόμενη εβδομάδα ε, ε, ε, προβλέπει το rollout για την ε, περιοχή 17 για την Ουκρανία είναι η πιο δύσκολη περιοχή για τα, ε, ως προς ε, τα σύνορα με τη Ρωσία. Στη συνέχεια έχουμε την περιοχή 19 τον, ε, την, τον Οκτώβρη, η Κίνα, Μογγολία, τα Ιβάν και ούτω καθεξής και στη συνέχεια αρχές Νοεμβρίου roll out για την περιοχή 20, για τον Μπαγκλαντές, Μπουτάν, Ινδία, Μαλδίβες, Νεπάλ, Πακιστάν και Στριλάνκα. Θα χορηγηθούν αυτά τα προνόμια λοιπόν με το rollout ε, και στη συνέχεια θα έχουμε τις περιοχές 21, 22, 23, Ανδόρα, ε, Μονακό και Σαν Μαρίνο, Ιρλανδία και Ηνωμένο Βασίλειο και τα κράτη-μέλη Σέγγεν. Ε, βάσει του χρονοδιαγράμματος τέλη Νευρίου θα έχουμε πλήρες rollout του συστήματος VS και των προνομίων που συνεπάγεται. Ε, δεν έχουν παρατηθεί σοβαρά τεχνικά προβλήματα με το κεντρικό σύστημα θεωρήσεων ούτε και από πλευρά των κρατών μελών ε, και τη ε, πρακτική υλοποίηση των προνομίων. Δεν αναμένουμε παρά αύξηση του δυναμικού για τα βιομετρικά δεδομένα που θα ενισχύσει το rollout του συστήματο και των προνομίων. Το βλέπουμε λοιπόν ότι πληρούνται όλε τι τεχνικέ προποθέσει και το σύστημα θεωρήσεων μέχρι το τέλο του 2015 θα έχει επιτυχώ αναπτυχθεί με όλα τα προνόμια που αυτό συνεπάγεται. Ευχαριστούμε. Ο κύριος Γκούρτεμπερ. Σε ό,τι αφορά την ερώτησή σα, ε, σε ό,τι αφορά τη χορήγηση θεωρήσεων στα σύνορα, πριν από κάποια χρόνια ήμουν, ε, ε, και δούλευα στην ε, ναυτιλιακή ε, φύλαξη και τότε είχαμε 10.000 ε, θεωρήσεις ε, ανά έτος για ε, μέλη ναυτιλιακού προσωπικού, τα οποία χορηγούνταν στα, στους Η διαδικασία αυτή κοστίζει πάρα πολύ δουλειά και όντως στέκει ότι οι πληροφορίες που έχει η προξενική αρχή θα πρέπει να χορηγηθούν στα σύνορα. Δεν είναι δηλαδή ε, θα λέμε τα πράγματα. Δεν μπορεί κανείς να έχει το προνόμιο του να πηγαίνει στα σύνορα και να του δίνει κατευθείαν ε, μια τέτοια θεώρηση. Αυτό σημαίνει φυσικά επένδυση σε προσωπικό, σε πληροφοριακά συστήματα, σε χρόνο, αλλά δεν μπορεί να συμβεί αυτό πάρα αυτά και ακόμα και σε δεύτερη φάση προαπαιτεί μεγάλες επενδύσεις. Άρα πρόκειται ε, για μια δυνατότητα και ένα προνόμιο αλλά με πολλές ε, συνέπειες. Αυτό που μου φαίνεται λογικό είναι να κινηθούμε σε ένα σύστημα όπως αυτό τον ε, είπα, όπου έχει κανείς το προνόμιο να κάνει την, το αίτημα πριν από κάποιες ημέρες προκειμένου να προετοιμαστεί η αίτηση χορήγησης της ε, θεώρησης από ε, τις προξενικές αρχές και να δοθεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Ελπίζω να απάντησα στην ερώτησή σας. Μάλιστα. Όσον αφορά εκείνους που είναι πρόσφυγες στα σύνορα για λόγους ταξιδιωτικούς, στις Βρυξέλλες τη διαπιστώνουμε ότι υπάρχουν κάποιοι που παρουσιάζονται στα σύνορα και σαν αίτιο ταξιδίου παρουσιάζουν θέλουν να έχουν το προνόμιο να επισκεφθούν την Πρίου για να μελετήσουν τους φλαμανδούς ζωγράφους αλλά δεν δίνουν ούτε ένα όνομα ζωγράφου. Δεν ξέρουν που βρίσκονται οι Πρίους. Μπορεί να υπάρχουν αμφιβολίες αν έχουν κάνει την παιδεία και το επίπεδο να έχουν το προνόμιο για να πάνε να κάνουν το ταξίδι αυτό και τις σπουδές. Και εκεί στις Βρυξέλλες έχουμε 1.200-1.300 το χρόνο, τους οποίους απορρίπτουμε την είσοδο στα σύνορα. 60% από εκείνους τους οποίους απορρίπτουμε είναι για λόγους ταξιδιωτικούς, περίπου 2-2,5 στατιστικά, 2,5 άτομα την ημέρα. Ε, χρειάζεται χρόνο. Ε, τους φέρνουμε σε δευτεροβάθμια εξέταση Εκεί που δεν παλύσουμε το πρόβλημα, ε, που εκεί που θα γίνουν τα διαβατήρια, γιατί δημιουργούνται ουρές, στη δεύτερη, στη δευτεροβάθμια εξέταση, όταν ε, ερχόμαστε σε επαφή και ανακρίνουμε το ΣΥΠΗΝ, το άτομο αυτό, σε ελάχιστο χρόνο, βλέπουμε ότι εφευρίσκουν οτιδήποτε για το προνόμιο να μπουν στη χώρα. Δεύτερο στοιχείο, ότι κανονικά στο ΒΙΣ βλέπουμε να αναφέρεται ο λόγος του ταξιδίου στο ΒΙΣ σχεδόν σε όλες τις περιπτώσεις μάλλον εκεί που έπρεπε να λέει λόγος ταξιδίου υπάρχει κενό. Βλέπουμε το όνομα, το τόμα, αριθμός θεώρησης κλπ. κλπ. στο VIS αλλά αυτές οι πληροφορίες συμπροματικές που μπορούν να βοηθήσουν πάρα πολύ στα σύνορα για να ληφθεί μια απόφαση γρήγορη και σωστή θα ήταν καλό αν αυτές οι πληροφορίες θα ήταν ε, ε, μέσα στο VIS. Αυτό είναι θέμα συνεργασίας με τα προξενία τα οποία είναι πολύ φορτωμένα. Απάντησα στην ερώτησή σας. Ευχαριστώ. Thank you very much. I would like to ask Ευχαριστώ. Οι υπόλοιποι ε, ομιλητές θέλουν μήπως να προσθέσουν κάτι αδικήθηκε. Ναι. Να κάνω και κάποιες ερωτήσεις προς τον κύριο Μπόνι για τα τέλη των θεωρήσεων. Αυτό για την ε, τουριστική βιομηχανία είναι πολύ σημαντικό, σημαντική πτυχή. Μια οικογένεια με τέσσερα άτομα που έρχονται στην Ευρώπη Τώρα πληρώνουν 240 ευρώ μόνο και μόνο για τι θεωρήσει, για θεωρήσεων. Δεν ξέρω τι μπορεί να συμβεί αν αυτή η πτυχή καταστεί θέμα επιτροπολογίας. Αλλά η πρώτη μου αντίδραση με πάντα, με κάθε σεβασμό προς τα κρατημέλη είναι ότι μπορεί να χρησιμοποιήσουν την ε, ε, επιτροπολογία για να καλύψουν το κόστος τους. Και τελικά θα καταλήξουμε με τέλη 80-90 ευρώ τα οποία θα δικαιολογούνται από τα προξενία με λειτουργικά, ως λειτουργικά έξοδα και τελικά θα καταλήξει η Ευρώπη να είναι ένας ε, ακριβώς προορισμός. Και ήδη είμαστε ακριβώς προορισμός με όλους τους φόρους, τα τέλη, τους δασμούς που ισχύουν στα κράτη-μέλη για την παροχή των τουριστικών υπηρεσιών. Ευχαριστώ. Ένα σχόλιο να κάνω για την ερώτηση του κ. Μπονή, για τις διευκολύνσεις, τις συμφωνίες διευκολύνσεων θεωρήσεων. Έχει μειωθεί σε 35 ευρώ. Νομίζω λοιπόν ότι αυτό είναι θετικό. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Πέτρος. Τώρα θα δώσω το λόγο στην κυρία Γιολάντα Καλαϊκό Κασίλικα από τη Γενική η Διεύθυνση Home της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ και τον εισηγήτρια για τις πρώτες ιδέες και τροπολογίες στην πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και για τη συνολική της υποστήριξη. Σας ευχαριστούμε και για την υποστήριξή σας αγαπητοί ομιλητές. Η πρόταση παρουσιάστηκε ήδη στην Επιτροπή. Ως εκ τούτου δεν θα υπησέλθω σε λεπτομέρειες, αλλά θα αναφερθώ στο βασικό στόχο της αναθεώρησης της οδηγίας που είναι να μεταρρυθμιστεί η κοινή πολιτική για τις θεωρήσεις προκειμένου να καταστεί διαδικασία εναρμονισμένη και πιο φθηνή και να προσελκύσει πιο πολλούς ε, ταξιδιώτες και να μειωθεί και το άχθος ε, στις προξενικές αρχές λαμβάνονται υπόψη οι στόχοι της κοινή πολιτική για τις θεωρήσεις για την ε, δημιουργία ανάπτυξης στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχουμε λάβει υπόψη τον βασικό στόχο της πολιτικής για τις θεωρήσεις που είναι να αποτραπεί η παράνομη μετανάσταση και να είναι ασφαλής ε, η ζώνη Σέγγεν. Η διευκόλυνση δηλαδή των ε, νόμιμων ταξιδιωτών. Να αναφερθώ σε κάποια από τα βασικά ζητήματα τα οποία αναφέρθηκαν, δεν έχω το προνόμιο του χρόνου άλλωστε. Άλλωστε πολλά από αυτά καλύπτονται στον, ε, στις αναλύσεις του κώδικα. Για το ερώτημα που αφορά τις διάφορες διαδικασίες σε ό,τι αφορά για παράδειγμα τους ταξιδιώτες ΒΙΣ. Εκφράστηκαν διάφορες απόψεις και από την εισηγήτρια. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα εξετάσει τις διτάξεις αυτές μόνο όμως αν ο απότερος στόχος της διευκόλυνσης χορήγησης και έκδοσης θεωρήσεων για τα άτομα αυτά και ιδιαίτερα των θεωρήσεων πολλαπλής πολλαπλής εισόδου, ε, επιτυχάνεται ω στόχο. Αυτό θα δώσει το προνόμιο του χρόνου στα ε, προξενία που επεξεργάζονται τις ε, θεωρήσεις, τις ε, αιτήσει αυτές. Για το θέμα του αυτοματισμού. Πώς εφαρμόζεται. Μόνο εφόσον πληρούνται οι όροι. Και εδώ έχουν ένα περιθώριο ελιγμού τα προξενία. Μόνο τότε λοιπόν θα πρέπει και θα εκδοθεί θεώρηση. Δεν υπάρχει αυτοματισμός. Μόνο εφόσον πληρούνται όλοι οι όροι. Για δυνατότητα συμπλήρωσης ε, στο ίντερνετ της αίτηση. Αυτό ήδη διατίθεται ως δυνατότητα από διάφορα κρατημέλη, από προεξονικές αρχές, χρήσιμο και ωφέλιμο αυτό το πλεονέκτημα γιατί πρέπει να πούμε ότι υπάρχουν κάποιες χώρες που έχουν ακόμα δυσκολίες συνδεσιμότητα στο διαδίκτυο, άρα θα πρέπει να υπάρχει δυνατότητα συμπλήρωσης ε, γραπτού εντύπου. Για τα τέλη. 60 ευρώ είναι το ποσό του τέλους. Το ίδιο και για το τέλος υπηρεσιών μέχρι 30 ευρώ. Αυτό λοιπόν αποτελεί το μέγιστο που μπορεί να επιβληθεί ως τέλος στον ετούντα. Τι έκανε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Κάποια από τα προαιρετικά waiver έχουν καταστεί υποχρεωτικά και αυτό θα οδηγήσει και θα έχει το προνόμιο ότι θα υπάρχει πιο πολύ ομοιόμορφη εφαρμογή γιατί όπως έχουν τα πράγματα είναι άνηση η αντιμετώπιση των ετούντων για το 70% όλων των αιτήσεων ε, πληρώνουν 35 ευρώ βάσει των ε, συμφωνιών διευκόλυνσης θεωρήσεων. Και αυτό είναι σημαντικό σε τέτοιες εποχές ε, δυσνομικής στρατητάς. Δικαίωμα ένστασης. Αυτό το προνόμιο εισήχθη στο τρέχοντα κωδικό θεωρήσεων και διαδικασίες παράβασης κατά των 100 μελών αυτό εισήχθη σε δικασία από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή γιατί συνάδει με το χάρτη θεμελιδών δικαιωμάτων και πλέον αυτό το προνόμιο καλύπτεται. Εξωτερική παροχή υπηρεσιών, πολλά σχόλια για το θέμα αυτό. Ξέρετε ότι το εξηγήσαμε και στο παρελθόν. Είναι η άποψη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ότι η πρόσφυγη σε τέτοιους εξωτερικούς παροχούς υπηρεσιών ε, διευκολύνει τελικά την κατάθεση της αίτηση και δίνει το προνόμιο στην, ε, ε, στα προξενία ότι μπορούν να κάνουν πιο ενταλεχή έλεγχο των ατόμων που για πρώτη φορά υποβάλλουν τέτοια αίτηση. Είναι θετικά λοιπόν τα αποτελέσματα και τα προνόμια που προκύπτουν. Εδώ λοιπόν κάναμε κάποιες προτάσεις στην μεταρρύθμιση για να εξασφαλίσουμε και αυτή τη διάσταση των παροχών εξωτερικών υπηρεσιών. Αλλά δεν πιστεύουμε τελικά ότι αυτό θα βοηθήσει ούτε τα προξενία ούτε και τους ετούντε. Για τους διάφορους τρόπους ε, συνεργασίας μεταξύ προξενείων η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θέλει να δοθεί ένα ευέλικτο πλαίσιο. Έχουμε τις διδάξεις για τα κοινά κέντρα που δεν είχαν ακόμα χρησιμοποιηθεί επαρκώς από τα κράτη-μέλη. Εξακολουθεί να προβλέπεται η δυνατότητα, αλλά θα δώσουμε το προνόμιο πιο ευέλικτης διαμόρφωσης, ανάλογα με τις τοπικές ιδιαιτερότητες. Τα κράτη-μέλη θα έχουν το προνόμιο να αποφασίζουν ποια είναι η πιο σωστή μορφή προξενικής συνεργασίας. Τέλος, ναι. Για τις ανθρωπιστικές ε, άδειες ή θεωρήσεις, άδειες τις αποκαλεί η θεωρησεις αδειες της αποκαλει Επιτροπή. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή απέφτεινε έκκληση προς τα κράτη-μέλη για την Ευρωπαϊκή Ατζέντα για τη μετανάστευση το Μάιο να χρησιμοποιήσουν όλα τα ένομα μέσα για τα άτομα που χρειάζονται προστασία. Αυτό περιλαμβάνει α, χορηγίες, άντιες και το καθεξής. Επίσης, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σύστησε να δημιουργηθεί ένα σύστημα για την εκ νέου εγκατάσταση τέτοιων ατόμων που προβλέπει και τέτοιες αποφάσεις για εισδοχή βάσει κάποιων ελέγχων μεταξύ των οποίων και ειδικών ελέγχων. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν θεωρεί ότι αποτελεί ο κώδικα για τι θεωρήσει το σωστό ένομο μέσο για να ρυθμίσουν τα πράγματα αυτά, που αναφέρθηκε και από κάποιου ομιλητέ. Ο κώδικα για τι θεωρήσει βασίζεται σε αυτή την αρχή των 90-180 ημερών Όλοι οι κανόνες που ισχύουν για την έκδεση μιας θεώρησης Σέγγεν δεν καλύπτουν τέτοια άτομα τα οποία εξ ορισμού πρέπει να μείνουν παραπάνω στην Ευρωπαϊκή Ένωση και άρα θα πρέπει να έχουν άδεια παραμονής γιατί σε κάθε περίπτωση θα μείνουν για μεγαλύτερη διάρκεια. Αυτά λοιπόν τα σχόλια και σας ευχαριστώ για το προνόμιο που μου δώσετε να μιλήσω. Thank you very much. Uh, now I... Ευχαριστώ. Θα δώσω το λόγο στην κυρία Μόρια Ρόζα, πρόεδρο του Σωμάτου Εργασία και Θεώρηση τη Λετωνική Προεδρία, να μα ενημερώσει για την κατάσταση όσον αφορά τι εργασίε του Συμβουλίου. Ε, godātie deputāti, dārgie kolēģi, vispirms vēlos pateikties par sniegto iespēju ņemt dalību komitejas sanāksmē. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που μας καλήσατε να πάρουμε το λόγο. Θα ήθελα να σας ενημερώσω για τις εργασίες ε, στο Συμβούλιο για το πακέτο των θεωρήσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ξέρουμε ότι πρόκειται για την πρόταση για την αναθεώρηση του κώδικα των θεωρήσεων και για την πρόταση για τα ταξίδια, για τις θεωρήσεις ταξιδίων και για τις αλλαγές που γίνονται στον κανονισμό. Να απευθυνθώ και να στραφώ καταρχάς στο θέμα του κώδικα θεωρήσεων. Θα ήθελα να αναφέρω ότι με τον κώδικα αυτό έγινε το πρώτο μεγάλο βήμα για την κοινή πολιτική για τις θεωρήσεις. Δημιουργήθηκε ένα αναρμονισμένο σύστημα για τις νόμιμες, για τη διευκόλυνση των νόμιμων μέσων ταξιδιού στην Ευρωπαϊκή Ένωση και για ως ένα μέσο καταπολέμησης των παράνομων εισόδων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τον Απρίλιο του περσινού έτους κατέθεσε την πρότασή της και αυτό αποτέλεσε το επόμενο σημαντικό βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση. Χρειαζόμαστε μια κοινή πολιτική για τις θεωρήσεις η οποία θα συνεχίσει να ενημερώνεται προκειμένου να καταστεί η Ευρωπαϊκή Ένωση πιο ελκυστική για υπηκόους τρίτων χωρών. Προκειμένου να βελτιωθούν τα ζητήματα της ασφάλειας και της αξιοπιστίας. Τους τελευταίους μήνες λοιπόν συνεργαστήκαμε και εμείς προκειμένου να επιτευχθούν με τον καλύτερο τρόπο αυτοί οι κοινοί στόχοι για αντιμετώπιση τη πρόταση τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή από την Ομάδα Εργασία του Συμβουλίου και η επεξεργασία τη πρόταση ξεκίνησε πέρσι τον Απρίλιο, όπω σα αναφέρα. Και ήδη τότε, με την ε, Ελληνική Προεδρία, στη συνέχεια με την Ιταλική Προεδρία, επεξεργάστηκαν την πρόταση αυτή και κατά τη διάρκεια της Λετωνικής Προεδρίας στις αρχές του έτους τον Ιανουάριο ολοκληρώθηκε η κατάρθρον εξέταση του κειμένου η οποία είχε ξεκινήσει ήδη από τις δύο προηγούμενες προεδρίες. Η πρόταση λοιπόν αυτή για την Λετωνική Προεδρία είναι εξαιρετικά σημαντική γιατί της δίνουμε προτεραιότητα. Κάναμε πολλές συμβαστικές προτάσεις και είχαμε έντονη ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των κρατών μελών, προκειμένου να συλλέξουμε όλες τις διάφορες απόψεις, τις διαφορετικές απόψεις και συνολικά στην ομάδα εργασίας για τις θεωρήσεις συνεδριθήκαμε πέντε φορές κατά τη διάρκεια της Λετωνικής Προεδρίας. Προκειμένου να δομήσουμε λοιπόν και να διαθράσουμε τις συζητήσεις, κάναμε συμβιβαστικές προτάσεις για τα επόμενα θέματα. Καταρχάς, σε ό,τι αφορά τον ορισμό του καταχωρισμένου ετούντα. Ο, ο ορισμός του κανονικού ταξιδιώτη στο σύστημα ΒΙΣ, καθώς και οι προβλεπόμενες ελαφρύνσεις για τους ετούντες αυτούς. Σε ό,τι αφορά τώρα το θέμα των προθεσμιών για την διαβούλευση πριν την ε, αίτηση και πριν τη λήψη απόφασης. Και για το σημείο αυτό, όπως ε, τα θέματα της ασφάλειας ταξιδίου και του τέλους ε, θεωρήσεων. Και εδώ προετοιμάσαμε συμβαστικές προτάσεις. Θα πρέπει να διευκρινίσουμε ότι ασφαλώς δεν απασχολούν μόνο αυτά τα ζητήματα. Αλλά επειδή δεν έχουμε πολύ, χρόνο και πολλά μέσα, θεωρούμε ότι ήταν σκόπιμο να περιοριστούμε σε έναν περιορισμένο αριθμό συγκεκριμένων ζητημάτων. Επιλέξαμε λοιπόν τα συγκεκριμένα θέματα βάσει της σημασία τους για τα κρατημέλη. Με κάθε μέσο προσπαθήσαμε να λάβουμε υπόψη όλε τι απόψει όλων των κρατών μελών κατά τη σύναψη των συμβαστικών προτάσεων. Στου συμβασμού τώρα έχουμε το θέμα της ισορροπίας μεταξύ της ε, διευκολυμένης παροχής θεωρήσεων σε ταξιδιώτε Bona και των θεμάτων ασφαλείας και των μέσων εξασφάλισης της ασφαλείας. Και σκοπός ήταν να πετύχουμε μια σημαντική πρόοδο σε ό,τι αφορά τα θέματα αυτά. Μπορούμε να ισχυριστούμε ότι υπήρξαν λοιπόν συγκεκριμένες εξελίξεις και συγκεκριμένη πρόοδος στα πιο πολλά ζητήματα τα οποία εντοπίσαμε ως προτεραιότητες. Σε ό,τι αφορά για παράδειγμα τον ορισμό, της διευκολύνσης αλλά και τις προθεσμίες. Στο σημείο αυτό θα ήθελα να υπογραμμίσω ότι οι συζητήσεις για την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στο Συμβούλιο συνεχίζουν να διεξαγάγονται οι συζητήσεις ε, και οι εργασίες είναι εντατικές. Το Συμβούλιο δεν κατανοεί απόλυτα πόσο σημαντικές είναι οι προτάσεις αυτές για την κοινή πολιτική θεωρήσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και επίσης γενικότερα η πρόταση αυτή είναι πάρα πολύ σημαντική για τον τουρισμό, τις εξωτερικές θέσεις, ε, την ανάπτυξη. Και τέλος, θα ήθελα εκ νέου να τονίσω το εξή. Το θέμα αυτό αποτελεί θέμα προτεραιότητας για μας, προκειμένου να είναι ισορροπημένη τελικά η πολιτική για τις θεωρήσεις και η Ευρωπαϊκή Ένωση να καταστεί πιο ελκυστική για τους επικόστρες των χωρών, για τους νόμιμους ταξιδιώτες μιλάω ασφαλώς. Εκ παραλληλού, θα πρέπει να αποτρέψουμε τυχόν παραβιάσεις και να διασφαλίσουμε με το μέσο αυτό ε, στον χώρο του Σέγγεν υψηλά πρότυπα ασφαλείας. Η Λιθωνική Προεδρία λοιπόν θα υποβάλει την πρόταση αυτή στη, στο τρίο, στην Τρόικα των Προεδριών, στο Λουξεμβούργο συγκεκριμένα και θα συνεχίσει το Λουξεμβούργο να ασχολείται με το θέμα αυτό. Ευχαριστώ πολύ. Thank you. Thank you very much. Ευχαριστώ, ευχαριστώ πολύ. Τώρα πρέπει να καταλήξουμε σε συμπεράσματα. Ε, κυρία Φαϊούμ, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους ομιλητές μέσω των οποίων μπορέσαμε να συζητήσουμε αυτή την, αυτό το πολύ σημαντικό θέμα ανταλλάξαμε πολλές ιδέες, συζητήσαμε τα αναγκαία μέσα που χρειαζόμαστε για να εξυγχρονίσουμε το σημαντικό αυτό πακέτο μέτρων για τις θεωρήσεις σας διαβεβαιώ ότι θα λάβω υπόψη μου όλα τα σχόλιά σας ακούσατε τις πρώτες ιδέες μου τις διαβάσατε επί χάρτου και πράγματα που δεν εξετάσαμε σήμερα. Δεν θα θέσω τώρα τις ερωτήσεις παρόλο που έχω νέες ερωτήσεις και νέες ιδέες. Θα τις συζητήσω ξεχωριστά. Φερρυπίν, τα διάφορα δικαιολογητικά, να μην υπάρχει πλέον έγγραφο για την ιατρική ασφάλιση. Το υποστηρίζω, όπως και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν εκαλύφθη αυτό όπως και άλλα θέματα, αλλά έχουμε ακόμα πολλές δυνατότητες συζήτησης. Ε, μία σκέψη κλείνοντας πρέπει να λάβουμε υπόψη και τις προπτικές για τον ετούντα. Θέλουμε να διευκολύνουμε τον ταξιδιώτη. Δεν θέλουμε να αυξήσουμε το κόστος για τον ταξιδιώτη, θέλουμε να καταστήσουμε ελκυστική την Ευρώπη για την οικονομία, για την νεολαία, για τον τουρισμό, για όλες τις κατηγορίες των ταξιδιωτών. Προς αυτή την κατεύθυνση θα κινηθώ με κάθε μέσο και δεν θα εστιαστώ τόσο πολύ α, επί της ασφαλείας, διότι σήμερα συζητήσαμε μετανάστες και λοιπά και αυτά που συμβαίνουν στην Ευρώπη και εστιάζονται όλα αυτά, όλες οι συζητήσεις της ασφαλείας και όχι να γίνει ελκυστική η Ευρώπη για τους ε, τουρίστες και να προσπαθήσουμε να διευκολύνουμε τους ταξιδιώτες. Ευχαριστώ πάρα πολύ και προσβλέπω ε, σε συνεργασία με όλους. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ τους διακεκριμένους προσκεκλημένους μας σας ευχαριστώ για τα πολύ ενδιαφέροντα πράγματα που μας είπατε και εδώ κλείνω το μικρόφωνο της Προέδρου και την ακούμε. Reporter. And now we need one minute break because we have to Λοιπόν, θα πρέπει να αλλάξουμε τώρα θέσεις. Θα δημιουργηθεί μια αναστάτωση. Ευχαριστώ πολύ για αυτή τη συζήτηση. Σε ένα λεπτό θα ξεκινήσουμε την επόμενη φάση των συζητήσεων. we invite uh, our next speakers, uh, Mrs. Lais Martens. κυρία Λάις Μάρτενς είναι η επόμενη που Και Yes. Yes. Yes. Yes. Thank you. Thank you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 Maybe. Yes. Okay. Dear colleagues, may I ask you to take a seat? Καθίστε παρακαλώ. How do pam pam pam. Okay, we we start the... Ξεκινάμε τη το δεύτερο μέρος συνεδριάσεως μας. May I politely ask you to finish? to fi we we finish we just already finish our break and Τελείωσε το διάλειμμά μας και ξεκινάμε το δεύτερο μέρος της ακροασής μας που θα εστιαστεί επί της προτάσεως για τη νέα θεώρηση για τον τουρισμό, νέο τύπος θεώρησης που επιτρέπει τον κάτοχο να ταξιδεύει εκτός του χώρου Σέγγεν για πάνω από 90 μέρες σε μια περίοδο 180 ημερών υπό τον όρο ότι δεν χρησιμοποιεί κάθε μέσο για να μείνει σε μια χώρα πάνω από 90 μέρες. Δίνω το λόγο στον κύριο Ορτόφο για μια σύντομη για μια σύντομη παρουσίαση και μετά θα ακούσουμε τους ομιλητές. Σας υπενθυμίζω ότι πρέπει να τηρήσετε το χρόνο που σας διατίθεται. Και ο οχτωφε έχει το λόγο. Ευχαριστώ κυρία Αντιπρόεδρε. Πριν δώσω το λόγο στους παρεμβαίνοντες θα πω κάποια λόγια για την βίζα αυτή που αναφέρατε. Είναι νέο δημιούργημα, νέο μέσο που επιτρέπει στο δικαιούχο να παραμένει μέχρι ένα χρόνο στο χώρο Σέγγεν ή και δύο χρόνια αν ανανεωθεί η θεώρηση. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην πρότασή της επέμενε επί των ωφελών των οικονομικών άμεσων και μέσων της θεωρήσεως της τουριστικής που μπορεί να κυκλοφορεί κανείς 500 εκατομμύρια μέχρι ένα δις ε, ευρώ το χρόνο μπορεί να παράγει για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ανέφερε επίσης ότι πρέπει να υπάρχουν κριτήρια επιλεξιμότητας είναι αρκετά υψηλά τα κριτήρια αυτά για να περιορίζεται, να μειώνεται ο κίνδυνο παράνομη μετανάστευση με αυτό το μέσο και να δημιουργηθεί ένα κίνδυνο ανασφάλεια που πρέπει να είναι ε, κοινή μέρημνα έναντι των πολιτών μα. Αυτή η πρόταση θεωρείται κενό ασφαλείας και ένα κίνδυνο παράτυπης μεταναστεύσεως που συνδέεται με την ύπαρξη διμερών συμφωνιών που έχουν συναυτεί σήμερα μεταξύ των κρατών μελών και κάποιων τρίτων χωρών όπω παραδείγματο χάρη η Νέα Ζηλανδία ή η Ιαπωνία. Το λέω άμεσα ότι προσωπικά σπανίω άκουσα να μιλάμε για παράνομε ροέ μεταναστών ή κινδύνου από αυτέ τι χώρε που πενθυμίζω το ε, ποσοστό ανάπτυξη και το ΑΕΠ είναι πολύ ψηλότερο, ο ρυθμό ανάπτυξη και το ΑΕΠ είναι πολύ ψηλότερο από τη Ευρώπη, άρα ο καθένα μπορεί να αμφιβάλλει. Αλλά θα, θα είχα αμφιβολίε όσον αφορά τον οικιστικό χαρακτήρα τη θεωρήσεω για τον Ιαπωνέζο, τον Νεοζηλανδό τουρίστα, που ε, δεν πρέπει να περάσει μέχρι τώρα από τέτοιες διαδικασίες. Ε, είμαι πολύ προσεκτικός όσον αφορά τα θέματα της ασφαλείας και είχα την ευκαιρία αυτό να το υπογραμμίσω και κατά την παρουσίαση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις 5 Μαρτίου ε, και η περιφερειακή αστάθεια είτε στη Μέση Ανατολή, είτε στην Υποσαχάρη Αφρική, είτε στο κέρας Αφρικής και οι τρομοκρατικές απειλές κατά της Ευρώπης είναι πιο μεγάλες παραποτέ τώρα. Δεν μπορούμε λοιπόν να μην κάνουμε έναν προβληματισμό όσον αφορά την διάσταση ασφαλείας, την πολιτική χορηγήση θεωρήσεων και αυτός ο προβληματισμός εφαρμόζεται βέβαια και στο μέσο αυτό τη θεώρηση ε, κυκλοφορίας και ταξιδίων εντός Ευρωπαϊκή Ένωσης. Ο κίνδυνος της παράτυπης μετανάστασης ήδη υφίσταται με την ε, θεώρηση μακράς διαρκείας. Αλλά θα ήταν αφελές να ισχυριζόμεθα ότι θα ήταν ανύπαρκτος ε, για την θεώρηση αυτή της κυκλοφορίας. Γι' αυτό θα πρέπει αν ε, είναι ξεπέραστο εμπόδιο η πρόθεση διαμονής. Μήπως θα μπορούσε να κυρωθεί το ρεπορικό εισιτήριο και η κράτηση μετά την απόκτηση της θεωρήσεω. Εξυπακούεται και αυτό και για τα μέσα διαβίωσης. Μήπω είναι απίθανο να υπάρχει ένα ποινικό δίκτυο που πλαστογραφεί ε, τα μισθολόγια και τι αποδείξει πληρωμή μισθού και, και κάποιοι, κάποιες ομάδες έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον. Οι καλλιτέχνες, οι αθλητές, οι ξενοδόχοι, η βιομηχανία πολυτελείας, θεωρώντας ότι αυτή η θεώρηση θα μπορούσε να διευκολύνει τις μετακινήσεις και τον οικονομικό θετικό αντίκτυπο που θα ήταν κάτι χρήσιμο για τα κρατημένη. Λοιπόν, εγώ από τους σημερινούς παρεμβαίνοντες θα ήθελα να ακούσω να μας πούν σε τι ε, επιτυχάνει τη ισορροπία μεταξύ οικονομικού δυναμικού και της, δυνα... της ανάγκης για την ασφάλεια από την άλλη. Λοιπόν, χαίρομαι που η κυρία Λίζ Μάρτενς είναι παρούσα, που γνωρίζει πολύ καλά τα θέματα ατιστικά, τα καλλιτεχνικά συγγνώμη, διότι είναι πρόεδρος μιας ε, της Ίθμαν που παρουσιάζει ε, έργα καλλιτεχνικά και επιφορτισμένη για τη διοργάνωση διαφόρων εκδηλώσεων ε, και φεστιβάλ. προσθέτω η κυρία Μαρτένς επίσης είναι υπεύθυνη για... είναι σύμβουλος όσον αφορά τους εργοδότες των καλλιτεχνών και γνωρίζει πολύ καλά τα θέματα αυτά της συγκεκριμένης θεωρής από την αρχή του προβληματισμού. Χαιρετίζω και την παρουσία του Μισελ Ντεζεζέρ, ο οποίος, όπως υπενθύμησε προηγουμένως, εξετέλεσε πολλά διπλωματικά καθήκοντα ε, ε, σε ένα περίπλοκο ε, τομέα και έχει εμπειρία όσον αφορά την κεντρική διοίκηση έχει εμπειρία λοιπόν και επιτόπια και διοικητική και είναι απαραίτητη για τον προβληματισμό μας. Ευχαριστώ την κυρία Γιολάντα Αγκαλέδο και την κυρία Μυραρός ε, που αντιπροσωπεύουν την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την Προεδρία τη Λετωνική. Αντίστοιχα, εδώ κυρία Αντιπρόεδρε, αυτά που ήθελα να πω και να μοιραστώ μαζί σας στην αρχή αυτή της συζητήσεων και θα αφήσω το λόγο στους ε, παρεμβαίνοντες. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Τώρα η κυρία Λις Μάρτεν σε 10 λεπτά. Ευχαριστώ. Θα ήθελα να ευχαριστήσω το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για την πρόσκληση στη σημερινή ακρόαση. Εγώ εκπροσωπώ ε, τον ε, τομέα των ε, καλών τεχνών και της μουσικής. Μάλλον των τεχνών και της μουσικής θα θέλαμε να τοποθετηθούμε για την τουριστική θεώρηση, διότι είναι κέρια σημασίας για τους καλλιτέχνες και για τους μουσικούς. Εργάζομαι σε μια εταιρεία που λέγεται Eastman, ίσως γνωρίζετε την εταιρεία, τον κύριο Σεχκό. Η έδρα μας είναι στο Βέλγιο και ε, όσο ε, χορευτής και χορογράφος είχε μια πολύ μακρά σταδιοδρομία και έχουν βραβευτεί πολλές παραγωγές του. Ε, ως επίσης παραγωγό το ξέρετε από την Άννα Καρένινα και Επίση, ήταν και πρέσβη ε, καλή θέλης ε, του, της UNESCO το 2015, συμμετείχε στο Σεκ του Σολέγε, στην ε, Σκάλα του Μιλάνου, στην Όπερα των Βρυξελών. Τώρα κάποια στοιχεία για την εταιρεία το 2013 είδαμε 120 παραστάσεις από διάφορους τομείς της τέχνης, πολλές διαφορετικές ειδικότητες, 13 από την Ευρώπη. Ε, και ε, φτάνουμε ε, τις 100 παραστάσεις ε, και πλέον ετησίως. Θα ήθελα να παρουσιάσω και μια παράσταση, το Puzzle, διότι πήρε βραβείο για την καλύτερη χορευτική παραγωγή παρά τα περιορισμένα μέσα. Υπάρχουν καλλιτέχνες, μεταξύ των οποίων και δύο Καναδοί από την Ιαπωνία, από την Κορέα. Έχουμε καλλιτέχνες επίσης και 70 παραστάσεις ετησίως για τα 3 τέταρτα στο χώρο Σέγγεν. Και τώρα θα σας πω πω πιο ενδιαφέροντα πράγματα, διότι έχουμε θέματα ε, με την τουριστική βίζα. Ε, Παραδείγματο χάρη, η Καναδοί καλλιτέχνη ε, πρέπει να απελευθερωθεί από έναν καταβλισμό προσφύγων. Έχουμε το χορευτή από την Κορέα που δεν μπόρεσε να μπει στο αεροπλάνο στην Κορέα, στη Σεούλ. Έπρεπε να του βρούμε νέα, νέο αεροπορικό εισιτήριο. Ο μουσικό από την Ιαπωνία αντί να χάσει τρει ημέρες ε, ε, για αποφάσεις να κάνει εργαστήρια στο Λονδίνο και παρά τα περιορισμένα μέσα μπόρεσε να ε, αντιμετωπίσει τα προβλήματα και να κάνει αυτά τα εργαστήρια. Δεν μπορούμε όμως να τους αντικαταστήσουμε τους καλλιτέχνες διότι ή έχουν ειδική εκπαίδευση ή δεν έχουμε αρκετά μέσα στη διάθεσή μας ή χρειάζονται υπερβολικά πολλές πρόβες μετά για νέους καλλιτέχνες και δεν έχουμε τα μέσα. Ε, βλέπουμε ότι η βελική κυβέρνηση μα υποστηρίζει και παραδείγματο χάρη αν οι ίδιοι οι καλλιτέχνες ε, πρέπει να πάνε στη Λισαβόνα τελικά περνάνε μέσω Βρυξελών και ε, ορισμένε φορέ χρειάζεται να ακυρώσουν και παραστάσει. Έχω κάνει λόμπινγκ σε διάφορου υπουργού για να του παρουσιάσω τα προβλήματα όμω υπάρχουν διαφορετικές ερμηνείε και υπάρχει και πανικό και συναισθηματική φόρταση από πλευρά των καλλιτεχνών γιατί υπάρχει και θέμα φήμης πέρα από τα πρακτικά μέσα. Πέρλ τώρα. Pearl, ε, ε, η Πέρλ εκπροσωπεί 700 ε, εταιρείε στον τομέα της μουσικής και των τεχνών του θεάματος. Η Ευρωπαϊκή Ένωση που αναγνωρίζεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και ε, τα μέλη μας διαπραγματεύονται και συλλογικές συμβάσεις σε, σε, σε εθνικό επίπεδο. Θα ήθελα να σας δώσω και ε, κάποιες ε, κάποια στοιχεία για τις ζωντανές παραστάσεις. Το ζωντανό θέμα είναι ένας από τους πιο δυναμικούς τομείς με τη μεγαλύτερη ανάπτυξη και εκπροσωπεί 4,2% του ΑΕΠ στην Ευρώπη και έχουμε πάνω από 70 εκατομμύρια εργαζόμενους και περίπου 20 είναι νέοι. Γιατί χρειαζόμαστε την τουριστική βίζα για αυτό το τομέα είναι στο DNA μας, το ζητάει το κοινό, ε, έχουμε περιοδίες και ε, φυσικά ε, θέλουν οι καλλιτέχνε να δείξουν τις ε, παραγωγέ του σε ολόκληρο τον κόσμο διότι τροφοδοτούνται από διαφορετικούς ε, πολιτισμούς. αυτή είναι η βασική πηγή εισοδήματο, η περιοδία δηλαδή και είμαστε όλοι πρέσβει του καλλιτεχνικού μηνύματο που θέλουμε να περάσουμε και εκπροσωπούμε τις παραστάσεις μας. για την υπηκότητα δεν έχει καμία σημασία για μας. το θέμα είναι οι δεξιότητες, η εμπειρία, τα πορτφόλια των καλλιτεχνών το background τους, ε, το πολιτιστικό μήνυμα που μεταφέρουν και ταυτόχρονα ε, εμπλουτίζεται ο πολιτισμός της Ευρώπης από όλους αυτούς τους ε, καλλιτέχνες. Τι πιστεύουμε για τη συνεργασία με διάφορες υπηκότητες. Κανείς δεν ασχολείται με την υπηκότητα των καλλιτεχνών. Αυτό που θέλουν είναι μια καλή παράσταση, καλό περιεχόμενο, καλή παραγωγή και να, υπάρχει, να ε, έχει ένα καλό όνομα το συγκρότημα ή ο θείασος. Στην ΠΕΡΛ ε, κάναμε και μία, κάποιες προσωμιώσεις ε, υπολογισμούς, διότι έχουμε το περιορισμένο αυτό μέσο τις 90 ημέρες, όπου βλέπουμε ότι ε, χάνουμε μεγάλο μέρος του εισοδήματος. Κάνουμε την προσωμείωση λοιπόν σε, τρεις, ε, σε τρία επίπεδα. Σε επίπεδο καλλιτέχνη που πρέπει μετά από τους τρεις μήνες οπωσδήποτε να επιστρέψει στην ε, πατρίδα του και μην ξεχνάμε ότι δαπανώνται 1.000 έως 2.000 ευρώ για να πληρωθούν οι θεωρήσεις, τα τέλη κτλ. Και όταν έχουμε ε, δηλαδή με 6 εκατομμύρια όταν μιλάμε για 3.000 ε, περίπου οίκους ε, καλλιτεχνικής παραγωγής στην Ευρώπη. Επίσης, δεν είναι σίγουρα τα μελλοντικά σύμβολα, τα μελλοντικέ συμβάσει και αυτό να την περαιτέρω και την ούτω ή άλλω μακροσχελή διαδικασία έκδοση θεώρηση. Δεύτερον, έχουμε έναν έμεσο αντίκτυπο. Τα τέλη για τι παραστάσει ε, κυμαίνονται από τις 7 στους 25.000 και πάλι παίρνουμε 300 οίκους παραγωγής και καταλήγουμε σε 122 75 εκατομμύρια ευρώ την Ευρώπη και ε, είναι περιορισμένες οι εκτιμήσεις που έχουμε κάνει διότι πέρα από την, ε, το, το, την Eastman έχουν ε, κάποιες εταιρείε 10 παραστάσεις το μήνα. Καταλαβαίνετε αυτό είναι πολλαπλάσιο πόσο ε, σε σχέση με το κόστος αν το υπολογίσουμε ετησίως στη συνέχεια. Ε, για ε, ε, δεν ξέρουμε τι θα γίνει με το καλλιτέχνη, αν θα έχει καλύτερη σύμβαση στη χώρα του ή αν θα επιστρέψει στην Ευρώπη. Αυτό τα λέω για τις θεωρήσεις πολλαπλών εισόδων. Υπάρχει το πρόβλημα λοιπόν του σχεδιασμού και τίθεται και ένα αμφιβόλο η βιωσιμότητα της εταιρείας παραγωγής. Επίσης υπάρχει, υπάρχουν και εξωτερικά αγαθά και υπηρεσίες που χρησιμοποιούν οι εταιρείες, ε, τεχνικοί, ηχολήπτες, ε, ε, μετακινήσεις, εστίαση, και ο, το τέλος κυμαίνεται περίπου, ε, μάλλον ο μισθός ε, ε, ε, στα 200 ευρώ την ημέρα και φτάνουμε τα 8 εκατομμύρια απώλεια λόγω ακυρωμένων παραστάσεων, παραστάσεων που δεν γίνονται αν υπολογίσουμε για τους 300 οίκους παραγωγής στην Ευρώπη. Επίσης, Ε, επίσης, ε, ε, πέρα από αυτό υπάρχουν και παράπλευρα κόστη, δηλαδή δεν, καταλα... δεν καταναλώνει το κοινό, δεν υπάρχουν χορηγίες και ούτω καθεξής. Οπότε πολλαπλασιάζεται το κόστος άνετα. Μπορούμε να κινηθούμε σε μια ψαλίδα από 500 εκατομμύρια μέχρι 3-4 δισεκατομμύρια απώλεια το χρόνο λόγω των δυσκολιών έκδοσης θεωρήσεων. Ο πολιτισμός είναι μια οικονομική μηχανή, ε, κινητήριος δύναμη, δεν είναι ένα κόστος για τις απαιτήσει. Υπάρχουν μεγάλε διαφορέ ανάμεσα στι χώρε. Υπάρχουν κάποιε όπω ε, ο Καναδά, η Νότιο Κορέα, η Ιαπωνία που ενθαρρύνουν τον πολιτισμό και δεν υπάρχει ε, κίνδυνο παράνομης μετανάστευση όπω είπε ο κύριο Οχτεφ. Η πρόταση για τη νέα τουριστική θεώρηση ζητάει εγγυήσει από την εταιρεία. Συμφωνούμε. Μιλάμε για εταιρείε ε, bona fide. Είναι νομικέ οντότητε με αναγνωρισμένη αναγνωρισμένο το ρόλο τους από τις εθνικές αρχές. Ε, επίσης, ε, το ίδιο ισχύει και για τους χώρους των συναυλιών, παραδείγματο χάρη, που προστατεύονται από συμβάσεις. Ε, υπάρχουν χρονοδιαγράμματα περιοδίας που είναι γνωστά πολύ νωρίτερα και καλύπτονται όλα η στέγαση, η εστίαση, όχι μόνο η ίδια η αλλά και η οι ημέρες ανάμεσα στις παραστάσεις. Ε, ε, σε σχέση τώρα με το μεταναστευτικό κίνδυνο, δεν αυξάνεται το κόστος, ε, διότι μιλάμε για επαγγελματίες καλλιτέχνες που έχουν μακροχρόνιες σχέσεις με τον εργοδότη και μετά θα έχουν και τις συστάσεις και αυξημένα μέσα για τις παραστάσεις τους στην Ευρώπη. Ε, για την νέα τουριστική θεώρηση και για την ε, τροποποιημένη πρόταση είναι ε, εκ των όνου για τον τομέα μας. Εδώ και 10 χρόνια κάνουμε λόμπινγκ για να έχουμε τα απαιτούμενα μέσα ώστε να είμαστε επιτυχείς. Ε, και αυτό που υποσχόμαστε αντίτιμο είναι νέες θέσει εργασία και πρέπει να συνειδητοποιήσετε ότι θα χάσουμε πάνω από ένα δις ευρώ ε, ετησίως για τις ε, χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης το ίδιο ισχύει επίσης και για τα τέλη, για το ΦΠΑ, μια σειρά από άλλα συνδεδεμένα κόστη θα ασχοληθούν να υπάρξει πολιτική θεώρηση και μπορούμε να ε, έχουμε και πολλαπλασιαστικό αποτέλεσμα, διότι υπάρχουν και μη ευρωπαϊκέ χώρε που παρόλα αυτά εφαρμόζουν το κεκτημένο του Σέγγεν. Θα χαθούν και άλλα μέσα λοιπόν έτσι. Βλέπουμε ότι θα είναι πολύ καλό το εργαλείο τουριστική θεώρηση, θα είναι win-win επικερδής για όλους, οι κυβερνήσεις, ε, οι καλλιτέχνες, οι καταναλωτές. Είναι απεριόριστο το δυναμικό που έχουμε που δεν αξιοποιείται στο έπακρον λόγω των περιορισμών στις τουριστικές θεωρήσεις. Σας ευχαριστούμε. Μισελ uh, έχουμε τώρα πρώην Γενικό Πρόξενο Γάλλο για το θέμα της προτάσεως αυτής, για την θεώρηση αυτή για τις περιοδίες. Πέρασα ε, ε, euh, euh, euh, 15 χρόνια της ζωής μου σαν γενικός πρόξενος στην Ιαπωνία, στον Καναδά, στην ακτή του Ελεφαντοστού και στην Αλγερία. Στην καριέρα μου άκουσα να μιλάνε 5-6 φορές για προβλήματα ατόμων που χρειαζόταν μία θεώρηση για πάνω από 90 ημέρες σε πολλές χώρες ε, Σέγγεν. Η πρώτη μου προσέγγιση λοιπόν είναι ότι θεωρώ ότι είναι ένα πρόβλημα το οποίο δεν είναι τόσο σημαντικό, είναι λεπτομέρεια. Υπάρχει ένα νομικό κενό, πράγματι. Συμφωνώ αλλά αυτό το νομικό κενό δεν ισχύει για όλες τις υπηκότητες με την Ιαπωνία Φερρυπίν, με τον Καναδά. Έχουμε διμερείς συμφωνίες παλιές για εξαίρεση από τις θεωρήσεις και οι περισσότερες χώρες έγκαιν έχουν αυτού του είδους τις συμφωνίες. Ένας Ιάπων που ωφελείται από διμερή συμφωνία με την Γαλλία μπορεί να παραμείνει για ένα τρίμηνο, 180 ημέρες, αν ταυτόσιμη συμφωνία υπάρχει με Ολλανδία, Βέλγιο και άλλη χώρα Σέγγεν μπορεί να παραμείνει επίσης και εκεί 90 ημέρες. Το πρόβλημα είναι αρκετά περιορισμένο θα έλεγα. Πράγματι όμως αντιμετώπισα αυτό το πρόβλημα και για πολύ συμπαθητικούς ανθρώπους, για σπουδαστές που δικαιούνται κάποιο πρόγραμμα, το Erasmus Mundus νομίζω, και μου έλεγαν ότι λαμβάνεται υπόψη ότι θέλω να περάσω δύο μήνες στη Γαλλία και μετά δύο μήνες στη Γερμανία και εν συνεχεία δεν ξέρω κάπου αλλού, στην Ισπανία Φερρυπίν. Κάθε φορά λοιπόν χρειάζομαι διαφορετική θεώρηση. Πράγματι εκεί υπάρχει ένα πρόβλημα. Πρέπει να βρεθεί μια λύση, ένα μέσο. Λοιπόν, η θεώρηση αυτή του τουρισμού ή περιοδίας είναι μια λύση. Ε, κοιτάξτε, υπό την παρούσα διατύπωση πρέπει να πω το κείμενο ακόμα και για τους ειδικού είναι δυσνόητο. Μπορώ να το καταλάβω διότι παραπέμπει σε πολλαπλές διάταξεις του κώδικα της, ε, των θεωρήσεων και δεν χρειάζεται να επαναλαμβάω τα πάντα. Υπάρχει πρόβλημα περιεχομένο όμως διότι η ορολογία θεωρώ ότι είναι ιδιαίτερα αόριστη. Ποιος μπορεί να ζητήσει με τέτοια θεώρηση, καταρχάς. Όλος ο κόσμος να το ψάξει κανείς. Οποιοςδήποτε. Δεν είναι μια θεώρηση που αφορά μόνο τους καλλιτέχνες, αλλά αφορά όλο τον κόσμο. Οι κανόνες είναι οι ίδιοι όπως οι κανόνες για ένα αίτημα για βίζα ε, Σέγγεν βραχίας δακρύας. Χρειάζεται να έχει κανείς ταυτότητα ε, φωτογραφία, να συμπληρώσει ένα αίτημα να συμφωνήσει για τη συλλογή βιομετρικών στοιχείων και μπορεί να καταθέσει ένα τέτοιο αίτημα για θεώρηση. Θα μου πείτε ότι υπάρχουν ε, σχετικά λίγοι δικαιούχοι. Εγώ ως πρόξενος τι με ενδιαφέρει, δεν με ενδιαφέρει ο δικαιούχος, αλλά ο αριθμός των ετούντων. Εγώ αυτούς που έχω απέναντί μου και τους φακέλους που έχω να εξετάσω ε, με αφορά, δηλαδή ζητούν θεωρήσεις, είναι θεωρήσεις που απαιτούνται μετά από μία εξέταση που όταν αρνούμε μία θεώρηση πιθανότατα και πολύ συχνά θα μου ρωτήσουν, θα μου ε, ζητήσει περισσότερη δουλειά από μία θεώρηση που θέλω να δώσω διότι έχω παρεμβάσεις πίσω από αυτό, ευρωβουλευτές π.χ. Θα έχω προσφυγές, θα πρέπει να απαντήσω σε πολλές ερωτήσεις μέσω και στην κεντρική διοίκηση. Θα μου πει γιατί αρνηθήκατε αυτό το μέσο, αυτή τη θεώρηση. Νομίζω ότι θα πρέπει να προσέξουμε το τι συνέπειες έχει για το προξενείο μια τέτοια θεώρηση. Είδα ότι διατηρήσαμε τις διατάξεις σχετικά με τις κατεπίγουσες περιπτώσεις. Οποιοδήποτε μπορεί να έρθει να χτυπήσει την πόρτα του προξενείου και να πείτε «Θέλω αμέσως μια θεώρηση», να μας πει είναι ένα μέσο για να κάνω ένα γύρο εντός του χώρου Σέγγεν. Πολλοί κόσμος λοιπόν να ζητήσει μια τέτοια θεώρηση. Μετά υπάρχει και ένα πρόβλημα της αρμόδιας χώρας. Αρμόδια χώρα είναι η πρώτη χώρα, η χώρα της πρώτης εισόδου. Ας φανταστούμε λοιπόν το εξή ενδεχόμενο. Ε, μία ομάδα καλλιτεχνών που έρχεται μέσω Άμστερνταμ, διότι είναι και πιο φθηνότερο πορικό εισιτήριο, για να πάει να εργαστεί στη Γερμανία, στην Ελβετία κλπ. Το προξενείο των κάτω χωρών θα πρέπει να αντιμετωπίσει το θέμα. και θα πρέπει να παρουσιαστούν δικαιολογητικά για να πάει ο θείασος να εργαστεί σε άλλες χώρες. Υπάρχει και αντίφαση στο κείμενο, διότι λέει αν πρέπει να εργαστεί αυτό το άτομο πρέπει να ζητήσει άδεια εργασίας από την πρώτη χώρα εκείνη που είναι αρμόδια για την κατάθεση του αιτήματο θεώρηση. Αν δεν εργάζεται αυτή τη χώρα, τι κάνουμε. Ε, δεν θα πρέπει να ζητηθεί τίποτα, δηλαδή. Πρέπει να φέρει την ενδειγμένη απόδειξη της πρόθεσης διαμονής. Τι είναι αυτό. Άντε να εξηγήσει κανείς σε κάποιον υπάλληλο του προξενείου τι είναι η ενδεδειγμένη απόδειξη πρόθεσης διαμονής για πάνω από 90 μέρες από τις 180. Ε, έχουμε την εντύπωση ότι υπάρχουν δυσκολίες για τη σύνταξη ενός κειμένου και η δυσκολία παραπέμπει τελικά το πρόβλημα ε, στα προξενία ζητώντας να τα βγάλουν πέρα τα προξενία και να ξεμπερδεύσουν Μετά η ασφάλεια ασθενείας. Είναι αόριστη διατύπωση. Πρέπει να καλύπτει ασφάλεια όλου του κινδύνου που κανονικά ασφαλίζονται για του υπηκού των κρατών μελών στα οποία προβλέπεται να επισκεφτεί. Αν πάει σε 5-6 χώρε αυτό ο άνθρωπο, φανταστείτε τι δουλειά έχει να κάνει ο πρόξενο, το προξενείο. Μετά πρέπει να έχει τα μέσα για ε, να επιβιώσει μια οικονομική σταθερή κατάσταση. Να δείξει ότι έχει ένα μισθό και να αποδείξει ότι έχει λογαριασμό σε τράπεζα και το περιεχόμενο του τραπεζικού λογαριασμού. Αυτό ισχύει σε κάποιες χώρε, σε κάποιε άλλες χώρες όμως αυτό το, η απόδειξη του μισθολογίου και οι αποδείξει του λογαριασμών τη Τράπεζα δεν είναι τόσο εύκολο να αποκτηθούν. Πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί. Αναφέρθηκα στην εργασία μετά και υπάρχει και εξέταση του, της υποθέσεως. Έχουμε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα, 20 μέρες, Αν έχω 20 μέρες εγώ για να καθορίσω κατά πόσο αυτός ο άνθρωπος έχει το δικαίωμα να εργαστεί εδώ ή εκεί, αυτό θεωρώ ότι είναι εξαιρετικά ε, σύντομο χρονικό διάστημα. Το πρόβλημα των καλλιτεχνών ποιο είναι. Σας εμπιστεύομαι κυρία μου. Ο οργανισμός σας είναι εξαιρετικά αξιόπιστος. Αλλά δεν είσαστε μόνο εσείς. Γιατί να δώσω θεωρήσεις σε καλλιτέχνες που σχετίζονται με εσά και όχι σε άλλους. Πρέπει να αποφύγουμε τη διάκριση. Για να αποφύγουμε τη διάκριση πρέπει η οδήποτε οργανωτή περιοδίων καλλιτεχνικών να τον θεωρήσουμε σαν ικανό και κατάλληλο να καταθέσει μια αίτηση για χορήγηση θεωρήσεως. Μετά δίνουμε δικαίωμα ιονή διαμονής στον χώρο Σέγγεν. Αυτό ισχύει για τους τουρίστες. Αν έχω ένα φίλο, ο οποίος μένει στη Γαλλία και από την άλλη πλευρά των συνόρων στο Βέλγιο, αν με καλέσει, διότι μια πρόσκληση είναι και αυτή δικαιολογητικό. Με καλεί τρει μήνε στη Γαλλία και τρει μήνε στο Βέλγιο, εδώ απέναντι, στον δρόμο απέναντι. Έτσι μπορώ να μείνω δύο χρόνια στο χώρο Σέγγεν με αυτό το μέσο. Και αν κάποιος έχει αυτό το δικαίωμα, θα έχουμε πολλά προβλήματα να μπορέσουμε να του πούμε να εγκαταλείψει την, το χώρο. Ε, πρέπει να είμαστε αρκετά προσεκτικοί. Και στα δύο χρόνια μπορούν να συμβούν πολλά πράγματα όσον αφορά τα θέματα ασφαλείας. Θα πρέπει ίσως να θετήσουμε πιο συνετή προσέγγιση, να το ψάξουμε, να είμαστε πιο συνετοί. Στον παρόντα κώδικα των θεωρήσεων υπάρχει δυνατότητα παρατάσεως μιας θεωρήσεως Σέγγεν που έχει χορηγηθεί. Άρθρο 33. Γιατί να μην προσανατολιστούμε περισσότερο προς αυτό το μέσο, προς αυτή την κατεύθυνση. Α, να παρατείνουμε μια θεώρηση Σέγγεν ούτως ώστε να παραμείνουμε σε ένα ισχύον πλαίσιο. Εδώ δημιουργούμε κάτι το οποίο αισθάνομαι έτσι ότι είναι τεράστιο ε, σε σχέση με τις ανάγκες και ανοίγουμε μια πόρτα και για να το πω έτσι ειλικρινά δεν ξέρω τι κρύβεται πίσω από την πόρτα. Ευχαριστώ. Okay, thank you very much. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Τώρα έχουμε το γύρο απαντήσεων. Έχει το λόγο. Ε, ευχαριστώ. Αναρωτιόμουν αν ο κύριος Ντεγιάγκερ, λέει ο κύριος Ντεπρούσε, όχι Ντεζέγκερ, Ντεγιάγκερ λέμε ε, εδώ στο Βέλγιο. Εσείς το, το προφέρετε αλλιώς στη Γαλλία. Συγγνώμη, φλαμανδός, ε, Φλαμαντικής καταγωγής, δεν είσαστε. Καλά τα λέω. Ντεγιάγκερ κύριε Οχτεφέ, Ντεγιάγκερ, όχι Ντεγιάγκερ. Μήπως ήσασταν εισαγγελέα σε προηγούμενη ζωή. Διότι ε, ε, ένα ε, πολύ ισχυρό κατηγορό εδώ πέρα. Όχι αστείευομαι. Ξέρετε, εγώ δεν θα υπερέβαλα τόσο πολύ. Παρόλα αυτά, αυτά που είπατε για τα 33 με ενδιαφέρουν και μπορούμε ε, να δούμε αν ε, με το νέο μηχανισμό, τα νέα μέσα, έχουμε ε, μία μεγαλύτερη ευελιξία. Λοιπόν, έχω προφανέστατα διάφορα ερωτήματα που εν μέρει συμπίπτουν με τα δικά σας. Όπως και εσείς, με εντυπωσιάζει που οποιοδήποτε μπορεί να υποβάλει αίτημα. Συγγνώμη, αλλά αυτά τα μέσα που έχουμε στη διάθεσή μας ε, δεν έχουν ακριβή εμβέλεια, διότι επιχειρηματικός πώς ε, βλέπουμε ότι δεν υπάρχει ταυτοποίηση των ανθρώπων και άρα και των μέσων που μπορούν να χρησιμοποιήσουν. η απόδειξη της πρόθεσης ε, μου φαίνεται έως και αστείο. Ε, δίκη προθέσεων δηλαδή. Πρέπει κάποιος ε, να τεκμηριώσει την πρόθεση που έχει να διαμείνει για κάποιο καιρό σε κάποια κράτη-μέλη. Αυτά λέει το γαλλικό κείμενο, μα είναι αστείο. Ε, αποδεικτικά μέσα για την πρόθεση κάποιου. Πώς θα έχετε αποδεικτικά μέσα για την κράτηση, ναι, αλλά μέχρι εκεί. Ε, νομίζω ότι είναι στοιχειώδες ε, το να θεωρήσουμε ότι δεν υπάρχουν εμπράκτος τα μέσα για να αποδείξει κανείς κάτι τέτοιο. Ε, ζητώ συγγνώμη να μας εξηγήσει ο, ο εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, μου φαίνεται, τι να σας πω, ε, ότι ήταν λίγο ελαφρόμυαλη η πρόταση. Δεν υπάρχουν λοιπόν τα μέσα στη διάθεσή μας για να υλοποιηθεί αυτό. Για να περάσουμε στα επόμενα ζητήματα. Με τα νέα μηχανισμό και τα νέα μέσα ε, μπορούμε να απαλλαγούμε από αυτή την έγκριση για ένα χρόνο παράταση ε, άλλους 12 μήνες ε, για να μην μείνετε 90 μέρες σε διάστημα 190 μερών ε, στην ίδια χώρα. Μάλιστα, πολύ ωραία. Και μετά τι θα γίνει, αν μετά αυτά τα δύο χρόνια υποβάλει κάποιο ένα νέο αίτημα χωρίς να έχει φύγει από το χώρο ε, Σέγγεν, γιατί δεν μας λέτε ακριβώς τι συμβαίνει σε αυτή την περίπτωση. Μπορεί να φύγει κάποιος από εκεί που είναι, μέσα στο χώρο Σέγγεν, να υποβάλει ένα αίτημα, το αποκλείεται αυτό, το προβλέπετε ή το λέτε κάπου και δεν το καταλάβαμε, διότι ε, Εάν θέλετε κάποιος να παραμείνει μόνιμο, ας ε, πείτε ότι δίνεται αόριστη άδεια διαμονής. Αλλά τα μέσα όπως τα περιγράφετε τώρα δεν επιτρέπουν να ξέρουμε τι ε, εμποδίζει αυτόν που είναι στο χώρο Σέγγεν και που έχει παρατείνει τη διαμονή του με τα υφιστάμενα μέσα για ένα χρόνο να υποβάλει και νέο αίτημα. Ε, θα αναγνωρίζω λοιπόν ότι ε, ε, μπορεί εσείς να είσαστε σοφότεροι μόνο και μόνο λόγω αριθμητικής υπεροχής. Τι να πω εγώ φτωχός ευρωβουλευτής, δεν έχω και τα μέσα στη διάθεσή μου. Ε, yeah, Mr. Ortofo, eh, you have the floor. Κύριε Σαχτεφέ. Oui, en tant que rapporteur, madame la vice-présidente, je naturellement ε, θα έχω πολλά ερωτήματα. Θέλω να υποβάλω ένα ερώτημα προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ξέρετε ότι με την πρότασή σας έχουμε ερωτηματικά για το θέμα του πεδίου των δικαιούχων, διότι ο αριθμός τους είναι ε, τουλάχιστον αβέβαιος. Ε, ερωτηματικά για τον αριθμό, για τα οικονομικά μέσα που θα εξοικονομήσουμε ε, και για την διάσταση της ασφάλειας. Ζήτησα εγώ αξιολόγηση αντικτύπου ε, ήδη, διότι κατά τη γνώμη μου δεν μπορούμε να δημιουργήσουμε νέο μηχανισμό θεώρησης χωρίς να γνωρίζουμε ακριβώς τον αντίκτυπο. Σε ποιο σημείο βρίσκεται η αξιολόγηση αντικτύπου, χρησιμοποιείτε όλα τα μέσα που έχετε στη διάθεσή σας. Ε, παιδί εφαρμογής και αριθμός των δικαιούχων. Γράφεται ότι αυτό μπορεί να έχει σχέση και με τους τουρίστες. Όμως, όπως είπε ο πρώην πρόξενος, παρότι είναι φλαμαντικής καταγωγής, ε, είναι γαλλικής ε, υπηκότητας, είναι Γάλλος υπήκος, λέει ότι μπορεί να είναι τουρίστες. Δεν μπορούμε να φανταστούμε λοιπόν εκατοντάδες, εκατομμύρια δικαιούχους. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τις Υπηρεσίες Εγκύτητας λοιπόν προέβλεψε ότι θα ε, ασφικτιούν τα προξενία λόγω περιορισμένων μέσων, όπως πολύ σωστά ε, ακούσαμε νωρίτερα. Βλέπουμε ότι ε, αυτές, αυτού του είδους οι θεωρήσεις ανταγωνίζονται τις άδειες διαμονής που εκδίδουν τα κράτη-μέλη και αυτό από πλευράς κοινωνικών δικαιωμάτων μπορεί να έχει σοβαρό αντίκτυπο. Είναι κάποιο και μετακινείται και δουλεύει στο χώρο Σέγγεν τι συμβαίνει γιατί αυτή η περίπτωση, πρώτη ερώτηση, δεύτερη ερώτηση προς τον, την κυρία Μάρτενς. Μπορείτε να μας πείτε συγκεκριμένα ποιες είναι οι εταιρείε οι ευρωπαϊκές που μπορούν να αναλάβουν ευρωπαϊκή περιοδία 90 ημερών. Έχουν τα μέσα για να εγγυηθούν μια τέτοια περιοδία. Και ε, ο αριθμός των καλλιτεχνών και των επαγγελματιών που απασχολούνται από αυτές τις εταιρείες. Ε, αν πρόκειται για εταιρείες που αναγνωρίζονται διεθνώς ή περιφερειακώς, ε, όπως το ΣΕΧ και το Σολέγη, παραδείγματος, το Τσίρκο του Ήλιου, όπως είπατε και στη παρουσίασή σα, Οι μικρές οι με μικρότερα, λιγότερα μέσα μπορούν να έχουν ε, τις απαιτούμενες ε, Η Διεθνής Ένωση Τσίρκων μας ε, έδωσε ένα πρόγραμμα ε, μας λένε ότι γίνεται, υπάρχει εξέμνους σε προγραμματισμός, προβλέπονται οι καλλιτέχνες, οι επαγγελματίες, η μετακίνηση κτλ. Ωραία, υπάρχει το επιχειρηματικό σχέδιο, όμως αυτό δεν σημαίνει ότι περιοριζόμαστε ε, σε κάποιες εταιρείες ε, που ε, ούτως ή άλλως εξορισμού είναι επαγγελματίες και μόνο εκείνες μπορούν να μας δώσουν εγγυήσεις. Ε, μιλήσαμε για πιο ευέλικτα κριτήρια επιλεξιμότητας. Αναφίβολα αυτή θα είναι η τάση. Δεν μπορούμε να φανταστούμε όμως δομές ε, αναψυχής που συγκροτούνται ε, μάλλον ε, ε, εταιρείε βιτρίνας θα έλεγα που έχουν ως στόχο να παρακάμψουν τον κανονισμό και να χρησιμοποιήσουν τα μέσα τους για έκνομες ενέργειες και να επωφεληθούν από τα νομικά κοινά παρακάμπτοντας και καταχρώμενοι κάποιους κανόνες. Ε, μιλήσατε για το πεδίο εφαρμογή για τους δικαιούχου για την παράταση, για τον κατάλογο με τα παραστατικά ε, και αυτό δεν καλύπτει το κενό της ασφαλείας και εγώ είμαι πεπισμένο γι' αυτό. Μπορείτε να μου πείτε όμως εσείς τι θα προτείνατε, ποια μέσα θα προτείνατε ούτω ώστε το κοινό, δηλαδή οι εταιρείε που αναλαμβάνουν τις περιοδίες ε, ή οι διεθνεί αθλητέ που συμμετέχουν σε αγώνε κτλ ποια μέσα μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε ούτως ώστε να κυκλοφορεί κάποιο ε, πιο ελεύθερα μέσα στο χώρο Σέγγεν χωρίς όμως να υπάρξει παράκαμψη της διαδικασίας και των μέσων ε, που έχουμε. Ε, λοιπόν, για την ε, απαλλαγή μας είπατε... Μας δώσατε ένα παράδειγμα Το του φοιτητή τι πιστεύετε, μπορείτε να φανταστείτε ένα ε, σύστημα λιγότερο περίπλοκο σε σχέση με αυτή την ε, ε, θεώρηση, την νέα θεώρηση που προκύπτει τώρα η Ευρωπα... προτείνει τώρα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ευχαριστούμε κυρία Φαγιά. Yeah, um, thank you very much. I, actually will not have any Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν έχω ερωτήσεις. Νομίζω ότι εξαντλήσαμε όλα τα θέματα στο γύρο των ερωτήσεων. Νομίζω ότι η πρόταση αυτή για τις ε, θεωρήσεις αυτές αποτελεί μια καινοτομία. Ελπίζω να βελτιωθεί ως προς το περιεχόμενό της προκειμένου να είμαστε ικανοποιημένοι σε τελική ανάλυση. Θέσατε τη σημασία του Erasmus Mundus εσείς για τους καλλιτέχνες. Ε, αναφέρατε την εικόνα των ε, ε, φοιτητών που έρχονται στην Ευρώπη και μας λέτε λοιπόν ότι θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε το θέμα των ε, ταξιδιωτών αυτών και το πώς μπορούμε να ε, ικανοποιήσουμε τις ανάγκες τους. Νομίζω λοιπόν ότι σε κάθε περίπτωση δεν θα πρέπει να αφήσουμε κατά μέρος αυτή την ιδέα γιατί είναι πραγματικά υπέροχη. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ λέει η Πρόεδρος, ωραία, πολύ καλά. Έχουμε λίγο χρόνο για τις απαντήσεις. Να δώσω το λόγο στην κυρία Μάρτεντς. Σας ευχαριστώ πολύ. Άκουσα διάφορες ερωτήσεις. Καταρχάς, για τους φοιτητές. Δυστυχώς δεν μπορώ να απαντήσω. Εγώ εκπροσωπώ τον τομέα των επαγγελματικών τεχνών. Μιλάμε για καλό εκπαιδευμένους καλλιτέχνες, επαγγελματίες που ε, ασχολούνται πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα και έχουν εισοδήματα από τη διαδικασία αυτή. Για αυτό που ρωτήσατε. Όπως σας έδειξα στη διαφάνεια, έχουμε θέμα εταιρείας, ε, τοποθεσίας ε, και άρα ο καλλιτέχνης θα πρέπει να μεταβεί στη χώρα του, να ζητήσει την θεώρηση με όλα τα μέσα, με όλα τα δικαιολογητικά και κανονικά μιλάμε για ένα είδος ε, διανομής της και αυτές οι εταιρείε ναι, είναι γνωστές. Και όντω είναι μεγαλύτερο το διάστημα των τριών μηνών. Δεν εξίζει τον κόπο λοιπόν σε κάποιες περιπτώσεις να τους στείλουμε στην Κορέα, στην Ιαπωνία, στον Καναδά. Πολλές εταιρείε λοιπόν στην Φλάντρα πραγματικά πλήττονται. Να σας ε, μιλήσω για την χωραστική εταιρεία της Ανατερέζα Αντικάς επίσης και για άλλες εταιρείε ε, για μουσικές ε, ορχήστρες. Ε, μίλησα και με την φιλαρμονική. Πληττόμεθα λοιπόν. Και όταν έχουμε τέτοια προβλήματα μου λένε με τι μέσο αντιμετωπίζετε τα προβλήματα αυτά. Πώς τα αντιμετωπίζετε, τι κάνετε. Δεν φροντίζετε τους υπαλλήλου σας. Κατήστανται αυτοαπασχολούμενοι. Αν έχουν βίζα, έλθουν. Αν δεν έχουν, δεν μπορούν να έλθουν. Αυτό ίσως είναι ε, αποδεκτό μέσω για τους μουσικούς, αλλά δεν ισχύει για τις ορχήστρες, δεν ισχύει για τους χορευτές, γιατί μιλάμε για περίοδους πολλών εβδομάδων, άρα χρειάζονται πραγματικά εβδομάδες για πρόβες. Δεν επιτρέπεται αυτό μέσω μέσο της βίζας για όλους. ο Υπουργό Πολιτισμού συχνά λαμβάνει μέσα χρηματοδοτικά από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και υπάρχουν κατάλογοι σε ό,τι αφορά τα κριτήρια που πρέπει να πληρούνται. Όχι φυσικά να ισχύει αυτό για όλους, αλλά από πλευρά ε, των εταιριών μπορούν πολλά να δοθούν ως μέσα εγγύησης. Κάτι άλλο τώρα κατά πόσον υπάρχει αυτή η θεώρηση. Υπάρχει αυτό το φάσμα. Έχουμε και τις χώρες που εξαιρούνται από θεωρήσεις, οι Καναδοί, οι Άπωνες. Και όταν ε, κάνουν περιοδίες 6-7 μηνών, ιδιαίτερα αυτές οι εθνικότητες Ζητώ από τη βελγική κυβέρνηση να τους χορηγήσει θεώρηση. Τους ε, λέω, κοιτάξτε, έχω όλα τα δικαιολογητικά, αλλά παρόλα αυτά δεν χορηγείται θεώρηση. Υπάρχει λοιπόν αυτό το κενό. Πρέπει να το καλύψουμε. Υπάρχει από το letter of intent, ε, η επιστολή προθέσεων στα αγγλικά, που αναφέρει ποιε είναι οι εγγυήσει και στη συνέχεια ένα θέατρο, για παράδειγμα, δηλώνει ότι μας ενδιαφέρει ε, αυτό το άτομο. Τους ε, δίνουμε τις, ε, τη σύμβαση και μετά τους δίνουμε και την επιστολή προθέσεων. Και από τη συνέχεια, στη συνέχεια αναπτύσσουμε μια, ένα συμβόλαιο. Γραφίζουμε ένα συμβόλαιο το οποίο και χρησιμοποιείται στον ιδιωτικό τομέα. Τέλος. Κατά πόσον ε, η ασφάλεια υγείας, τα τραπεζικά αποκόμματα, η κοινωνική πρόνοια στην οποία θέλουν να υπολογίζουν. Τα άτομα αυτά είναι επαγγελματίε. Λαμβάνουν μισθό σε περιπτώσεις ε, της ε, εταιριών ε, χορευτών έχουν συμβάσεις Τους υποχρεώνουμε επίσης να έχουν τραπεζικό λογαριασμό για να μπαίνουν τα χρήματα αυτά στον τραπεζικό λογαριασμό. Άρα η εγγύηση τη σύμβαση είναι και βαρύνει την πλευρά τη εταιρεία και όχι τόσο του καλλιτέχνε. Κατά πόσον ε, έχουν τώρα κοινωνική πρόνοια στο Βελγίο, το πληρώνουν. Αλλά σε γενικέ γραμμέ δεν πληρώνουν του όρου για να μπορούν να έχουν ωφέλη συνταξιβατικά, επιδόματα ενεργεία αλλά δεν είναι το βασικό θέμα που του απασχολεί. Αυτές ήταν οι βασικές ερωτήσεις, αν δεν κάνω λάθο, που ετέθησαν. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ, λέει πρόεδρο. Ο κύριο Ντεγιάγκερ έχει το λόγο. Ευχαριστώ. Πράγματι, τα άτομα που προσλαμβάνονται από τον οργανισμό της κυρίας παρουσιάζουν όλα τα χέγγια αλλά δεν είναι μόνο εκείνοι που θα παρουσιάζει οι καλλιτέχνε. Δεν είναι μόνο εκείνοι που θα ζητήσουν αυτή τη θεώρηση. Θα πρέπει, να σκεφτούμε το πόσοι μπορεί να είναι οι ετούντε τελικά. Αν υπάρχουν άνθρωποι καλή την πίστη ζητούν τη θεώρηση, δεν θα υπάρξουν προβλήματα. Το πρόβλημα είναι αυτοί ακριβώ που θα μας ε, υποβάλουν έγγραφα σχετικά αμφίβολα, λένε είναι αρκετά περίπλοκο να ξέρουμε αν είναι ακριβή αληθή ή όχι. Χρειάζεται συνεπώς έρευνα και αυτό είναι χρονοβόρο. Ε, αυτό παίρνει χρόνο, όχι οι καλλιτυπίστοι ε, άνθρωποι, όχι εσείς, όχι οι καλλιτέχνες σας, αλλά εκείνοι για τους οποίους δεν είμαστε σίγουροι. Θα είναι ένας, μια μικρός θεία όταν ήμουν γενικός πρόξενος στην ακτή ελεφαντοστού, ε, είχα πολλές έτσι, πολλούς μικρούς θειάσους που ερχόταν με συμβάσεις, με επιτροπές της γειτονιάς, με διάφορες οργανώσεις στη Γαλλία, που να ξέρω εγώ. Αυτή η θίαση ήταν σοβαρή, δεν ήταν, διότι μπορούσαν να αγοράσουν έγγραφα επίσημα, νόμιμα, που θα έλεγαν ότι αυτός ο θείασος είχε καταχωρηθεί και ανήκε δεν ξέρω σε ποιο φορέα καλλιτεχνών δεν υπάρχουν εγγυήσει για κάποιους οργανισμούς στην ε, Γαλλία. Πρέπει να προσέχουμε. Δεν είναι ο δικαιούχος το πρόβλημα. Το πρόβλημα είναι η ποσότητα των ενδεχομένων ετούντων. Αυτό είναι το πραγματικό πρόβλημα και υπάρχει φόρτος που θα μπορούσε να είναι πολύ μεγάλος για τα προξενία. Ανοίγουμε τεράστιο πεδίο. Τι ούτω τρόπος. Ο κύριος Χτεφέ μου έθεσε ένα ερώτημα. Δηλαδή, πώς να βελτιώσουμε την κατάσταση. Διαφυλάσσοντας το οικονομικό όφελος. Ειλικρινά δεν το πολύ σκεφτικά. Αυτό είναι ένα σχέδιο που ανακαλύπτω τώρα που καταφθάνει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Πώς τα βλέπω εγώ τα πράγματα το να έχουμε έναν κανονισμό ειδικό για μια τόσο ιδιαίτερη περίπτωση αυτό μόνο αυξάνει τα κείμενα που θα πρέπει να εφαρμόσουν τα προξενία. Το καλύτερο θα ήταν να κωδικοποιήσουμε τα πράγματα και έχουμε ένα ενιαίο κείμενο. Να καλύπτει τα πάντα. Ε, ε, ε, και να μην είναι δυσανάγνωστο όταν το διαβάζει κανείς. Καλύτερο θα ήταν αυτή η περίπτωση να συμπεριληφθεί στα ήδη ισχύοντα και υφιστάμενα. Έχουμε τη δυνατότητα της παράτασης. Από εκεί ας ξεκινήσουμε. Εκεί υπάρχουν διέξοδοι. Στο άρθρο 33 που προανέφερα. Διότι αν παρατηνούμε, εν τη αυτή περιπτώση, η διοικητική αρχή που ασχολείται με την παράταση θα έχει ένα ιστορικό των τριών περασμένων μηνών και θα μπορεί να κρίνει και να αποφασίσει όσον αφορά την αξιοπιστία του οργανισμού που προσκαλεί αυτούς τους ανθρώπους και μπορεί να κρίνει τα χέγγια που δίνει ο οργανισμός αυτός. Το να δημιουργήσουμε εξ αρχής μία θεώρηση περιοδίας τουριστική για αόριστο αριθμό κατηγοριών Νομίζω ότι αυτό θα δημιουργούσε μεγάλο φόρτο εργασίας για τα προξενία και θα υπήρχε και κίνδυνος εν πάση περιπτώσει σώρευσης εργασιών για τα προξενία. Και τα προξενία έχοντας προσωπικό που δεν είναι και πολύ άριθμο και ξέρω τι γίνεται να μειώνεται το προσωπικό. Πώς θα τα βγάλουν πέρα. Αν ασχολούμαι με τούντες ε, τη θεώρηση αυτή ε, δεν θα μπορώ να ασχοληθώ πλέον με τους άλλους είναι όπω αυτοί που θέλουν άμεσα ένα ραντεβού. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να βγάλω κάποιον άλλον, Όπω με τον γιατρό. Θα πρέπει κάποιον άλλον να βγάλει τη μέση ο γιατρό για να δεχτεί αυτόν που έχει επίγουσα ανάγκη. Ε, όσο δίνουμε στου μεν δεν δίνουμε στου δε. Ε, πρέπει να είμαστε προσεκτικοί. Έχουμε έναν κώδικα θεωρήσεων, θα πρέπει να είμαστε εφάνταστοι αν θέλουμε να γίνουν ιδέωσε προσαρμογέ για να υπησέλθει εντό αυτού του πλαισίου η κατηγορία αυτή και αξιόπιστοι άνθρωποι που πραγματικά χρειάζονται αυτού του είδους θεωρήσεις. Το αναγνωρίζω. Υπάρχει ένα νομικό κενό. Okay, now we have a time for European. Να ακούσουμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Την κυρία Γιόλαντα. Να πάρει το λόγο. Σα ευχαριστώ, ευχαριστώ και όλους τους μελητέ. Έχω... Ακούσαμε πολλά ερωτήσει. Να ξεκινήσω με το κατά πόσο υπάρχει ανάγκη για αυτή την ανάγκη, για τη θεωρία περιοδιά. Ναι, θεώρηση περιοδίας. Ναι, υπάρχει ένα μικρό κενό και πρακτικές δυσκολίες. Μπορεί να υπάρχει λοιπόν θεμητό συμφέρον και ε, ανάγκη να ταξιδέψουν οι υπήκοοι αυτοί χωρών, άλλων χωρών παραπάνω από 50 μέρες. Υπάρχει και οικονομική απώλεια. Θα πρέπει λοιπόν να βρούμε ένα μέσο να αντιμετωπίσουμε το ζήτημα αυτό. Το κάνουν αυτό κάποια κράτη-μέλη, αλλά με περιορισμένο τρόπο και αυτό δεν συνάδει με τους κανόνες του Σέγγεν για τις διμερείς συμφωνίες που συνήφθησαν την προηγούμενη αιώνα και στη θεωρία μπορεί να δίνει τη δυνατότητα για έναν πολίτη της Νέας Ζηλανδίας να μένει μια παραπάνω από τέσσερα χρόνια στην περιοχή Σέγγεν. Συνάντη αυτό με την πολιτική πρακτικές δυσκολίες τώρα για τους ελέγχους στα σύνορα όταν φεύγουν τα άτομα αυτά αν δεν γνωρίζουν τις διμερείς συμφωνίες το οποίο και ισχύει συχνά θα τους θεωρούνται ως ε, άτομα που έχουν παραμείνει παραπάνω από τη διάρκεια τη θεωρήση του. Είναι καλή, θεωρούμε λοιπόν η πρόταση για να αντιμετωπίσουμε τα ζητήματα αυτά και να βρούμε μια λύση. Είμαστε ανοιχτοί προ συζήτηση, εξέβρεση μέσων συμβιβασμού και αντιλαμβανόμαστε τι ανάγκε. Δεν είμαστε κατά τη συγχώνευση με τον κώδικα των θεωρήσεων κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων. Βλέπουμε ότι υπάρχουν πολλέ ε, τέτοιε αναφορέ, γιατί πολλέ από τι διατάξει του κώδικα των θεωρήσεων ισχύουν εδώ. Δεν θα υπάρξουν τόσε πολλέ διτάξει που θα είναι διαφορετικέ. Το ίδιο άτομο που ε, επεξεργάζεται τι θεωρήσει αυτέ θα με κάποια επιπρόσθετη κατάρτιση να επεξεργάζεται και τι άλλε θεωρήσει. Θα μπορούσαμε να δώσουμε και μια προθεσμία για την εκπαίδευση αυτή, αλλά πραγματικά δεν θα σημαίνει αυτό τεράστιο φόρτο για τα προξενία γιατί είναι χαμηλές, ε, χαμηλός ο ρυθμός των αιτήσεων και πολλές από τις διδάξεις ήταν ίδιες. Ισχύουν για όλους. Όλοι θα παίρνουν ε, τέτοιες θεωρήσεις ε, περιοδίας, όχι μόνο όσοι πληρούν τους όρους αυτούς που ορίζει ο κανονισμός. Έχουμε λοιπόν αυτό το θέμα Για να έχουν μέσα διαβίωση μέχρι από ένα έτος θα πρέπει λοιπόν να αποδεχτεί ότι υπάρχουν αυτά τα μέσα διαβίωσης. Η απόδειξη για παραμονή 90 ημερών. Επίσης απόδειξη ότι σκοπεύουν να επιστρέψουν στη χώρα τους και αυτό λοιπόν το εκτιμά το προξενείο κατά πόσον υπάρχει πρόθεση. Αυτό πάντα εκτιμάται και είναι σημαντικό μέσο. Αν αυτές, αυτοί οι όροι πληρούνται και είναι πιο αυστηροί από ότι στα άλλα μέσα θεωρήσεων. Τότε λοιπόν, αν δεν πληρούνται οι όροι αυτοί, πολύ απλά δεν χορηγείται η θεώρηση. Είναι πιο αυστηρές λοιπόν αυτές, ε, αυτοί οι όροι. Γιατί δεν υπάρχει περιορισμός τώρα σε κάποια συγκεκριμένη ομάδα ατόμων. Στην αρχή, όταν υποβάλαμε την πρόταση, και πάντα αυτό το παράδειγμα χρησιμοποιούμε. Λαμβάναμε πάρα πολλές ενστάσεις και παράπονα από τους καλλιτέχνες. Είναι πιθανό λοιπόν αυτοί να υποφεληθούν, αλλά γιατί αν υπάρχει κάποιο μονόμενος ταξιδιώτης που θέλει να ταξιδέψει για παραπάνω από 90 ημέρε στην περιοχή Σέγγεν και δεν αποτελεί ιδιαίτερο κίνδυνο, Αμερικανοί, Ιάπωνες έχουν χρήματα, γιατί να με, μη βρεθεί ένα μέσο να βοηθηθούν και αυτοί. Που και αυτοί μπορεί να έχουν το συμφέρον και ανάγκη να ταξιδέψουν. Γι' αυτό λοιπόν δεν θεωρήσαμε ότι είχε, ότι ήταν σκόπιμο να περιορίσουμε το πεδίο εφαρμογή του κανονισμού, αρκεί να πληρούνται, επαναλαμβάνω, οι όροι που αναφέρονται, που είναι επιπρόσθετοι σε σχέση με αυτούς της κανονικής ε, θεώρησης. Το πόσο επιβαρύνονται τα προξενία σε ό,τι αφορά το άρθρο 33. Δεν πιστεύουμε ότι το άρθρο 33 ε, του κώδικα θεωρήσεων αποτελεί μέσο που εγγυάται τέτοια ζητήματα δεν πιστεύουμε ότι αν στην ε, κατηγορία αυτή ετούντο. Τώρα, για τα θέματα που έθεσε ο κύριος Ντεπρέ, για το τι γίνεται μετά από δύο χρόνια, θα πρέπει να φύγουν από, το, από την ζώνη του Σέγγεν και να κάνουν αίτηση εκτός του χώρου Σέγγεν. Πρώτα λοιπόν θα πρέπει να καταλήψουν τον χώρο του Σέγγεν και μετά να κάνουν καινούργια ε, αίτηση. Αυτό ε, θα θέλαμε να δούμε πώς θα δημορφωθεί, γιατί αναφέρεται στον κώδικα των θεωρήσεων αλλά αν υπάρξει συγχώνευση νομίζω ότι θα είναι λίγο πιο σαφή τα πράγματα. Αυτά λίγο πολύ. Σας ευχαριστώ. Half a minute. λεπτό, 30 δευτερόλεπτα. κύριος Ντυπρέ, μία ερωτησούλα. Αν κατάλαβα καλά, τα, οι διατάξεις ε, του κώδικα παραμένουν εφαρμοστές και το ίδιο και η προθεσμία. Δηλαδή η προθεσμία εννοώ για την υποβολή της αίτησης. Καλά κατάλαβα. Αυτό τι σημαίνει. Αυτός που έμεινε ένα χρόνο και έγινε η παράταση, φεύγει για 15 μέρες και μετά υποβάλλει ένα αίτημα μπορεί να ξαρχίσει από την αρχή. Ε, δηλαδή είναι ένα σύστημα μόνιμης διαμονής. Προσπαθώ να καταλάβω το μηχανισμό. Δεν είναι κριτική. Προσπαθώ να καταλάβω. Well, it's, he should leave, if I may reply, he should leave and then he should... Ε, ναι, θα πρέπει να φύγει και μετά να, αποφασίσει, να αποδείξει συγγνώμη αν πληρεί τις ε, προϋποθέσεις. Αλλά ο στόχος δεν είναι η μόνιμη διαμονή, αλλά κατανοούντα το όριο 90 ημέρες κτλ. Πρέπει να πληρούνται όλες οι απαιτήσεις. Okay, everything is clear. Uh, now... Τώρα είναι ξεκάθαρα τα πράγματα. Η κυρία Μόιρα Ροζ, που εκπροσωπεί το Συμβούλιο για τη Λιτανική Προεδρία, θα πάρει τώρα το λόγο. Mm. Ευχαριστώ. Αγαπητοί βουλευτές, Κοιτάξτε. Ε, λοιπόν, όσον αφορά το θέμα που συζητούμε, θέλω να αναφερθώ στην πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για αυτή την θεώρηση για ε, περιοδία. Ο στόχος της προτάσεως είναι να προσφέρουμε ένα καινοτόμο μέσο, μια νέα λύση σχετικά με το πώς μπορούμε να καλύψουμε το κενό που υπάρχει μεταξύ των θεωρήσεων βραχίας διαρκείας για τον χώρο Σέγγεν και από την άλλη πλευρά έχουμε τους κανόνες Ευρωπαϊκής Ενώσης και των Κατών μελών για τις θεωρήσεις ε, μακράς διαρκείας, μακράς ε, διαμονής. Τον Απρίλιο του 2014 κατέθεσε την πρόταση η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ταυτόχρονα έγινε μια πρόταση για αναθεώρηση του κώδικα ε, για τις ε, θεωρήσεις. Θα ήθελα να σας ενημερώσω πως οι αρχικές ε, συζητήσεις που έγιναν για την εν λόγω πρόταση έμειναν με αυτές που είχαμε Ήδη τον Απρίλιο του 2014 ε, με την Ελληνική Προεδρία. Εμείς εστιάσαμε την προσοχή μας σε αυτές τις προτάσεις, συνεχίσαμε ε, τη δουλειά των δύο προηγούμενων προεδριών και κατά τη διάρκεια της Λετωνικής Προεδρίας Ε, Εξεργαστήκαμε τρεις φορές αυτή την πρόταση για τις θεωρήσεις. Έγινε κατάρθρο εξέταση της πρότασης ε, και στην τελευταία συνεδρία του Συμβουλίου που έγινε πριν από δύο ημέρες ολοκληρώθηκε αυτή η κατάστρο εξέταση της πρότασης. Η πρόταση αυτή της ε, θεώρησης ε, περιοδίας ε, συνδέεται άρρηκτα με την αναθεώρηση του κώδικα θεωρήσεων διότι πολλές διατάξεις αντιγράφηκαν και επαναλαμβάνονται και φυσικά το έλαβε αυτό υπόψη το Συμβούλιο στις εργασίες του. Εν κατακλείδη θα ήθελα να τονίσω πως ε, ο στόχος της Λατινικής ε, Προεδρίας ήταν να προωθήσει στο μέτρο του δυνατού την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ε, επιτυχώς ολοκληρώσαμε την πρώτη κατάστροφη εξέταση της πρότασης ε, όπως και με την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το νέο κώδικα θεωρήσεων, θα συνεχιστεί η εργασία ε, και θα παραδώσουμε τη σκητάλη στην επόμενη προεδρία, την Μουριανή. Σας ευχαριστώ για την προσοχή που δείξατε. Σας ευχαριστούμε και τέλος για να κλείσει αυτή, αυτό το τμήμα της συζήτησης θα δώσω το λόγο στον κύριο Μπρίς Οχτεφ για τα συμπεράσματα. Παρακαλώ, κύριε Οχτεφέ. Ευχαριστώ, κύριε Αντιπρόεδρε. Νομίζω ότι ακούσαμε παρεμβάσεις υπέρ της ε, θεώρησης ε, περιοδίας αυτής. Επίσης, ακούσαμε κάποιον που βασιζόμενος στην ευρύτατη εμπειρία που είχε, ε, προσπάθησε να θέσει και κάποια όρια εγώ προσωπικά καταλαβαίνω στις ευρωπαϊκές περιοχές ποιες δυσκολίες θα αντιμετωπίζουν οι καλλιτέχνες. Ταυτόχρονα όμως προσθέτω πως υπάρχει και η διάσταση της ασφάλειας και οι ανησυχίες που έχω δεν έρονται από αυτά που άκουσα. Ζητώ συγγνώμη, θα κάνω μια μεταφορά, ε, μεταπαρομοίωση. Ε, ανοίγουμε μια πόρτα χωρίς να ξέρουμε τι κρύβεται πίσω από την πόρτα. Δεν άκουσα απάντηση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το πώς θα μπορούσαμε να έχουμε ένα ε, υδατοστεγές ε, σύστημα. Μπορούμε λοιπόν να μιλάμε και να λειτουργούμε βάσει ενός ατελού συστήματος ε, ενώ ως προς τις τρομοκρατικές απειλές είμαστε στο ανώτερο το επίπεδο παγρύπνησης. δηλαδή θα εκθέσουμε τους πολίτες σε πρόσθετους κινδύνους. Ε, αυτοί λοιπόν που ε, ε, αυτοχαρακτηρίζονται ως τουρίστες μπορούν και να διαιτήσουν οι ορισμένες προϋποθέσεις την θεώρηση περιοδίας και από ό,τι ακούσαμε μπορεί να υπάρξει παράκαμψη της διαδικασίας. Ε, δεν πρόκειται για 60 με 120 όπως μας λέει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Εκατομμύρια επί εκατομμυρίων μπορεί να είναι αυτοί οι άνθρωποι. Θα ήθελα να σας πω κάποια πράγματα για την ε, αποστολή που κάναμε τον Απρίλη στην Κωνσταντινούπολη που είναι ε, διαφωτιστική για την έκδοση των θεωρήσεων. Δεν είναι θεωρία, είναι ε, πράξη. Επί το που παρατηρήσαμε, ήσασταν και εκεί κάποιοι, επισκεπτόμενοι τα προξενία της Γαλλίας, Γερμανίας και της Ισπανίας και βλέποντας την το που εφαρμογή του κεκτημένου Σέγγιν, α, και σε συνεργασία με τον εξωτερικό πάροχο, τον VFS ε, ε, Global, που ακούσαμε στο πρώτο τμήμα της συζήτηση, Κάναμε πολύ επικοδοματικές παρατηρήσεις και ακούσαμε επιτόπου πράγματα που ε, έχουν μεγάλο νόημα και πρέπει να, στα οποία πρέπει να αποδώσουμε μεγάλη σημασία. Καταρχάς υπάρχουν πολλοί αυτοί είναι ασχετικός αριθμό αυτών που δεν τηρούν το κανόνα των 90 ημερών. Και για τα ε, πρόξενη είναι πολύ δύσκολο να ε, επιτευχθεί αποτελεσματικό έλεγχο. Λοιπόν, ποιο είναι ο ρόλος μας εμάς να φτιάξουμε ένα νέο είδος θεώρησης ε, που θα οξύνει περαιτέρω αυτό το φαινόμενο παράκαμψη των κανόνων δεύτερον. ο αριθμός των πλαστοποιημένων, παραποιημένων, πλαστών ή παραποιημένων εγγράφων είναι ανησυχητικά ε, υψηλό, το ακούσαμε και από πρώην πρόξενο, στην ε, τουρκική αγορά όπως μας είπαν, τα πλαστά διαβατήρια κάνουν από 2 έως 10.000 τιμή αγοράς. Για φανταστείτε λοιπόν σε ε, ανοργάνωτες χώρες ή σε εμπόλεμες ζώνες ή όπου δεν υπάρχει διοικητική δομή, δηλαδή είναι αστείο να βρει κάποιος πλαστό διαβατήριο. Πανεύκολο. Λοιπόν, ε, φανταστείτε ότι έχουμε προξενία με περιορισμένους πόρους που πρέπει να εξετάζουν την ε, γνησιότητα αυτών των εγγράφων. Υπό το φως λοιπόν αυτών που ακούσαμε και πραγματικά άκουσα μεγάλο ενδιαφέρον όλες τις απόψεις, δεν έχουμε τέτοια δυνατότητα να έχουμε μια θεώρηση που στο πεδίο εφαρμογή τους ε, ε, ουσιαστικά εντάσσονται όλοι αδιακρίτως. Η παρά είναι αφηρημένη η έννοια του τουρίστα. Ε, μπορεί να ερμηνευτεί η έννοια με τρόπο που δεν μας επιτρέπει με τα μέσα που έχουμε στη διάθεσή μας να αντιμετωπίζει, να αντιμετωπίσουμε την κατάσταση. Ε, έχουμε την, ε, τις θεωρήσεις σύντομης διαμονής, τις άδειες διαμονής των κρατών μελών, τις ετομιακές οδηγίες για τους φοιτητές και τις, ε, τους ερευνητές, πολλές διαφορετικές κατηγορίες. Όλοι αυτοί μπορούν να ζητήσουν λοιπόν αυτή την λεγόμενη θεώρηση περιοδία τι σημαίνει αυτό. Ε, από διοικητική πλευράς εάν παραταθούν, ε, συγγνώμη, εκταθούν τα κοινωνικά δικαιώματα σε ε, πρόσθετους δικαιούχους. Τα έλεγα και προηγουμένω. Αυτό είναι, είναι συνάρτηση τη πολιτικής που ακολουθεί κάθε κράτος μέλος. Όμως προ το παρόν δεν έχουμε ε, πιστικά στοιχεία. Παρακαλώ να με πίστα αν έχετε επιπρόσθετα στοιχεία. Εγώ ζητώ αξιολόγηση αντικτύπου για αυτήν την, ε, αυτό το είδο της και τα αναμενόμενα κοινωνικά ωφέλη αλλά και τον αντίκτυπο για το, τις πληθυσμιακές ομάδες που απαλλάσσονται από υποχρέωση θεώρηση. Θέλουμε την ανάλυση να συλληφθεί υπόψη το κόστος ε, για το προσωπικό, για τις θέσεις στα προξενία στις χώρες που μέχρι τούδε δεν εκδίδουν ε, θεωρήσεις. Επίσης ε, πρέπει να εντοπιστούν οι κίνδυνοι που ολοχεύουν για την ασφάλεια και την παράνομη μετανάστευση και σας ευχαριστώ όλους για την υποστήριξη που μου προσφέρετε στο διάβημά μου αυτό. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ, ευχαριστώ. Ευχαριστώ όλους που πήραν το λόγο, τους φιλοξενούμενους, τα μέλη μας. Ευχαριστώ για τη συνεισφορά σας, την καρποφόρα και ενδιαφέρουσα συζήτηση. Η Επιτροπή ΛΥΜΠΕ θα συνεχίσει τις εργασίες της επί του θέματος. Είμαι βέβαιη ότι θα προχωρήσουμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ και τους διερμηνείς. Ευχαριστούμε. Καλό σας βράδυ.